Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των ευρωβουλευτών απουσιάζει, ελπίζω μέσα στο επόμενο ημίωρο να μπορέσουν να έρθουν περισσότεροι συνάδελφοι εδώ στην αίθουσα αυτοί που είμαστε παρόντες ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα να ακούσουμε τους τέσσερις προσκεκλημένους μας για να μας ε, μιλήσουν για αυτή την τόσο σημαντική ακρόαση της ε, διαχείρισης των αλληλευτικών αποθεμάτων και τη διαχείριση του αλληλευτικού στόλου. Έχουμε τέσσερις προσκεκλημένους και ε, επειδή απουσιάζουν και προσκεκλημένοι, όχι μόνο ευρωβουλευτές, θα ήθελα να κάνω την εξής πρόταση. Για κάθε ένα από τα δύο τμήματα έχουμε περίπου μία ώρα και τρία τέταρτα, την οποία φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό να εξαντλήσουμε. Και επομένως ο καθένας από τους αγορητές θα μπορεί να λάβει το λόγο ε, το πολύ για μισή ώρα, ούτε και αυτό είναι υποχρεωτικό. Κατόπιν θα έχουμε ένα ημίωρο για συζήτηση. Ε, και για το δεύτερο τμήμα θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή έχουμε δύο μιλητές και επαναλαμβάνω, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβετε το λόγο για μισή ώρα. Αλλά εάν θέλετε να μιλήσετε λίγο περισσότερο από ό,τι είχαμε προβλέψει αρχικώς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερο χρόνο. Να καλωσορίσω λοιπόν όλους σας και πριν περάσουμε στο πρώτο τμήμα της ακρόασης για τη διαχείριση των αλληλευτικών αποθεμάτων, να σας πω ότι έχουμε δύο προσκεκλημένους εγνωσμένου κύρους. Ε, πρώτος είναι ο κύριος Ενρίκε Λόπες Βέγγα. Εδώ λέει ότι είναι ε, θαλάσσιος βιολόγος, αλλά πέραν αυτού είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ε, είχε θέσεις και σε κυβερνητικό επίπεδο και στον κλάδο και είναι ένας από τους ε, μεγάλους γνώστες της αλίας, ιδίως της ισπανικής αλίας και πιο συγκεκριμένα της αλίας στη Γαλλικία θα πρέπει να σας πω ότι πρόκειται για έναν ε, ε, επιστήμονα ο οποίος μπορεί να μας παρουσιάσει πολλά στοιχεία για τις πτυχές που θα συζητήσουμε σήμερα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον Ντόν Ενερίκε και τον καλό να έρθει εδώ γιατί νομίζω ότι έχει και μια παρουσίαση PowerPoint. Pues nada, tiene usted la palabra. Cuando quiera puede empezar. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε. Θα κάνω μία απόπειρα να προσπαθήσω να απαντήσω εν συντομία. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστώ μισή ώρα στη διάθεσή μου, διότι μας είχαν πει ότι θα μιλήσουμε για πολύ λιγότερο. Θα κάνω τουλάχιστον μία απόπειρα να δώσω μία εικόνα από προσωπικής ε, σκοπιάς, αλλά βασισμένη στην ε, επαγγελματική μου εμπειρία η οποία είναι ε, μεγάλη γιατί είμαστε κυλοκυωμένοι μεταξύ άλλων. Καταρχάς λοιπόν, σε αυτό το πρώτο τμήμα της παρουσίασή μας υπάρχει το ερώτημα ποιοι θα πρέπει να είναι οι στόχοι της ε, διαχείρισης της αλίας. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά και έχει σχέση με το σεβασμό με κάθε λεπτομέρεια στην νομοθεσία που έχουμε στις συνθήκες. Πρέπει να ομολογήσω ότι εμένα προσωπικά μου είναι λίγο αποθητικό το να διαπιστώνω στη νέα νομοθεσία ότι γίνεται μια νέα απόπειρα να ορίσουμε εκ νέου τους στόχους της ελευτικής πολιτικής. Οι στόχοι της ελευτικής πολιτικής, κατά την άποψή μου, είναι σαφέστατοι. Δεν είναι κακοί, είναι πολύ συγκεκριμένη, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι που διαφωνούν, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι πολύ συγκεκριμένη και διατυπώνονται στο άρθρο 39 της συνθήκης, στο οποίο όχι μόνο απαριθμούνται με απόλυτη ακρίβεια, αλλά καθορίζεται και πώς πρέπει να εφαρμόζονται, ιδίως η αρχή της ασότητας και της πρόληψης. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να κάνω είναι Δεδομένου ότι θεωρώ ότι πρόκειται για καλούς στόχους για την αλληλευτική πολιτική, Αφενός έχουμε ε, δυνατότητες να κάνουμε προτάσεις ε, στη μεταρρύθμιση για να βελτιωθούν καλύτερα οι στόχοι, αλλά θα ήταν νομικό πρόσχημα πρώτης τάξεως να προσπαθήσουμε να βρούμε τι ακριβώς ε, πρέπει να κάνουμε για την εφαρμογή των στόχων που έχουμε στη συνθήκη. Και νομίζω, και σε αυτό θα επικεντρώσω και την παρουσίασή μου, ότι η συνθήκη είναι πολύ συγκεκριμένη και τονίζει κυρίως τον άνθρωπο, τον άνδρα και τη γυναίκα, τους ανθρώπους. Και λέει ότι πρέπει να αυξηθεί η γεωργική παραγωγή, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι παραγωγικοί παράγοντες και κυρίως η εργασία, που είναι το κοινωνικό σκέλος. Είναι σαφές λοιπόν ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ένα βιωτικό επίπεδο το οποίο θα είναι το πλέον κατάλληλο και αυτό φυσικά δεν μπορεί να το καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα πρέπει να γίνει ε, βάσει των ανθρώπων που επηρεάζονται, τους οποίους πολλές φορές αγνοούμε. Και από την άλλη υπάρχουν και τα υπόλοιπα σκέλη τα οποία ε, είναι η διασφάλιση της αγοράς, να υπάρχει σωστή διαχείριση και να υπάρχουν και λογικές τιμές. Αν συγκρίνουμε λοιπόν αυτό που έχουμε στη συνθήκη με αυτό που προτείνεται στη νέα νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω ότι ουσιαστικά κατακρεωργούμε τη συνθήκη χωρίς καμία ε, διαφορετική ερμηνεία. Μου φαίνεται ότι έχει γίνει ελάχιστη προσαρμογή ε, στα όσα γίνονται στην πλειονότητα των χωρών μας. Αυτό που λέω πάντα όταν συζητάμε το θέμα αυτό ε, τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι ότι είναι σαν να προσπαθούμε να μεταρρυθμίσουμε το Σύνταγμα μέσω Προεδρικού ή Υπουργικού Διατάγματος. Αυτό είναι αδιανόητο και νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τη μεταρρύθμιση κοινή ελευθερικής πολιτικής. Ο μόνος τρόπος να γίνει μια μεταρρύθμιση στους στόχους της κοινή ελευθερικής πολιτικής είναι αυτό που λέει εδώ, να υπάρχει μια παραπομπή στη συνθήκη. Αυτό άλλωστε καλείται ε, καλή νομική τεχνική. Δεν χρειάζεται να σας την ορίσω εγώ, την έχουν ορίσει ήδη άλλοι πριν από μένα. Δεν είναι αρκετά συγκεκριμένη οι στόχοι και θα πρέπει, ε, εδώ έρχεται και το επόμενο στοιχείο, να καθορίσουμε πώς θα επιτύχουμε να έχουμε τις τεχνικές που μας χρειάζονται για να καθορίσουμε τους στόχους, που είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με την απόπειρα να τους ξαναορίσουμε δεν ε, πρόκειται για περίεργα πράγματα και δεν ε, <coughs> προκύπτουν περίεργα πράγματα από την προηγούμενη νομοθεσία. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω στο γεγονός και μου είπαν ότι κάποιοι θα μου τραβήξουν το αυτοί για, τη, ε, για αυτό που θα σας πω στη συνέχεια. Τα συστήματα είναι προσαρμοσμένα στον άνθρωπο και όχι οι άνθρωποι στα συστήματα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να προέχει είναι η ευημερία των πολιτών που σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να υπάρχει και λογική εκμετάλλευση του περιβάλλοντος και να κρατεί και η κοινή λογική η οποία είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη σε οποιαδήποτε νομοθεσία. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περαιτέρω στους στόχους, καταρχάς διότι με αποθεί το να προσπαθούμε να καθορίσουμε άλλους στόχους πέραν αυτών της συνθήκης που είναι πλέον κατάλληλοι, είναι απόλυτα συγκεκριμένοι και που θεωρώ ότι είναι απόλυτα δυνατό μέσω νομοθεσίας να πούμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτού. Δεν χρειάζεται όμως να ορίσουμε εκ νέου στόχους που είναι σαφώς καθορισμένοι. Το επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον η μέγιστη βιώσιμη απόδοση είναι ο κατάλληλος στόχος. Και λέγεται, εγώ είμαι από τη Γαλλικία, μου λένε ότι στη Γαλλικία δεν είμαστε και ιδιαίτερα συγκεκριμένοι. Η φήμη μας είναι ότι είναι αμφίσιμη και σε αυτή την περίπτωση θα σας απαντήσω ίσως. Είναι κατάλληλος ο στόχος. Ίσως. Θα μπορούσε να είναι, θα μπορούσε και να μην είναι. Εξαρτάται από το πώς σκοπεύουμε να τον υλοποιήσουμε. Καταρχάς, από πού προέρχεται ε, το όλο θέμα της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Είναι αλήθεια ότι στο διεθνέ δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας λέγεται ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ρυθμίζουν την αλληλεία κατά τρόπον ώστε τα αποθέματα να έχουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Και είναι αλήθεια ότι στη διάσκεψη του Johannesburg, στη δήλωση που προέκυψε από εκεί, αναφερόμαστε στο ε, σχέδιο εφαρμογή και εκεί, στην παράγραφο 36, γίνεται μία στο γεγονός ότι θα πρέπει να ρυθμίζονται τα υποθέματα σε επίπεδα που να οδηγούν στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, αλλά εδώ σας ευχηθώ την προσοχή και ή δυνατόν το αργότερο το 2015. Ένα στοιχείο αυτό το κρατάμε. Ίσως βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οπισθοδρόμησε λίγο και να μην ε, επιμένει κατηγορηματικά στο 2015 διότι υπάρχουν και αποθέματα στα οποία θα ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί, ακόμα και αν ε, κλείναμε την αλληλεία για συγκεκριμένα είδη, δεν θα μπορούσαμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Ε, αυτό μας οδηγεί στο να σκεφτούμε στο κατά πόσον είναι λογικά τα όσα κάνουμε, που ε, ερχόμαστε και στην περίπτωση του γάδου, που είναι πολύ ε, δύσκολο να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι, θα είναι αδύνατο να έχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση το 2015, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε και στους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά και υπερβολικές ποινές, διότι στο κάτω-κάτω της γραφής αυτοί οι άνθρωποι που αλλιεύουν αυτά τα αποθέματα ε, τα οποία είναι σε κίνδυνο, είναι αυτοί οι οποίοι θα πληχθούν εάν εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι λογικό. Θα ήθελα όμως να πω το εξής είδα σε κάποια κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λέει ότι είμαστε υποχρεωμένοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη να επιτύχει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση το 2015, διότι μας υποχρεώνει αυτό το σχέδιο εφαρμογής. Εγώ διαφωνώ απολύτως. Δεν είναι αλήθεια ότι είμαστε υποχρεωμένοι νομικώς να υλοποιήσουμε το σχέδιο θα μπορούσαμε να δεσμευόμαστε ηθικώς, κάτι το οποίο είναι ε, διαφορετικό, διότι έχουμε μια δήλωση, αλλά δεν είναι συνθήκη η δήλωση αυτή και δεν ε, ε, προϋποθέτει οι υποχρεώσεις αυτής του μεγέθους στα κράτη-μέλη που έχουν προσυπογράψει αυτή την υποχρέωση. Και σας το λέω, όχι γιατί δεν θεωρώ ότι η μέγιστη βιώσιμη απόδοση είναι το επιθυμητό, αλλά γιατί δεν υπάρχει λόγος να δεσμευτούμε να επιτύχουμε το στόχο το 2015 όταν οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και οι ζημίες που μπορεί να προκληθούν για τους ανθρώπους που ε, πλήττονται από αυτά τα μέσα θα είναι ανυπόφορες. Θα ήθελα να υπενθυμίσω επίσης από πού αρχίζει, απορρέει η αρχή της μέγιστης βιώσιμης απο, αυτα τα μεσα θα ειναι ανυποφορες θα ηθελα να υπενθυμισω επισης απο που αρχιζει απορρεει η αρχη της μεγιστης βιωσιμης απο θα περάσουμε στο, στην Ιουρασική περίοδο που είχαμε τη διαχείριση των αποθεμάτων. Χρησιμοποιώ αυτό ως παράδειγμα διότι θα ήθελα να τονίσω κάποια στοιχεία. Η έννοια της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης προκύπτει από συγκεκριμένα μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται. Καταρχάς υπάρχουν δύο οικογένειες μοντέλων. Η μία οικογένεια είναι της γενικευμένης παραγωγής ε, που βασίζει τα μοντέλα της σε μία λογική που εφαρμόζεται τους ε, πληθυσμούς των ε, αλλιευμάτων αλλά και στους ανθρώπινους πληθυσμούς. Και εδώ έχουμε λοιπόν αυτή την ε, λογιστική καμπύλη την οποία ανέπτυξε πριν από αρκετούς αιώνες ένας Βέλγος και έλεγε το ίδιο ακριβώς πράγμα, ότι οι άνθρωποι δηλαδή συμπεριφέρονται και οι πληθυσμοί αυξάνονται όσο τους αντέχει το περιβάλλον. Και αυτή τη στιγμή δεν τους χωράει άλλο το περιβάλλον, σταματάει η ανάπτυξη. Και έρχεται λοιπόν η στιγμή στην οποία εφαρμοζόταν αυτό το μοντέλο και έχουμε και το κλασικό μοντέλο του Χέφερ, ε, του Σέιφερ, συγγνώμη, αλλά αυτό που θα ήθελα να τονίσω εγώ είναι ότι αυτά τα μοντέλα παραγωγής, της γενικευμένης παραγωγής, έχουν μια συγκεκριμένη στατιστική τεχνική. Δηλαδή, μπορεί να γίνει προσαρμογή στις μαθηματικές καμπύλες και μπορούμε να καθορίσουμε και περιθώρια ε, εμπιστοσύνης, σφάλματος. Αυτό που μας λέει λοιπόν το μοντέλο είναι ότι η μέγιστη βιώσιμη απόδοση του πληθυσμού αυτού αναμένεται να είναι 195 και μπορούμε να έχουμε και ένα ποσοστό ε, βεβαιότητας 95% και επομένως η πραγματική αξία θα είναι μεταξύ 370 ε, και 220 για τη μέγιστη δημοβιώσιμη απόδοση και εδώ έρχομαι και στο σημαντικό στοιχείο και για την αλλιευτική προσπάθεια, αντίστοιχα, μπορούμε να κάνουμε μια στατιστική εκτίμηση. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να περιμένουμε να είναι 37, αλλά από στατιστική σκοπιά μπορεί να είναι μεταξύ 34 και 40. Δεν γνωρίζουμε όμως επακριβώς ε, τι ποσοστά ε, έχουμε να επιτύχουμε το σωστό αριθμό. Κάνουμε λοιπόν εκτιμήσεις ε, μεταξύ δύο ανώτατων ε, ορίων, ανώτατο και κατώτατο όριο. Και γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί στη συνέχεια στα αναλυτικά μοντέλα αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού. Η λογική που τα διέπει, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να αντικατοπτρίζει το ίδιο, δεν το κάνει, διότι τα μοντέλα αυτά προκύπτουν από μια σειρά από τιμές, βιολογικές τιμές, ε, ε, οι οποίες ε, ένα τμήμα τους είναι γνωστό και ένα τμήμα τους είναι υποθετικές τιμές. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι η θνησιμότητα ανααλία για κάθε αλληλευτικό είδος είναι πάντα 0,2 και ποτέ δεν καταφέραμε να εξηγήσουμε για ποιο λόγο. Υποθέτουμε ότι είναι 0,2 και αυτό φυσικά έχει συνέπειε και για την εξέλιξη των μοντέλων αυτών, διότι υπάρχουν και άλλε παράμετροι εδώ πέρα που συνυπολογίζονται, όπω είναι για παράδειγμα η αύξηση. Εδώ έχουμε την ε, καμπύλη για την ε, μέγιστη βιώσιμη απόδειξη ε, για το γάδο του Ατλαντικού. Και βλέπετε ότι εδώ έχουμε ένα μέγιστο ποσοστό θνησιμότητα, το F maximum, και αυτό που μας δίνει το αναλυτικό μοντέλο είναι μία εκτίμηση. Δηλαδή, αντίθετα από αυτό που είχαμε προηγουμένω στο μοντέλο, όπου μα έλεγαν μια εκτιμηση δηλαδη αντίθετο απο αυτο που ειχαμε προηγουμενω τιμή και ένα περιφέρειο άνω και κάτω όριο, εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Χρησιμοποιούμε τεχνικές πολύ περίπλοκες, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσον μας δίνουν και το απαιτούμενο αποτέλεσμα. Πρόκειται για μία εκτίμηση και καθορίζουμε ένα F maximum που είναι το μέγιστο ε, ε, σημείο και αυτό, προσέξτε, δεν είναι εκνησιμότητα αναμέγιστη βιώσιμη απόδοση, είναι ένα άλλο σημείο το οποίο χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς. Δεν το απορρίπτω εδώ, αλλά θα πρέπει να το δούμε για αυτό που πραγματικά είναι. Από πού προκύπτει το πρόβλημα τώρα. Το πρόβλημα προκύπτει όταν μας ρωτάει κάποιος ποια είναι η μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Και εμείς κάνουμε μια ερμηνεία και λέμε ότι βγαίνει από μοντέλα γενικευμένης ε, ε, παραγωγής και εμείς το εφαρμόζουμε σε μοντέλα που χρησιμοποιούνται πολύ περίπλοκες και πολύ καλές αναλυτικές τεχνικές όμως. Υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ της ε, ονομαστικής ε, ε προσπάθειας που είναι το F μικρό και τη συνηθιμότητα που είναι το F το κεφαλαίο, που είναι ε, μια στιγμία τιμή, ενώ το F μικρό αντιπροσωπεύει ουσιαστικά τα σκάφη και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, το F το κεφαλαίο είναι ε, μια μαθηματική τιμή και ένα μαθηματικό ποσοστό και αυτή είναι διαφορά. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια θνησιμότητα αναείδος αλίας που να ανταποκρίνεται στο σημείο της αλληλευτικής προσπάθειας, το FMSY που έχουμε εδώ, το οποίο ανταποκρίνεται στην πραγματική μέγιστη βιώσιμη απόδειξη, απόδοση. Το πραγματική το τονίζω και εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα. Το πρόβλημα είναι ότι σε γενικές γραμμές αυτά τα αναλυτικά μοντέλα δεν ε, μας δίνεται το FMSY, αλλά χρησιμοποιούμε το F maximum, αυτό το μέγιστο, το οποίο είναι πολύ πιο περιοριστικό από το FMSY, εάν το είχαμε υπολογίσει από ένα μοντέλο γενικευμένης παραγωγής. Τι θέλω να σας πω με αυτόν τον τύπο. Όλες αυτές οι τιμές, και επαναλαμβάνω, δεν σας λέω ότι δεν χρησιμοποιούνται ή ότι είναι λανθασμένες. Είναι τα στοιχεία που έχουμε και πρέπει να τα χρησιμοποιούμε ως σημείο αναφοράς. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι δεν είναι συγκεκριμένες. Και δεν είναι ακριβείς. Δεν υπάρχει ακρίβεια. Και αυτό ε, είναι ε, ότι το σημαντικό χρησιμοποιούμε αξίες ε, και τιμές στις οποίες ξέρουμε ότι είμαστε γύρω-γύρω αλλά δεν ξέρουμε ακριβώ ποια είναι η ορθή τιμή. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να προσέξουμε εδώ είναι να μην αρχίσουν ε, οι δογματικές τάσεις, το οποίο έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν, που δημιουργεί πολλά προβλήματα και ειδικά αν θέσουμε ως ορίζοντα το 2015 είναι μεγάλο το πρόβλημα διότι χρησιμοποιούμε το F maximum και λέμε ότι πρέπει να έχουμε μείωση κατά 40% και θεωρούν ότι ε, με βάση αυτή την τιμή πρέπει να έχουμε μείωση 40%. Αυτό που προσπαθώ να σας πω εγώ είναι ότι παρά το γεγονός ότι φαίνεται πολύ λογικό και επιθυμητό να προσπαθούμε να επιτύχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, δεν είναι στην πραγματικότητα όταν ε, κάνουμε δύο πράγματα. Προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται με τα προβλήματα που υπάρχουν. Να σας θυμίσω την υπόθεση του Μερλούκιο όπου το F maximum ήταν 0,18 και τώρα είναι 0,29 ε, γιατί είχαμε κάνει λάθος στον υπολογισμό του ποσοστού ανάπτυξης. Επειδή όμως ε, εφαρμόζονται πολύ συγκεκριμένε περιοριστικές πολιτικές, ουσιαστικά προκαλούμε ζημία σε όσους συμμετέχουν στην αλία αυτού του είδους και δεν απαραίτητο να γίνει αυτό, θα το είχαμε αποφύγει αν είχαμε χρησιμοποιήσει μια βαθμιδόν προσέγγιση. Και δεν λέω ότι αυτό αποτελεί πρόσχημα για να μην κάνουμε τίποτα, απλώς πρέπει να έχουμε μια βαθμιαία εξέλιξη του μοντέλου. Τώρα, η μέγιστη βιώσιμη απόδοση πώς εφαρμόζεται. Μέχρι το ΔΕΗ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί φαίνεται ότι τελευταίως αλλάζουν λίγο τα πράγματα, ερμήνευε την αρχή αυτή λέγοντας ότι πρέπει να φτάσουμε στο F maximum για όλα τα αλλιευτικά είδη. Και εγώ σας λέω ότι αυτό είναι αδύνατο. Και είναι αδύνατο διότι αυτό που, απλουστεύουμε, που κάνουμε εδώ είναι ότι υπεραπλουστεύουμε. Έστω ότι έχουμε αλληλεία τριών ειδών. Το F1, το F2 και το F3. Και το καθένα έχει αλληλευτική προσπάθεια F και την οποία εφαρμόζουμε και στα τρία. Η αλλιευτική προσπάθεια F δημιουργεί διαφορετική θνησιμότητα ανά είδος για κάθε ένα από το είδος, ανάλογα με το εργαλείο που χρησιμοποιείται και με τον τρόπο με τον οποίο ε, αλλιεύουμε. Τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί αυτό που έχουμε στο ε, διάγραμμα, δεν είναι δικό μου αυτό το διάγραμμα, το βρήκα από την επιστημονική βιβλιογραφία και όταν χαράσουμε τις καμπύλες απόδοσης για κάθε μία από αυτές τις αλληλευτικά είδη, όχι σύμπτωση δεν έχουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να συμπέσουν ποτέ. Είναι αδύνατον. Στη θεωρία, αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τόσα πολλά μέτρα ώστε να φαίνεται η αλληλεία ότι είναι σχεδόν ενός είδου, θα, θα μπορούσε να γίνει, αλλά αυτό είναι ουτοπία και θα χάσουμε χρόνο τον οποίο δεν υπάρχει λόγος να χάσουμε, δεν θα το σύστηνα ποτέ. Θα πρέπει λοιπόν τη δεδομένη χρονική στιγμή να κάνουμε μία επιλογή. Εάν κάποιο αλεύει το πρώτο είδο, θα πρέπει να υπεραλιεύσουμε το είδο 2 και να υποαλλιεύσουμε το είδο 3. Ή να επιλέξουμε άλλη εναλλεκτική, να αλιεύσουμε το είδο 2 και να υποαλλιεύσουμε το είδο 1 και το είδο 3. Αυτό δεν είναι πονοκέφαλος, είναι πώς έχουν τα πράγματα εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε τους κανόνες αυτούς. Έχουμε πάντα την τάση να πιστεύουμε ότι είναι διαφορετική η αλία. Δεν είναι διαφορετική η αλία. Είναι μια οικονομική δραστηριότητα όπως όλες οι υπόλοιπες. Και στην οικονομία η καμπύλη που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το διάστημα παράδειγμα που μαθαίνουμε όλοι μας όταν κάνουμε πρώτο έτος οικονομικό. Το, ε, των κανονιών και του βουτύρου. Μία χώρα μπορεί να παράγει ή μόνο κανόνια ή μόνο βούτυρο ή ένα συνδυασμό των δύο που σου δείχνει όμως τις καμπύλες ποιο είναι το μέγιστο της παραγωγής που μπορούμε να έχουμε σε μια χώρα. Μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό στις στατιστικές καμπύλες για την αλία. Βεβαίως και μπορούμε. Στο κάτω διάγραμμα έχουμε το ίδιο παράδειγμα προηγουμένω, αλλά με δύο είδη. Το είδος α και το είδος β. Τα μέγιστα δεν συμπίπτουν Επομένως, τι πρέπει να κάνει αυτός που διαχειρίζεται την αλία. Ο διαχειριστής της αλίας θα πρέπει να δημιουργήσει μια καμπύλη δυνατοτήτων παραγωγής σαν αυτή που έχουμε στα δεξιά, που έχει προκύψει από αυτές τις ποσότητες, όπου προφανώς ε, δεν ξεκινούμε από το μηδέν, ξεκινάμε από τη μέγιστη βιώσιμη υπόδοση για το καθένα από τα δύο και μπορούμε να κάνουμε αυτό το συνδυασμό. Ή να αλλιεύσουμε το μέγιστο για το είδος β και να υπολέψουμε το α ή το αντίστροφο. Δεν μπορούμε όμως να βελτιστοποιήσουμε και τα δύο είδη ταυτόχρονα. Και αυτό, όσο πιο γρήγορα το αναγνωρίσουμε με σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να φτάσουμε στη σωστή ιδέα της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης ως στόχο. Και εδώ επανέρχομαι και στο πρώτο μου ερώτημα. Μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό σε όλα τα είδη. Ναι, μπορούμε και έχει γίνει στο παρελθόν. Διότι έχουμε περάσει στη δεύτερη ορασική περίοδο πλέον και θυμάμαι τι έλεγε η ΝΑΦΟ, ε, μάλλον η ICNAF που είναι ο προκάτοχός της. Στα αλλιεύματα της George Bank που είναι στο διάστημα μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών οι αναλύσεις που έγιναν για ένα είδος δεν ήταν καλές, διαπιστώθηκε και αυτό προέκυψε από μια προσαρμογή που έγινε σε μια μελέτη στην οποία ελήφθη υπόψη το σύνολο της αλλιευτικής προσπάθειας για όλα τα βαθυπελαγικά είδη και για το πότε μπορούμε να έχουμε μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Τότε που τα μοντέλα αυτά θεωρούνταν ακόμα αξιόπιστα και ίσως θα έπρεπε να τους προσδώσουμε λίγη από την αξία που είχαν στο παρελθόν. Αν θέλουμε να έχουμε μέγιστη βιώσιμη απόδοση για το σύνολο των αλλιευτικών ειδών, ε, αυτό έγινε στο παρελθόν και για κάποια χρόνια ρυθμιζόταν έτσι. Είναι λίγο πιο συντηρητικό από το να ρυθμίσουμε το F maximum ε, και τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Η απάντηση είναι όχι θα είχαμε ε, διπλό ποσοστό. Ένα για τα είδη μεμονωμένα και ένα διαφορετικό ποσοστό για το σύνολο των ειδών. Διαφορετικό είναι τα στοιχεία που θα λάβουμε όταν έχουμε κάθε είδος και διαφορετικό ποσοστό θα έχουμε από το σύνολο. Και το ποσοστό είναι κατώτερο από το αν προσθέσουμε το F maximum του κάθε είδους. Ουσιαστικά πρόκειται για μία πρόταση που δεν είναι πιο συντηρητική από την άλλη, είναι απλώς πιο λογική και πιο ρεαλιστική. Και αυτό κατά την άποψή μου είναι αυτό που έχει σημασία και προασπίζομαι εγώ εδώ. Το να φτάσουμε δηλαδή στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση για τα είδη, ναι μεν, αλλά για να το ξαναπώ. Η απάντηση είναι θετική καταφατική. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε ως σημεία αναφορά είναι εκτιμήσεις και δεν είναι ακριβές τιμές. Επομένως δεν μπορούμε να είμαστε δογματικοί, ιδίω όταν προτείνουμε υπερβολικές περικοπές. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα περιοριστικά μέτρα πρέπει πάντα να υιοθετούνται με φιδό. Και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όχι μόνο για θέματα διατήρησης του αποθέματος, αλλά και για το πώς εφαρμόζονται και πώς ε, ε, επηρεάζουν τους αλείς, που είναι ο, ο τελικός φορέας. Στη συνθήκη, βάσει των όρων, γίνονται απόλυτα σεβαστά αυτά και θα μπορούσαμε να το συζητάμε για ώρα. Αλλά εγώ ε, για μένα δεν έχει σημασία από πού είναι ένας ψαράς, όλοι ίσοι είναι. Δεν θα πρέπει να υπάρχει όμως υπερβολικό κόστος, ιδίως σε ε, υπερβολικές περικοπές, συγγνώμη, ιδίως σε περιοχές ε, χαλεπές όπως αυτές που βιώνουμε και επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχει περικοπή στο εισόδημά τους. Εάν δεχτούμε ότι οι περικοπές δεν μπορούν να πάνε πέρα από το 10% δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα λάβουν και δεν θα τους κάνουμε καμία περικοπή πέρα από αυτό, γιατί δεν θα μας πιστέψουν. Διότι αν κάνουμε περικοπές και βάλουμε περιοριστικά μέτρα κατά τρόπον ώστε να τους οδηγούμε σε αδύνατες καταστάσεις, σίγουρα δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα και από εκεί και πέρα οι νομοθέτες ε, χάνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών τους. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι εάν κάνουμε τα εξή μπορεί να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Αν το εφαρμόσουμε για όλη την ε, αλία και όχι είδο προς είδο, αν η μέγιστη βιώσιμη απόδοση, που νομίζω ότι αυτό λέει το πνεύμα του νομοθέτη της ε, ε, δήλωσης του Johannesburg, να εφαρμόζουμε αυτή τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση για όλα τα είδη. E και επιμένω, δεν είναι απλή ε, αλία γάδου και μερλούκιο. Υπάρχουν κάποιες ε, πελαγικές ε, τράτες που μπορούν να αλλιεύουν ένα μόνο είδος, αλλά οι περισσότεροι δεν μπορούν. Εάν εφαρμόζουμε το σύστημα αυτό, θα πρέπει να εφαρμόσουμε και ένα διαφορετικό σύστημα ελέγχου. Το παρόν σύστημα είναι πολύ δαπανηρό, πολύ περίπλοκο και δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό. Και εάν χρησιμοποιήσουμε μία τεχνική που είναι προσαρμόσιμη. Δηλαδή, να κάνουμε το εξής. Να δούμε τι είναι αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε καταρχάς. Αν εγώ έπρεπε να διαχειριστώ τα ίδια σαν ήταν δικά μου, που δεν είναι βέβαια, αλλά αν έπρεπε να τα διαχειριστώ εγώ, θα έλεγα ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε ασφαλή βιολογικά όρια. Και όταν μιλάμε για ασφαλή βιολογικά όρια, σημαίνει να είναι ασφαλή, να μην υπάρχει πρόβλημα για την ε, παραγωγή, μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη ή μικρότερη, αλλά να υπάρχει μια κάποια ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή όμως, εάν ε, για παράδειγμα ε, προτείνουμε για το μερλούκιο να φτάσουμε στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση στο 2015, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μία μείωση κατά 26% της αλληλευτικής προσπάθεια ας για να φτάσουμε μόνο σε ένα 4% μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Αυτό είναι πολύ δυσανάλογο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Να κάνουμε μείωση 26% για να φτάσουμε σε μια βελτίωση της τάξης του 4% σημαίνει ότι θα πρέπει να συνειδητοποιούμε πλήρως τι επιβάλλουμε στους πολίτες που ε, ζουν βάσει της αλληλεία του συγκεκριμένου είδους. Εγώ πάντα λέω ότι το σύστημα των ποσοστώσεων δεν είναι σωστό, δεν είναι καλό, διότι αν εδώ δούμε τα τρία είδη που αναφέρουμε, εάν ρυθμίσουμε με ποσοστώσεις θα πρέπει να έχουμε 1, 2, 3 και μετά ε, να έχουμε τα μέτρα 4 και 5 για να μην έχουμε επιπτώσεις από το ένα στο άλλο. Ενώ αν ρυθμίσουμε συνολικά την αλληλευτική προσπάθεια θα έπρεπε να λάβουμε ένα μέτρο για όλα. Γιατί έτσι προσαρμόζουμε αυτόματα τη θνησιμότητα αναείδος και τεχνικώς αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό λοιπόν ήθελα να σας πω και νομίζω ότι με αυτό εξάντλησα και το χρόνο μου. Ε, κατά πόσον προλαβαίνουμε, βεβαίως και μπορούμε. Ε, μέχρι τώρα είχαμε κάποια είδη τα οποία είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε ανασύσταση των ειδών. Για κάποια αποθέματα θα πρέπει να γίνει μια επιπλέον προσπάθεια, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, αλλά αυτό που λέω είναι ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να προχωρήσουμε σταδιακά, ε, να είμαστε αποφασιστικοί και να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση για όλα τα είδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με λογικό τρόπο και με τρόπο ο οποίος θα είναι κοινωνικός αποδεκτός. Έτσι, μπορούμε να απαντήσουμε καταφατικά στο ερώτημα ε, για το αν προλαβαίνουμε. Μπορούμε και σας ε, ε, επισημαίνω ότι αυτό δεν ε, θα πρέπει να γίνει μια, ένα πρόσχημα για να μην γίνει τίποτα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρα. Ε, όπως θα βλέπετε την εξαντλήσατε τη μισή σας ώρα, επομένως δεν ήταν και τόσο πολύ ο χρόνος που σας είχαμε δώσει στη, να μιλήσετε αρχικώς. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν λίγο δύσκολο να την παρακολουθήσουμε, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και μας εξηγεί πάρα πολλά πράγματα για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Στη συνέχεια θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μαρτίν Παστόρ, ο οποίος είναι διευθυντής του Κέντρου Θαλάσσιας Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Βάγκε Μίνκεν, στο Κέντρο Έρευνας ε, των Κάτω Χωρών. Να καλωσορίσω και εσάς και σας δίνω το λόγο. Δεν ξέρω αν θα έρθετε στη θέση του κυρίου Λόπεθ Βέγκα. Uh, Ευχαριστώ που με καλέσετε να σας παρουσιάσω εδώ το θέμα των ε, αντικειμενικών στόχων για τη διαχείριση της αλίας. Το όνομά μου είναι Μάρτιν Παστός και βρίσκομαι εδώ υπό δύο ιδιότητες. Καταρχάς ως Προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την διαχείριση της αλίας και έχω εκτελέσει βουλευτικό ρόλο εδώ και αρκετά χρόνια. Η άλλη μου ιδιότητα είναι ότι εργάζομαι σε ένα νέο ερευνητικό κέντρο στην Ολλανδία, στο κέντρο για την θαλάσσια πολιτική, το οποίο ερευνητικό κέντρο εξετάζει ολοκληρωμένες λύσεις για μία ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Υπό αυτή την ιδιότητα ασχολούμαι με την χωροταξική, θαλάσσια, με τη χωροταξική μελέτη των θαλασσών και άλλα παρόμοια ερευνητικά προγράμματα. Σήμερα όμως θα μιλήσω για την διαχείριση της αλίας και τον ρόλο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης ως πιθανού στόχου η ουσία της ε, παρουσίασής μου αναφέρεται στο ρόλο των επιστημόνων και στο πώς ε, ανταποκρίνονται, πώς αντιδρούν οι οικονομικοί ρυθμιστές, οι οικονομικοί φορείς σε όλο αυτό το πλέγμα των ε, κανονισμών. Το βασικό ερώτημα το οποίο θέτω είναι παρόμοιο με αυτό του προηγούμενου ομιλητή. Εάν δηλαδή η μέγιστη βιώσιμη απόδοση είναι ο κατάλληλος στόχος για τη διαχείριση της αλίας. Ε, άλλοι λένε ότι ε, το στοιχείο αυτό ε, είναι πάρα πολύ χαμηλό, δηλαδή η μέγιστη βιώσιμη απόδοση τίθεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα ε, αυτό είχε ελεγχθεί όταν το, γινόταν επεξεργασία του, της σύμβασης για το δίκαιο της, ε, των θαλασσών, το δίκαιο της θαλάσσης πριν από πολλά χρόνια. Άλλοι λένε ότι είναι υπερβολικά υψηλό. Το θέμα είναι, είναι η σωστή ε, λύση, είναι σωστό στόχος, είναι μια πανάκια. Όχι, πανάκια δεν είναι, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο για να δείξει την κατεύθυνση της σωστής διαχείρισης. Και η κατεύθυνση κατεύθυνση την οποία ακολουθούμε στις ε, συζητήσεις για την μέγιστη βιώσιμη απόδοση δείχνει ότι επιδιώκουμε μια χαμηλότερη θνησιμότητα των αποθεμάτων των ε, ψαριών, των ε, λιευμάτων. Όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν είναι τόσο πολύ τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά αυτό που μας αφορά είναι το πώς ε, ε, καταλήγουμε σε αυτά τα στοιχεία. Αριστερά βλέπετε έναν ε, πύργο απομονωμένο, απομακρυσμένο. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτόν τον, στον υψηλό πύργο των ερευνών και των στοιχείων και δεξιά βλέπετε την άλλη εικόνα, μια ομαδική προσπάθεια, ένα διάλογο όπου γίνεται μια αξιολόγηση της ποιότητας των σημείων αναφοράς. Για μένα όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, συνεργασία, διαφάνεια, αξιοπιστία, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να υπολογίσουμε τα σωστά σημεία αναφοράς. Η θεωρία είναι των MSI, δηλαδή των ε, μέγιστων βιώσιμων επιδόσεων, είναι πάρα πολύ απλή. Εάν έχουμε πάρα πολύ ψηλή αλία, δεν έχουμε αλιεύματα. Εάν έχουμε πολύ λίγη, θα έχουμε πολλά αλιεύματα. Κάπου μεταξύ των δύο αυτών άκρων βρίσκεται ο, ο ισοσταθμισμένος δείκτης της μέγιστης βιώσιμης απόδυσης. Ε, το θέμα είναι ότι σε, αυτή την, σε αυτό το διάγραμμα πρέπει να επισέλθει και το στοιχείο του κόστους. Όσο πιο αποδοτική, τόσο πιο ακριβή. Όσο λιγότερο αποδοτική, τόσο και πιο φτηνή, φτηνό το κόστος. Και πάντοτε όσον αφορά την ελληνική απόδοση, η, ο δείκτης μέγιστη βιώσιμης απόδοξης βρίσκεται πάντοτε κλείνει προς τα αριστερά. Είναι λοιπόν πολύ καλά, καλύτερα να ασχοληθούμε με το στοιχείο της ε, μικρότερης ε, ε, θνησιμότητας των αλλιευμάτων παρά της μέγιστης απόδοσης. Τώρα, ο δείκτης της μέγιστης κοινωνικής απόδοσης βρίσκεται προς τα δεξιά της καμπύλης της ελευτικής προσπάθειας. Αυτά λοιπόν για τη θεωρία. Στην πρακτική όλα αυτά τα στοιχεία είναι περίπλοκα, δημιουργούν μία περιπλοκότητα και θα σας εξηγήσω γιατί. Έχετε τρεις δείκτες, την μέγιστη βιώσιμη απόδοση, την μέγιστη οικονομική και τη μέγιστη κοινωνική απόδοση. Έχετε την έννοια της απόδοσης, δηλαδή το αλίευμα το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί από το συνολικό απόθεμα και το δεύτερο είναι, όπως σας είπα, το στοιχείο της θνησιμότητας, το οποίο συνδέεται άμεσα με τις ε, βιώσιμες αποδόσεις. Αυτή λοιπόν είναι, η, είναι το σημείο εκκίνησης ε, για την επεξεργασία του συστήματος. Και το τρίτο στοιχείο του MSI είναι η βιομάζα. Ο αριθμός των ψαριών στη θάλασσα. Αυτά τα τρία στοιχεία, αυτές οι τρεις πτυχές ε, της βιώσιμης, μέγιστης βιώσιμης απόδοσης δεν ορίζονται επακριβώς στον κανονισμό. Ε, βάσει της δήλωσης του Johannesburg, ο στόχος μας είναι να διατηρήσουμε αποθέματα σε ένα επίπεδο το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει στην παραγωγή της μέγιστης ε, βιώσιμης απόδοσης. Γενικά όμως αυτό το οποίο διαπιστώνεται σε κείμενα όπως το δικό μου αλλά και στο σχέδιο ψηφίσματος και στα, στη σκηνή αλληλευτική πολιτική είναι ένα μείγμα μεταξύ της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης με την έννοια κάποιας βιομάζας, κάποιας έννοιας βιομάζας ή αριθμού αλλιευμένων ψαριών και από την άλλη πλευρά ε, την ερμηνεία της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης σε σχέση με τη θνησιμότητα των αλλιευμάτων. Εάν σκεφτείτε ε, βασικά προς την κατεύθυνση της βιομάζας θα πρέπει να λάβετε υπόψη την αντίδραση του φυσικού συστήματος ε, με τις παράμετρους της φύσης, δηλαδή τις φυσιολογικές παραμέτρους. Εάν τώρα σκεφτείτε προς την κατεύθυνση της θυσιμότητας, πρέπει να λάβετε υπόψη τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητα. Δύο πλευρά, πλευρές λοιπόν υπάρχουν δύο πτυχές βασικές. Η μέγιστη βιώσιμη απόδοση, έτσι όπως χρησιμοποιείται, αναφέρεται σε μεμονωμένα είδη. Δηλαδή, ε, μπορούμε να υπολογίσουμε λίγο πολύ ε, τη βιομάζα, τη mortality, την θνησιμότητα, <laughs> συγγνώμη. Αλλά δεδομένου ότι οι φώκες ας πούμε τρώνε τα ψάρια και αν θέλουμε να υπολογίσουμε και τη βιομάζα και την συνεισιμότητα πρέπει να συνυπολογίσουμε αυτά τα δύο στοιχεία διότι επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η, η φώκια τρώει το γάβρο, αλλά ο γάβρος τρώει και τα οπλανκτόν, τρώει τα, το ζωοπλανκτόν ο γαβ, οι ρέγγες τρώνε το γάβρο ο οποίος έχει φάει το πλανκτόν και ούτω καθεξής. Εάν λοιπόν έχουμε πολλές φώκες οι οποίες τρώνε γάδο, ε, τότε θα είναι δύσκολο να υπολογίσουμε τη βιομάζα, ε, τον αριθμό των, φω, των φωκιών. Και δεν λέω ότι είναι ε, αυτός ο στόχος να υπολογίσουμε τον αριθμό, να βασιστούμε στον αριθμό των φωκιών. Εάν τώρα υπολογίσουμε τη βιομάζα θα δείτε ότι όλες αυτές οι μετρήσεις είναι βιομετρικές. Όσον αφορά την άλλη πτυχή, η ρυθμισιμότητα των ψαριών, εδώ είναι πιο εύκολη εφαρμογή ε, των ε, υπολογισμών ε, στην κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε. Μπορεί λοιπόν η επιστήμη έχοντας όλες αυτές τις περίπλοκες παραμέτρους να υπολογίσει επακριβώς τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Στη θεωρία ναι, αλλά στην πρακτική εφαρμογή μόνο κατά προσέγγιση. Δεν έχουμε επακριβή αριθμητικά στοιχεία τα οποία μπορούμε να συνάψουμε στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Και αυτό που συμβαίνει στην επιστημονική διαδικασία στην Ευρώπη έχουμε κατά προσέγγιση ε, στοιχεία για τη θνησιμότητα και για τη μέγιστη απόδοση. Εξαρτάται βεβαίως και η τοποθεσία που κάνουμε τους υπολογισμούς σε περιοχές ή ζώνες. Αλλά όταν έχουμε ε, ε, όταν υπάρχει μικρότερη ε, θνησιμότητα στα ψάρια, μικρότερα στοιχεία, μπορούμε να πούμε ότι αναφερόμαστε ας πούμε στο τέλος, στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Πριν αρχίσουμε λοιπόν την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης βάσει της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, καλύτερα να συζητήσουμε λίγο την προληπτική προσέγγιση, η οποία εμφανίστηκε προς το τέλος της δεκαετίας του 1990 και προέρχεται αυτό το precautionary approach από μια πολιτική απόφαση που ελήφθη τότε. Αυτό το οποίο συνέβη ήταν ότι οι επιστημονικές ερμηνείες για την προληπτική προσέγγιση μπορούσαν να εφαρμοστούν μόνο σε αποθέματα ε, για τα οποία είχαμε πολλές πληροφορίες. Μόνο εκεί. Ε, καταλήξαμε λοιπόν σε μια προληπτική προσέγγιση η οποία εφαρμόστηκε ε, στα βασικά εμπορικά λιεύματα και στα αποθέματα για τα οποία είχαμε λιγότερες πληροφορίες δεν μπορούσαν να καλυφθούν τόσο καλά. παραδείγματος χάρη τα ε, βενθοπελαγικά είδη, ειδή κλπ. Ε, για τα είδη αυτά για τα οποία είχαμε λιγότερες πληροφορίες, λιγότερα στοιχεία, δεν μπορέσαμε να εφαρμόσουμε τόσο καλά την προληπτική προσέγγιση. Αυτό το σύστημα που εφαρμόστηκε στις, ε, προς τα τέλη της δεκαετίας του 90, ε, είχε επίσης και άλλα μειονεκτήματα. Χαμηλό ποσοστό διαφάνειας και όχι εντελώς αξιόπιστα σημεία αναφοράς. Πολλές συζητήσεις έγιναν τότε ε, επί τη βάση της προληπτικής προσέγγισης και για το ότι δεν είχαν συμπεριληφθεί στην όλη συζήτηση όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη κλπ. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτό το στοιχείο όταν συζητάμε την εφαρμογή τώρα της ε, καινούργιας προσέγγισης, της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Τι σημαίνει λοιπόν η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης MSI. Λιγότερα ψάρια, με αυτό θα πρέπει να ζήσουμε, με αυτή την πραγματικότητα στον 21ο αιώνα. Εγώ πιστεύω ότι ε, γίνεται σιγά σιγά αποδεκτή, αποδεκτό το γεγονός ότι χαμηλές, ε, χαμηλές, ε, χαμηλή θνησιμότητα δημιουργεί μέσο και μακροπρόθεσμα ωφέλη. Αύξηση, ανασύσταση των αποθεμάτων των ειδών. Τώρα, όσον αφορά τα καταπροσέγγιση σημεία αναφοράς, αυτά βασίζονται σε μοντέλα τα οποία δεν είναι πολύ ακριβή. Δείχνουν προς μία κατεύθυνση τα στοιχεία αναφοράς ε, των μέγιστων βιώσιμων αποδόσεων, παρόλο που είναι κατά προσέγγιση και όχι εδρεωμένα, μελιωμένα σε τσιμέντο ας πούμε, δείχνουν μία κατεύθυνση αποδεκτή. Και άλλο ένα στοιχείο επιστημονικό προς, μέσα σε αυτό το πλαίσιο και έχοντας υπόψη τι είναι με την προληπτική προσέγγιση, εγώ πιστεύω ότι ο ρόλος της επιστήμης των επιστημών είναι διευκρινιστικός, είναι κατά πολύ επεξηγηματικός, να εξηγεί, να διευκρινίζει ε, τι είναι γνωστό, τι δεν είναι, ποιοι είναι οι κίνδυνοι εφαρμογή της α στρατηγικής ή της β. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε την επιστήμη ε, σε ρόλο δικαστή για να δικάζει και να βγάζει δικαστικές αποφάσεις ε, για να εκτελέσει σωστά το, το ρόλο του η προσέγγιση αυτή απαιτεί νομιμοποίηση, διαφάνεια και αξιοπιστία. Γι' αυτό η επιστήμη λοιπόν πρέπει να βοηθήσει στην ανάλυση της προσέγγισης μέγιστης απόδοσης. Ε, διότι εμείς θέλουμε να εδραιώσουμε ένα σωστό και κοινό πλαίσιο λειτουργίας. Για μένα λοιπόν η προσέγγιση της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης είναι μία διαδικασία την οποία συζητούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και η οποία δείχνει προς την σωστή ακολουθητέα κατεύθυνση όπως βλέπουμε τώρα και με προγράμματα σε άλλους τομείς όπου οι ε, επιστήμονες, οι, ε, τα ενδιαφερόμενοι φορείς, ε, το και τομείς της οικονομίας και της ε, κοινωνίας ε, προσπαθούν να βρουν μαζί μια κατάλληλη, ένα κατάλληλο πρόγραμμα, μια κατάλληλη πορεία. Και στο τέλος της ε, ημέρας όλοι θέλουμε να επιτύχουμε χαμηλότερες, ε, χαμηλότερα ποσοστά εκμετάλλευσης ε, ε, για να μην συνεχιστεί αυτή η καταστροφική πορεία. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω για τις συζητήσεις που γίνονται μέσα στους επιστημονικούς κύκλους της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Και τώρα μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση. κυρία Λοβέν. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τους δύο μιλητές ε, για τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις τους και σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που τονίσατε ότι ο κύριος ε, Λόπες Βέγκα δεν είναι μόνο ε, βιολόγος αλλά ήταν και υπουργός αλίας της περιφέρειας της Γαλλικίας και είναι και μέλος του Παρτίδο Popular, του Λαϊκού Κόμματος. Ε, είναι λοιπόν, επίσης ο δεύτερος ομιλητής μίλησε από την επιστημονική πλευρά και ε, ακούσαμε με ενδιαφέρον αυτά που είπατε και θα ήθελα τώρα και εγώ να σχολιάσω ορισμένα από τα συμπεράσματά σας. Καταρχάς, ε, παράγραφος 39 της συνθήκης της ε, Λισαβόνας. Όπως είπατε, ξεκάθαρα ότι είναι ο στόχος της αλλιευτικής πολιτικής. Το άρθρο αυτό μιλά για την αγροτική πολιτική και αναφέρεται στην αύξηση της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Αλλά εμείς εδώ μιλάμε για αλία και αλίευματα και όπως όλοι ξέρουμε η αύξηση της αλίας και η αύξηση των αλιευμάτων ε, ε, ε, δυσκολεύεται από την, ε, το γεγονός ε, ότι ε, υπερεκμεταλλευόμαστε και υπεραλλιεύουμε τις θάλασσές μας και πολλά από τα χρήματα των φορολογούμενων διοχετεύονται στο πλεονάζον αυτό δυναμικό της αλίας και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα καταλήξουμε σε μια τεράστια αλλιευτική προσπάθεια χωρίς ψάρια, χωρί αλλιεύματα. Ε, δεν είναι λοιπόν δυνατόν να ακολουθήσουμε εδώ ε, τις διατάξεις της αγροτικής πολιτικής η οποία λέει ε, ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται χι, ζυζανιοκτώνα ή παρασιτοκτώνα ή λιπάσματα. Μπορεί βεβαίως με αυτόν τον τρόπο και με τις διατάξεις της αγροτικής πολιτικής να αυξηθεί η παραγωγή τροφίμων. Όμως, αν εφαρμοστούν αυτά στις θάλασσες και στην αλία δεν μπορούμε να βοηθήσουμε την επιβίωση ή την ανάπτυξη των αλλιευμάτων, το αντίθετο αποτέλεσμα θα έχουμε. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να αναφερόμαστε μόνο στο άρθρο 39 της συνθήκης. Αναφέρεται επίσης ότι στην παράγραφο 3 της συνθήκης αναφέρεται υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρεί η Ένωση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, εκτός από το άρθρο 39 πρέπει να έχουμε υπόψη και την παράγραφο 3. Όσον αφορά τώρα τις μέγιστες αποδόσεις και τη δήλωση του Johannesburg, δεν είναι μια υποχρεωτική, ε, ε, δεν είναι μια υποχρέωση νομικής φύσεως. Ε, αυτό το αναφερόσαστε, αναφερθήκατε στο 1992 όπου δεν γινόταν αναφορά του MSI. Τώρα, στο άρθρο 61.3 λέει ότι θα πρέπει να ε, διατηρούμε την αλία σε επίπεδο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη βιώσιμη απόδειξη και το άρθρο 19 λέει πρέπει να εκπονούμε μέτρα τα οποία λαμβάνουν υπόψη τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα για την αλληλεία έτσι ώστε να εφαρμόζονται ε, οι μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις. Αυτά είναι τα νέα στοιχεία που έχουμε, οι νέοι στόχοι. Οπότε, Εσείς προτείνετε το στοιχείο αυτό της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης καλό θα ήταν να μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε σε όλο το οικοσύστημα. Ταυτόχρονα αναφέρεστε και στις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Εφόσον υλοποιηθεί αυτή η μέγιστη βιώσιμη απόδοση για τα πιο ε, ευαίσθητα ή ε, ψάρια, αλλιεύματα ή τα, τα αλλιεύματα τα οποία κινδυνεύουν. Έχουμε λοιπόν δύο-τρεις εναλλακτικέ λύσεις. Το ένα είναι να παραμείνει η κατάσταση ως έχει, το status quo και αφήνουμε τα πράγματα να εξελιχθούν μόνα τους. Η άλλη εναλλακτική λύση είναι να εφαρμόσουμε την αρχή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης υπάρχει και μία πρόταση να επικεντρωθεί στις πιο, στα πιο πολύτιμα είδη ή στη μεικτή αλληλεία ή στα πιο ευαίσθητα είδη. Όλα αυτά τα διαφορετικά σενάρια πρέπει να τα εξετάσουμε με προσοχή και πού θα καταλήξουμε. Διότι στην πρώτη οψιόν που έχουμε να παραμείνει η κατάσταση ως έχει, το status quo δηλαδή, είναι το καταστροφικό το σενάριο, το σενάριο που θα μας οδηγήσει στην καταστροφή όσον αφορά το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνική απόδοση. Ενώ όλα τα άλλα σενάρια, συμπεριλαμβανομένου και του πιο αυστηρού, για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα θα καταφέρει, θα επιφέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από την πρώτη οψιόν της αδράνειας. Σύμφωνα με τις καλύτερες εκτιμήσεις, ε, λέει η έκθεση, εάν τα αποθέμα, αν γίνει μάξιμο εκμετάλλευση των αποθεμάτων, θα έχουμε μια μείωση των αλλιευμάτων 20-22 ε, ε, του 70%. Τα κέρδη θα τριπλασιαστούν, τα, το επενδυτικό κόστος θα εξαπλιάσιασει και το κόστος ε, των επενδύσεων θα πρέπει να αυξηθεί περίπου κατά 90%. Σας ρωτώ λοιπόν, τι προτιμάτε εσείς, αυτό το καταστροφικό σενάριο στο οποίο οδεύουμε ή την εφαρμογή των νέων ε, προσεγγίσεων Σχετικά με τα οικοσυστήματα, λέτε ότι τα οικοσυστήματα είναι για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος ε, λειτουργεί για τα οικοσυστήματα. Ε, συμφωνώ με αυτό και πρέπει να σεβαστούμε αυτή την αρχή. Για τον Μάρτιν Παστόρς, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του της ΆΙΣΑΣ, θέλω να ρωτήσω μερικά πράγματα. Καταρχάς, Ποια είναι η απάντησή σας στον προηγούμενο μιλητή ε, που αφορά την εφαρμογή του MSI των μέγιστων αποδόσεων γενικά στα οικοσυστήματα. Είναι δυνατόν αυτό ή όχι. Θέλω να ακούσω την γνώμη ενός επιστήμονα για την ε, ολοκληρωμένη εφαρμογή των μεγίστων αποδόσεων. Ε, όσον αφορά την ε, μέγιστη βιώσιμη απόδοση, οικονομική και κοινωνική απόδοση, η μέγιστη κοινωνική απόδοση μου φαίνεται ότι ε, μπορεί να θεωρηθεί ότι θέλουμε τους, τον μεγαλύτερο αριθμό αλλιέων με τη, που θα έχουν όμως τα χαμηλότερα εισοδήματα. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι οι επιστήμονες θα πρέπει να λαμβάνουν αυτές τις ε, αποφάσεις, ε, να υποστηρίζουν, να συμβουλεύουν και να διευκρινίζουν, ναι, αλλά όχι λίγο αποφάσεων. Στη Φλόριντα είχαν εφαρμόσει, έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα, έναν ε, νόμο που λέει ότι δεν μπορούν να εγκριθούν ποσοστώσεις πάνω από τις μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις και όλοι προσαρμόστηκαν προς ε, αυτόν, στον κανονισμό, προσαρμόστηκαν έτσι. Ε, οι πολιτικοί λοιπόν λαμβάνουν τις αποφάσεις ε, και λένε ότι αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε και εν συνεχή οι επιστήμονες κάνουν τους υπολογισμούς. Ευχαριστώ. Και εγώ απευθύνομαι στον κύριο Λόπες Βέγκα. Θα ήθελα να σας πω καλώς ήρθατε στο, στην ομάδα μας. Στην ομάδα μας, αν κατάλαβα καλά, ήσασταν υπουργό Αλίας. Ε, αν και εγώ θα ήθελα εδώ περισσότερο να ασχοληθούμε με το επιστημονικό επίπεδο, επιστημονική διαβούλευση και όχι τόσο πολιτική. Αλλά αφού είσαστε και πολιτικός, ε, ε, θα αναφέρεστε ασφαλώς και στο άρθρο 39, όπως είπε και η κυρία Λούβε. Αναφέρεται στην κοινή αγροτική πολιτική και συμφωνώ απολύτως μαζί της ότι η πολιτική αλίας γίνεται, εκπονείται βάσει το άρθρο αυτού. Όμως η γεωργία και η αλία δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εάν οι παραγωγοί μας δουλεύουν περισσότερο, έχουν περισσότερα ωφέλη, περισσότερα κέρδη. Εάν οι μας εργαστούν, αλλιεύσουν περισσότερο, δεν ισχύει αυτό, ισχύει μάλλον το αντίθετο. Δεν μπορούμε λοιπόν να χειριστούμε με τον ίδιο τρόπο τα ψάρια και τα γεωργικά προϊόντα. Αυτή η παράγραφος 39 μπορεί, όπως ξέρετε πολύ καλά, και να συμπληρωθεί. Και πολλές φορές ε, θέτουμε στόχους ε, οι οποίοι βασίζονται σε πολιτικές αποφάσεις. Οι στόχοι μας ε, μετααναθεωρούνται, τροποποιούνται και συμπληρώνονται. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι μπορούμε να αναφερθούμε μόνο στο άρθρο 39, αλλά θα πρέπει με περισσότερο ευθύνη να αναφερθούμε και στο δίκαιο των της θαλάσσης, ε, στη σύμβαση για το δίκαιο της θαλάσσης του ΟΗΕ. Ξέρουμε όλοι ότι το 35 των αλλιευμάτων αλλιεύονται βάσει της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Ξέρετε επίσης ότι μας λείπουν σωρία στοιχείων και όταν ρωτώ ε, κατά πόσον τα κράτη συμπεριφέρονται αξιόπιστα και σέβονται αυτά τα στοιχεία φρίτο, φρίτο, διότι μας ε, καταθέτουν, μας λένε στοιχεία ε, τα οποία είναι εντελώς αντίθετα, εντελώς ε, εσφαλμένα και πολλές φορές δεν έχουμε, είμαστε στο σκοτάδι, δεν έχουμε καθόλου στοιχεία από τα κράτη-μέλη τα οποία χρειαζόμαστε, άρα δεν μπορούμε και να κρίνουμε. Ε, άκουσα με προσοχή την εισήγησή σας και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο λαμβάνετε υπόψη το γεγονός ότι τα, πολύ περιορισμένα λιευτικά αποθέματα εκπληρώνουν, δεν εκπληρώνουν σωστά το ρόλο τους στο οικοσύστημα. Πιστεύω ότι και στην, στον αντίποδα η υπεραλίευση δεν σέβεται τους νόμους της φύσης. Ούτε ε, δεν είναι λοιπόν, παρόλο που οι αλείς μπορεί να μην ενδιαφέρονται, να μην τους απασχολεί το θέμα, σωστή η, η καταστροφή των ε, αλλιευμάτων είτε ε, τα μικρά, οι μικρές, τα μικρά αποθέματα είτε η, υπεραλίευση και τα δύο βλάπτουν τη φύση, τη, τη φυσιολογική εξέλιξη. Επίσης, ε, οι ποσοστώσεις ή ας το πούμε διαφορετικά η ελευθερική προσπάθεια είναι πάντοτε υπερβολικά υψηλή. Ε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε στους στόχους μας εάν αφήσουμε αυτή την κατάσταση όπως έχει, με τις περιβολικά υψηλές υποσοστώσεις. Ε, ε, Προσωπικά εγώ πιστεύω ότι αυτά τα οποία έκανε το Συμβούλιο στο παρελθόν, ίσως ήσασταν και παρόν εσείς, ήταν πολύ κοντόφθαλμα, πολύ κοντόφθαλμη αυτή η πολιτική του Συμβουλίου μου ευχαριστήθηκα ιδιαίτερα που αναφέρατε τη μεικτή αλία και είπατε ότι η αρχή της ε, μέγιστης βιώσιμης απόδοσης μπορεί να εφαρμοστεί και στη μεικτή αλία, ενώ μέχρι τότε αυτό το αμφισβητούσαν. Το ερώτημά μου είναι μήπως μπορούμε με την κατάλληλη μεθόδευση συνεργασίας ε, των αλλιέων να αποφύγουμε την αλίευση των αδύναμων ειδών έτσι ώστε να μην κλείνει η περίοδος αλίες υπερβολικά νωρίς. Παραλιεύματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, ε, πάντοτε υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ε, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένες ζώνες ε, αλίες και να μειώσουμε αυτό το πρόβλημα ακόμα περισσότερο. Τονίσατε ότι ο άνθρωπος, ο, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι στο επίκεντρο, βεβαίως, όσον αφορά και την επιστημιστική επάρκεια, αλλά επιμένω, εάν κα, κα, συνεχίσουμε την υπεραλίευση των πόρων μας, των θαλασσών μας, ε, και βρισκόμαστε στο παραπέντε πριν από την καταστροφή θα, θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουμε την πολιτική μας ε, ε, και δεν μπορούμε να επιβιώσει, δεν, δεν μπορεί η ελία μας να επιβιώσει εάν δεν ρυθμίσουμε το, το θέμα των αποθεμάτων. Πιστεύετε ότι ο ελευτικός στόλος είναι, ε, κατά, είναι σωστός το μέγεθος ε, των αλλιευτικών στόλων είναι σωστό, είναι το κατάλληλο για την επιβίωση των αλλιευμάτων ή πιστεύετε ότι πρέπει να θέσουμε υπό αυστηρότερο έλεγχο το στόλο, τους στόλους. Μια διευκρίνηση. Ο κύριος είναι θαλάσσιος βιολόγος, επομένως ε, δεν είναι ε, εδώ ως ε, κάτι άλλο, μόνο ως θαλάσσιος βιολόγος. Γι' αυτό τον έχουμε προσκαλέσει. κυρία Πατράων στη συνέχεια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ τη σημερινή ευκαιρία για να σας πω ότι ε, ευτυχώς που έχουν και επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση κάποιοι Υπουργοί Αλίας. Και ε, βλέπουμε την αξία αυτού από τις ε, πολύ καλές ε, παρεμβάσεις που ακούσαμε. Ε, δεν θέλω να μακρηγορήσω, διότι προτιμώ να υποφεληθώ και άλλο από τους δύο εμπειρογνώμονε και τις γνώσεις τους. Από όσα άκουσα πάντως, ε, έχω έντονα την εντύπωση ότι το MSY ε, αυτή τη στιγμή και κατά τη γνώμη των δύο προσκεκλημένων είναι ένας προσανατολισμός μόνο. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία προς το παρόν. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε στο επίπεδο της ε, εφαρμογής ε, των ε, μέτρων από επιστημονικής πλευράς, ούτως ώστε, μάλλον τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να γίνουν ακριβέστερα αυτά τα επιστημονικά στοιχεία. Ε, εφόσον είναι ε, θαλάσσιοι βιολόγοι, θα μπορούσαν ίσως ε, να μας κατευθύνουν, να μας πούμε ποιο τρόπο μπορούν να γίνουν πιο ακριβή αυτά τα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τόσο ώστε να μπορέσουμε μεταγενέστερα να ε, υλοποιήσουμε το MSY. Η δεύτερη ερώτηση ε, είναι η εξής αυτή η καταπροσέγγιση εκτίμηση που μπορεί να εφαρμοστεί και, στις ε, καθαρέ, και στα καθαρά και στα μεικτά αλλιεύματα, Δηλαδή το MSY μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τα δύο είδη αλλιευμάτων όταν ε, γίνουν ακριβέστερα τα επιστημονικά στοιχεία. με στόχο το 2015 για την εφαρμογή του MSY πιστεύω ότι έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας αν εφαρμοστεί το MSY μόνο για τα καθαρά αλλιεύματα και όχι για τα μεικτά. Ίσως χρειαστεί να προβλέψουμε και μία περίοδο σταδιακής εκνοής phasing out. Μπορείτε να μας δώσετε και άλλα επιστημονικά στοιχεία ε, για την εκτίμησή σας ε, με την ιδιότητά σας σε σχέση με το MSY. Ευχαριστώ κύριε Αντρές Μπαρία. Ήρθα λίγο καθυστερημένη, αλλά διαπιστώνω ότι ο πρώτος και ο δεύτερος ομιλητής μας είπαν κοινά πράγματα. Ε, άκουσα τη δεύτερη ομιλία του δε, ολόκληρη και άκουσα να αναφέρεται στο MSY μόνο για την αλληλεία ενός είδου, και είπατε ότι μπορούμε να το εφαρμόσουμε μόνο με προσεγγιστικό τρόπο, είναι λίγο διάφανο το σύστημα και είναι ελάχιστα αξιόπιστο. Εάν πρόκειται για μαθηματικό τύπο, το οποίο δεν είναι ούτε ιδεολογία, ούτε κάποια ευαισθησία, ούτε κάτι άλλο, είναι ένας μαθηματικός τύπος ο οποίος οδηγεί σε τεχνικά, ε, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε, που είπε και ο δεύτερος ομιλητής, είναι να το συνειδητοποιήσουμε, το οποίο μας φαίνεται καλό, να προσπαθήσουμε να μην έχουμε υπερεκμετάλλευση, αλλά όχι να αποφύγουμε την εκμετάλλευση, την υπερεκμετάλλευση μόνο. Την η οικονομική και κοινωνική πτυχή θα μπορούσαμε να την καλύψουμε με περισσότερο χρήματα και περισσότερο χρώμα. Αλλά το τεχνικό ε, σκέλος πώς θα το εφαρμόσουμε. Θα ήθελα να μου πείτε πώς μπορούμε να προσδώσουμε αξία σε αυτό το μαθηματικό τύπο, ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά στοιχεία που διαθέτει για την επόμενη κοινή ελευτική πολιτική. Διότι πρόκειται για ένα μαθηματικό τύπο ο οποίος επινεώθηκε τη δεκαετία του 50 και εξακολουθεί να έχει διάφορα προβλήματα στην εφαρμογή του. Ευχαριστώ κύριο Στίβενσον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δύο μιλητές για τις παρουσιάσεις, αλλά για το θέμα του MSY είχαμε ε, με τον Klein Earth σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον γεύμα εργασίας και συζητήσαμε αυτό το θέμα. Για να επιτύχει κανείς το MSY θα πρέπει να καταφέρει και τις δύο πτυχές, ε, δηλαδή την θνησιμότητα ε, και την βιομάζα του αποθέματος γεννητόρων. Να αναπαραγωγήσουμε. Ε, νομίζω ότι ε, για την εφαρμογή των μέτρων μάλλον μιλάμε για το τέλος του 2013 και όχι την αρχή. Είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας, ώστε να ε, επιτύχουμε όλες, ε, να σημειώσουμε επιτυχία σε όλες τις διαφορετικές πτυχές της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αν μέχρι το 2015 μπορούμε να καταφέρουμε το FMSY για σε σχέση με τη θνησιμότητα δηλαδή και αν υποθέσουμε ε, ότι για τη βιομάζα θα τα καταφέρουμε μέχρι το 2020, ζητώ συγγνώμη για όλα αυτά τα ακρονίμια που χρησιμοποιώ, αλλά σε αυτή την επιτροπή είναι must. Για πώς μπορούμε να επιτύχουμε ε, και αυτούς και τους δύο στόχους, εφόσον υπάρχει μια σταδιακή απαγόρευση των απορρίψεων για ε, συγκεκριμένο αριθμό ειδών ε, αναχρόνων και δεδομένης έλλειψης επαρκών επιστημονικών στοιχείων για κάποια είδη. Βάσει των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, όπως μας είπε ο κύριος Έστη το γεύμα εργασίας, ε, το σύνολο των απορρίψεων αυτή τη στιγμή στα ενωσιακά ύδατα είναι 1,7 εκατομμύρια, δηλαδή 23% του συνόλου των αλλιευμάτων. Εάν δεν μπορούμε να καταφέρουμε αυτό, μα πώς το καλό... Ε, θα ε, καταφέρουμε το BMSY, αφήστε το FMSY. Δεδομένου του χρονικού περιορισμού. γιατί πρόκειται για βασικού στόχου τη κοινή αλληλευτική πολιτική, αλλά μήπω είναι υπέρμετρε φιλοδοξίε. Εγώ θα ήθελα να γνωρίζω στην πράξη πώ θα το κάνουμε αυτό, πώ θα το καταφέρουμε. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μια μικρή παρέμβαση με προκάλεσε άλλωστε η κυρία Λεβίν. Πράγματι, στην αξιολόγηση αντικτύπου γίνονται διάφορε αναλύσει για τι διάφορε εναλλακτικέ λύσει και μεταξύ αυτών η χειρότερη είναι ε, το status quo. Και δεν νομίζω ότι το status quo αποτελεί εναλλακτική λύση για τον οποιονδήποτε αυτή τη στιγμή. Αλλά η επιλογή που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αυτή που προτείνει η αξιολόγηση αντικτύπου. Υπάρχουν κάποιε άλλε εναλλακτικέ λύσει που είναι περισσότερο σταδιακέ και σε αυτό αναφέρθηκαν κάποιοι από του ομιλητέ. Δηλαδή υπάρχουν ε, μικρότερε κοινωνικο-οικονομικέ επιπτώσει και στο 2020 θα φτάσουμε στο ίδιο αποτέλεσμα για το RMS. Και γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να μα εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί επέλεξε την πιο ακραία λύση, αυτή που είναι αδύνατη αδύνατη, αυτή την οποία δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε και η οποία προφανώς, αυτό το λέει η αξιολόγηση αντικτύπου και το αναγνώρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δημοσίω, είπε θα διαλέξει όποια θέλει γιατί είναι δικαίωμά τη. Εντάξει, δικαίωμά τη είναι, αλλά αυτή δεν προτείνεται στην αξιολόγηση αντικτύπου και την έχω διαβάσει λέξη-λέξη την αξιολόγηση αντικτύπου. Δεν πρόκειται λοιπόν να δεχτώ τίποτα, το μελέτησα πολύ καλά το ζήτημα. Εάν λοιπόν το 2020 με άλλες πιο σταδιακές εναλλακτικές λύσεις και με λιγότερες επιπτώσεις φτάνουμε τελικώς λίγο πολύ στο 80 κάτι της 100 του RMS για τα αποθέματα, ίσως καλύτερο θα ήταν να επιλέξουμε άλλες λύσεις και όχι αυτές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να κάνουμε για την εξή ερώτηση όμως. Δεδομένου ότι υπάρχουν αβεβαιότητες και αμφίσιμα στοιχεία από τα επιστημονικά δεδομένα που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή για να έχουμε ε, κατάλληλη μέγιστη βιώσιμη απόδοση για όλα τα είδη ε, το 2020. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον το να επιλέξουμε κάποια ελάχιστα για να φτάσουμε στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση σταδιακά. Και φαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του 2015 και του 2020, γιατί υπάρχουν κάποια είδη που μπορούν να φτάσουν στη σωστή μέγιστη βιώσιμη απόδοση το 2015 και κάποια την έχουν ήδη. Να καθορίσουμε λοιπόν και στο βασικό κανονισμό τις ε, προληπτικές ελάχιστες παραμέτρους που θα μπορούσαμε να έχουμε και στις οποίες δεν θα πρέπει να φτάσουμε ε, σε καμία περίπτωση. Το να έχουμε προληπτική βιομάζα, προληπτική θνησιμότητα, βέβαια με στόχο πάντα να φτάσουμε στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση που έχουμε καθορίσει. Και επίσης εκκρεμεί και μια ερώτηση που σας είχα θέσει τις προάλλες, το πώς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέτει το η μέγιστη βιώσιμη απόδοση σε αλία πολλαπλών αδών. Όπω είδαμε υπάρχουν πολλέ εναλλακτικέ λύσει και επειδή ακόμα δεν μου απαντήσατε στην ερώτησή μου, θα ήθελα να ξέρω πώ ε, θεωρεί ότι θα εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση για τα ε, αλλοία πολλαπλών ειδών. Κύριε Πένα, έχετε το λόγο τώρα και κατόπιν θα δώσω το λόγο εκ νέου στους δύο ομιλητέ για να απαντήσουν στι ερωτήσει που του ετέθησαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να ε, εκφράσω την ικανοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι μπορούμε να συμμετέχουμε σε μια τόσο επικοδομητική συζήτηση. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε κάποια από τα θέματα στα οποία αναφέρθηκαν οι δύο πρώτες παρεμβάσεις και μετά θα απαντήσω και στις υπόλοιπε ερωτήσεις. Η μέγιστη βιώσιμη απόδοση δεν είναι νομική υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, το δεχόμαστε, αλλά θα θέλαμε να είναι. Γι' αυτό ακριβώς προτείνουμε σε ένα κανονισμό η έννοια αυτή, που αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο πολιτική παρανομική υποχρέωση, να μεταφραστεί αυτή η πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε νομική υποχρέωση. Γι' αυτό τη συμπεριλαμβάνουμε σε αυτόν τον κανονισμό. Ε, το κατά να ε, προσδιορίσαμε στόχους. Όχι, υπάρχουν δύο απαντήσεις, ίσως η πρώτη δεν είναι και τόσο πιστική, αλλά θα την επαναλάβω. Η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως γνωρίζετε και από άλλα θέματα, όπως αυτό της περιφερειοποίησης, έκανε ένα πολύ αναλυτικό έλεγχο της πρότασης και αφού διασφάλισε ότι αυτό που έχουμε προτείνει ως στόχοι ε, Εάν διαπίστωνε ότι δεν ανταποκρίνονται στο άρθρο 39 της συνθήκης, τότε η νομική υπηρεσία δεν θα μας επέτρεπε να τους εφαρμόσουμε. Υπάρχει όμως και μία εξήγηση η οποία έχει λίγο περισσότερη βάση και θα ήθελα να σας την αναλύσω και αυτή. Ο στόχος της αλίας θα πρέπει να είναι φυσικά οι στόχοι του άρθρου 39, που όπως γνωρίζετε είναι μία σειρά από πολυπίκυλους στόχους και μεταξύ των οποίων δεν υπάρχει καμία ιεράρχηση. Δηλαδή δεν μας λέει η συνθήκη ότι κάποιος από τους στόχους είναι πιο σημαντικός από τους υπόλοιπους. Όλοι είναι και πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των. Μέχρι τώρα στην κοινή ελευτική πολιτική και στον παρόντα κανονισμό δεν αντιμετωπίσαμε ποτέ πρόβλημα στο να μεταφρέσουμε τους στόχους του άρθρου 39 που είναι πανάρχαιοι. Είναι αυτό που είχαμε αυτή εξ αρχής στη συνθήκη της Ρώμης ε, και δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα να τους μεταφράσουμε στους διάσημους ε, τρεις ε, στόχους βιολογικής, οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας και νομίζω ότι εκεί δεν υπήρχε πρόβλημα. Το πρόβλημα προκύπτει όταν βρισκόμαστε σε περιπτώσεις και δυστυχώς είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ισορροπία. Έχουμε πάρα πολλά αποθέματα, υπάρχουν πάρα πολλά ιδιά ε, <coughs> για τις οποίες δεν υπάρχουν υψηλά εισοδήματα, δεν υπάρχουν καλές τιμές για τους καταναλωτές, δεν υπάρχουν επίπεδα ε, κατάλληλα πρόσβαση για του αλληλεί και ούτω καθεξή. Επομένω, το μεγάλο πρόβλημα τη κοινή αλληλευτική πολιτική είναι πώ θα οργανώσουμε αυτή τη μετάβαση. Το πρόβλημα δεν είναι να συμφωνήσουμε ω προ την ισορροπία ε, των στόχων μακροπρόθεσμα. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, μεταξύ αυτών. Τουλάχιστον για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υπάρχουν. Όταν όμω πρέπει να λάβουμε αποφάσει βραχυπρόθεσμα για τα πολιτή προγράμματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν όλοι οι στόχοι ταυτόχρονα. Επομένω, πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις ως προς το πού θα δώσουμε προτεραιότητα όταν καθορίζουμε ένα τάκ για την επόμενη χρονιά. Δεν μπορούμε να εγκρίνουμε ένα τάκ το οποίο θα ανταποκρίνεται πάντα σε αυτό που είναι καλύτερο από βιολογική σκοπιά, που θα είναι καλύτερο για, από πλευρά τιμών για τους καταναλωτές και ούτω καθεξής. Αυτή η βραχυπρόθεσμη απόφαση είναι αυτή που δημιουργεί πρόβλημα ως προς τους στόχους. Και εκεί μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιτρέψτε μου κυρία Πρόεδρε να σας επαναλάβω κάτι που είπα και σήμερα το πρωί. Η αναζήτηση της δέουσας ισορροπίας μεταξύ των ε, στόχων αυτών, στην πράξη, στα προηγούμενα χρόνια εφαρμογή της κοινή αλληλευτικής πολιτικής, μας οδήγησε σε πάμπολες βραχυπρόθεσμες υποφάσεις, στις οποίες κυριάρχησαν οι οικονομικοί στόχοι βραχυπρόθεσμα των υπολείπων. Εάν θέλουμε ισορροπία, όλη ισορροπία θέλουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισορροπία θέλει. Αλλά πρέπει να επισημάνουμε ότι στι ετήσιε αποφάσει δεν υπήρχε ποτέ ε, σχεδόν ε, ισορροπία. Πάντα δινόταν προτεραιότητα στον οικονομικό στόχο βραχυπρόθεσμα ει βάρο των υπολείπων. Αναζητούμε λοιπόν ισορροπία. Πώς θα κάνουμε λοιπόν τη μετάβαση. Αυτό προσπαθούμε να νομοθετήσουμε. Αυτό που προτείνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τουλάχιστον κάνει μια απόπειρα να προτείνει, είναι ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, στις οποίες πόρο απόχουμε των πολλαπλών στόχων του άρθρου 39, θεωρούμε ότι η βιολογική ανασύσταση των αποθεμάτων είναι προϋπόθεση για να έχουμε καλή προσχώρηση των αλλιών στον κλάδο και ούτω καθεξής, σε όλους τους υπόλοιπους δηλαδή στόχους. Δηλαδή, να έχουμε ισορροπία στους στόχους βάσει του άρθρου 39, αλλά στη μεταβατική φάση μέχρι να φτάσουμε εκεί πρέπει να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις και εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η ανασύσταση των αποθεμάτων είναι αρχική προϋπόθεση για να επιτύχουμε όλους τους υπόλοιπους στόχους. Ακούσαμε και το επιχείρημα του Ενρίκη Λόπες ε, ε, Βέγκα, ο οποίος έλεγε ότι είναι σχεδόν αδύνατο να φτάσουμε σε βιομάζα μέγιστης βιώσιμης απόδοσης σε όλες τις περιπτώσεις. Ε, σε αυτό συμφωνώ και νομίζω το έλεγα και εγώ σήμερα το πρωί, κυρία Πρόεδρε. Αναφέρθηκα στην περίπτωση του γάδου στη Βόρεια Θάλασσα στην οποία ε, τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα αυτή τη στιγμή, αλλά κάποια δεδομένη χρονική στιγμή ήταν ε, ε, σαφές ότι ακόμα και αν σταματούσαμε την αλληλεία, ακόμα και αν είχαμε μηδενική θνησιμότητα ε, για το είδος αυτό, δεν είχαμε καμία εξασφάλιση ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ανασύσταση μέχρι τους 120.000 τόνους του, της βιομάζας μέχρι τις βιώσιμες απόδοσης που θέλαμε να έχουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε λοιπόν καμία εξασφάλιση, κάνουμε ό,τι και αν κάνουμε, δεν μπορούμε να έχουμε βιομάζα που θέλουμε το 2015. Αυτό που μπορούμε όμως να κάνουμε είναι ότι η θνησιμότητα ανά είδος που αποκρίνεται σε αυτή τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση επιτυγχάνεται. Και εδώ αυτό που έχει σημασία είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και το έλεγα και σήμερα το πρωί, είναι ότι τα πολιετή σχέδια θα πρέπει να γίνουν επί τη βάση της θνησιμότητας αναείδος και όχι της βιομάζας αναείδος. Ε, και εδώ θα καταλήξουμε, όπως είπε σαφές και ο Ενρίκε Λόπες ε, Βέγα, ε, στο γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι μπορεί να το καταφέρουμε μέχρι το 2005 υπάρχει κοινωνικό κόστος και ορισμένες φορές απέχουμε πολύ από τον επιθυμητό στόχο και γι' αυτό θα πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις να ε, λάβουμε δυσανάλογα μέτρα ε, τα οποία μπορεί να είναι επιβαρυντικά και από κοινωνική σκοπιά για να, έχουμε αποκατάσταση ενό είδου. Ποιο είναι το πρόβλημα. Εντάξει, να πάμε σταδιακά. Αλλά μέχρι το 2020, στον οποίο γνωρίζουμε ότι πρέπει να έχουμε στο στόχο, το σταδιακό στοιχείο σημαίνει ότι δεν θα έχουμε λάβει τα αποτέλεσμα, ε, ε, τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε. Το είπε και ο Ερικέ Λοπεσβίδε, Βίδε, δεν είναι πρόσχημα αυτό για να μην κάνουμε τίποτα ό,τι έγινε βαθμιδών στην Αλία σε πολλές περιπτώσεις ήταν πρόσχημα για να μην προχωρήσουμε. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρόταση αυτή αποστέλει ένα σαφές μόνιμα. Ναι, σταδιακά, αλλά όχι ως πρόσχημα για να μην προχωρήσουμε. Και έτσι πρέπει να αντιλαμβάνεστε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί αυτό επιθυμεί. Από εδώ και πέρα, ως προς τη σταδιακή εφαρμογή, φυσικά συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποια καλύτερη απόδειξη ότι όλη η εξέλιξη των πολιετών προγραμμάτων διαχείρισης, που είναι, επιτρέψτε μου την έκφραση, ε, κυρία Πρόεδρε, μνημείο της σταδιακής εφαρμογής. Πρόκειται λοιπόν για ε, τρόπο να διασφαλίσουμε ότι θα προχωρήσουμε μεν σταδιακά, αλλά με ταυτόχρονα εξασφαλισμένα τα αποτελέσματα. Και αυτό κάναμε. Προχωρήσαμε βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο για τα ε, στάδια αυτά. Σταδιακή διαδικασία σημαίνει ότι προχωρούμε σταδιακά, όχι μένουμε στάσιμοι. Και αυτό είναι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έτσι πρέπει να την ερμηνεύουμε. Από εκεί και πέρα. η διαχείριση πολλαπλών ειδών. Βεβαίω, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της κοινή ελευτικής πολιτικής. Ότι έχουμε επικεντρωθεί σε ένα είδος κάθε φορά και το λέμε και μόνοι μα ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην αλληλεία πολλαπλών ειδών. Ε, νομίζω ότι η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι υπέρ των πολλαπλών ειδών. Νομίζω ότι διατυπώνεται σαφώς την πρότασή μας και αν δεν είναι επαρκώς ε, σαφής, σας διαβεβαιώ εγώ ότι είναι προς την κατεύθυνση που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα πολλαπλά είδη δηλαδή. Τώρα, εμείς θα ζητήσουμε από τους ε, επιστήμονες να μας ε, ετοιμάσουν εναλλακτικές εκδοχές. Ε, συμφωνώ με αυτό που είπε και ο πρώτος ομιλητές. Η θνησιμότητα για διάφορα είδη ε, δεν είναι συμβατή και θα πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση. Βεβαίως, Από εκεί και πέρα όμως αυτό που ζητάμε από τους επιστήμονες είναι εναλλακτικέ εκδοχές. Τι γίνεται αν το τάδε είδο φτάσει στην εκτίμηση για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση και τι συμβαίνει στα υπόλοιπα είδη. Και να μας δώσουν εναλλακτικέ εκδοχές για να μας πούνε ποιος είναι ο συνδυασμός ο οποίος σε γενικές γραμμές ανταποκρίνεται στην εφαρμογή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης όπως την αντιλαμβανόμαστε. Υπάρχει και κάτι το οποίο είπε και ο Μαρτίν Παστό και με το οποίο συμφωνώ. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση ω το μαγικό αριθμό που θα μα οδηγήσει στο αποτέλεσμα. Γνωρίζουμε ότι αυτέ είναι φυσικέ επιστήμες, το είπαμε και σήμερα το πρωί, δεν είναι απλά σαφή μαθηματικά, Έχουμε φυσικούς πόρους που έχουν διακυμάνσεις και επομένως μπορούμε να έχουμε προσεγγιστικά την πραγματικότητα. Ποτέ δεν μπορούμε να την επιτύχουμε 100% και επομένως θα πρέπει να κάνουμε μια ευφυή εφαρμογή της έννοιας αυτής αναπερίπτωση θα πρέπει να δούμε βεβαίω σε κάθε είδο ε, πώ ε, έχουμε την εικόνα της, ε, των διαφόρων μορφών εφαρμογής τη μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφή πολιτικός στόχο ο οποίος θα αποφεύγει Επιτρέψτε μου και πάλι την έκφραση, την έλλειψη προόδου γιατί οι μακροπρόθεσμοι στόχοι επειδή ε, είναι κινούμενος στόχος όπως το λένε και οι Άγγλοι και επειδή δεν ξέρουμε ακριβώς που πηγαίνουμε δεν θα πρέπει να αποτελέσουν πρόσχημα για να μην δράσουμε. Ο στόχος της πρότασης είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα σαφή στόχο για το μέλλον χωρίς να λησμονούμε ότι δεν είναι ένας ιερός μαθηματικός αριθμός πρέπει να πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε είδος, ανάλογα με την πολλοπλικότητά του, θα ζητήσουμε από τους επιστήμονες, όπως κάνουμε άλλωστε και στην πρώτη περίπτωση, να μας δώσουν εναλλακτικέ εκδοχές. Και βάσει αυτών των εκδοχών θα πρέπει να επιλέξουμε ευφυώς αυτό που ανταποκρίνεται στο σύνολο της αλληλείας, δηλαδή τον κατάλληλο συνδυασμό μέτρων που να ανταποκρίνονται στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση για την αλληλεία. Εγώ νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο θα το εφαρμόσουμε αυτό ε, στην πράξη θα ε, φανεί από το πρώτο ε, μοντέλο αλίας πολλαπλών ειδών που θέλει να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι η Βαλτική θάλασσα. Επειδή ακριβώς είναι πιο απλά τα πράγματα εκεί, οι επιστήμονες μας είπαν ότι μπορούν για πρώτη φορά να έχουν συστάσεις με εναλλακτικέ εκδοχές για ένα συγκεκριμένο μοντέλο και νομίζω ότι βάσει αυτού θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε λίγο πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Και αυτή η εφαρμογή θα γίνει με ευφυή και λογικό τρόπο. Από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι τουλάχιστον απάντησα σε αυτά που παρουσίασε ο Ενρίκε Λόπεθ Βέγα. Τα θέματα που έθιξε ο Μαρτίν Παστόρς απάντησα ήδη ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με τη βιομάζα ε, και τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση από αυτή τη σκοπιά και όπως σας είπα επιμένω ότι δεν θέλουμε να έχουμε ως εκτίμηση τη βιομάζα για να επιτύχουμε αυτή τη μάζα και να θυσιάσουμε τα πάντα στο βωμό της. Δεν γνωρίζουμε ποτέ και δεν θα γνωρίζουμε ποτέ τι ακριβώς θα κάνει η φύση. Θα πρέπει να ξέρουμε λοιπόν πόσα θα ψαρέψουμε εμείς από αυτά που μας δίνει η φύση και θα δεσμευθούμε να μην ψαρέψουμε πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό αυτού που μας προσφέρει η φύση. Επομένως αυτό θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε γιατί θεωρούμε ότι είναι το πιο λογικό και είναι αυτό το οποίο μας επιτρέπει να μην εξαρτώμαστε από τη φύση για το ε, κατά πόσον θα επιτύχουμε στόχους. Αν έχουμε θνησιμότητα ένα είδος ε, σε κάποιο επίπεδο αλλά για κλιματικούς λόγους η φύση δεν είναι και τόσο γενναιόδερα, μέχρι εκεί μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο. Αυτό αλλάζει με αν επικεντρωθούμε στη θνησιμότητα αναείδος. είδος. Ο Μαρτίν Παστόρ είπε ότι αυτά όλα είναι προσεγγιστικά στοιχεία. Βεβαίω και είναι προσεγγιστικά στοιχεία και σε καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να θεωρήσει ιερά τα στοιχεία που μας δίνει η επιστημονική κοινότητα. Αν δούμε για παράδειγμα τους στόχους που έχουμε αυτή τη στιγμή στα διάφορα σχέδια διαχείρισης τα οποία έχουμε σε εφαρμογή αυτή τη στιγμή, ε, θα δείτε ότι είναι διαφορετική η στόχη μας ως προς το τι θεωρούμε κάθε φορά κατά προσέγγιση ε, τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ε, νομίζω ότι η πρώτη εμπειρία που έχουμε από τα σχέδια αυτά καταδεικνύει ότι δεν θέλουμε οπωσδήποτε να έχουμε ένα ποσοστό το οποίο πρέπει να επιτύχουμε. Στο παρελθόν προσπαθήσαμε να το εφαρμόσουμε με ευφυή τρόπο, με μικρότερη μεγαλύτερη επιτυχία αναπερίπτωση. Ένα ακόμα σημείο στο οποίο αναφέρθηκε ο Μάρτιν Παστόρς είναι αυτό που σας έλεγα και σήμερα το πρωί κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει ένα σύστημα σαν το σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών αυτόματα θεωρεί ως δεδομένο ε, αυτό το οποίο λένε οι επιστήμονες. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι δεν μπορούμε ποτέ να ε, υποχρεώσουμε τους επιστήμονες ε, να λάβουν αυτοί ε, αποφάσεις πολιτικής φύσης που εφαρμόζονται απευθεία στους πολίτες. Δεν ισχύει. Οι συνομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτοί που είναι αρμόδιοι να λάβουν αποφάσεις. Αυτό είναι σαφέστατο και αν υπάρχει κάποιο στοιχείο στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δίνει την εντύπωση ότι εμείς ε, δίνουμε την αρμοδιότητα αυτή στους επιστήμονες, ε, λάθος κάνετε, αποκλείεται να συμβεί κάτι τέτοιο. Με αυτό νομίζω ότι απάντησα. Ε, σχεδόν εξαντλήσαμε τη μία ώρα και τρία τέταρτα. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Λοπεθ Βέγα και κατόπιν στον κύριο Παστόρος για να απαντήσει. Κύριε Λοπεθ Βέγα, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σταθώ στην ε, παρέμβαση της κυρίας Ρούπι. Ελπίζω να πιστεύετε όπως και εγώ ότι η πολιτική είναι λειτουργήμα, δεν είναι επάγγελμα. Και νομίζω ότι αυτό που ακούσαμε από τη δεύτερη ομιλήτρια το να έχει συμμετέχει κάποιος κατάσχει στην πολιτική ζωή σημαίνει ότι αναιρεί το επάγγελμά του, λάθος κάνετε. Εγώ ασχολήθηκα με την πολιτικά, είμαι πυροχνόμονας, είμαι θαλάσσιο βιολόγος αλλά και οικονομολόγος ταυτόχρονα και ασχολούμαι με πολλά σχέδια συνεργασία για την ανάπτυξη, γι' αυτό και έχω και κάποιε ευαισθησίε, οι οποίε ίσω ε, να είναι αντικρουόμενε γιατί δεν είναι απόλυτα πολιτικά ορθές, που να σας πω την αλήθεια αδιαφορώ, εγώ λέω την άποψή μου και κανένας δεν θα μου επιβάλλει τη γνώμη του. Υπάρχει πολιτική ελευθερία. Να σας πω για παράδειγμα ότι ήμουν δύο χρόνια στην Ιεμένη και εκεί η Αλία σαφώς χρειάζεται μείωση της αλληλευτική δυνατότητας, αλλά είναι αδύνατο να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει, διότι ουσιαστικά καταδικάζεται στην ένδια ε, εκατομμύρια ανθρώπους και αυτό είναι αδύνατο. Υπάρχει ένα μέγιστο κοινωνικό-οικονομικό στοιχείο, το ανέφερε και ο κύριος Παστόρ, και ο οποίο πρέπει να λαμβάνεται πότε, ε, ε, υπόψη. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν είπα ότι πρέπει να υπεραλλιεύουμε τα αποθέματα και δεν πρέπει να σεβόμαστε την νομοθεσία. Μπορεί να σας φάνηκε ότι αυτό έλεγα. Αυτό που αμφισβητώ είναι η ημερομηνία του 2015 ως ρεαλιστικός στόχος. Επίσης, δεν είπα σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να υπολογίσουμε μέγιστη βιώσιμη απόδοση για όλο το οικοσύστημα. Εγώ μίλησα για είδη. Εάν υπάρχει αλληλεία βακαλάου θα πρέπει να λαμβάνετε συνολικά υπόψη για το σύνολο του αλλιεύματος. Δεύτερον, Βεβαίω πιστεύω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Σα το είπα ότι δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να παραμείνουν τα πράγματα ω έχουν. Είναι λάθο. Πρέπει να ληφθούν μέτρα σταδιακά αλλά πρέπει να γίνει κάτι. Η κυρία που μίλησε, το συγγνώμη, δεν γνωρίζω το όνομά τη. Ε, δεν είμαι επέτροπο. Αν ήμουν επίτροπο θα είχα τελείω διαφορετική πολιτική, σα διαβεβαιώ. Εγώ είμαι υπέρμαχο τη ε, ρύθμιση, αναλευτική προσπάθεια και μόνον και θα αποφεύγαμε και όλο το πρόβλημα των απορρίψεων. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αξία και δεν υπάρχει δυνατότητα να ληφθούν αποφάσεις τέτοιε στο Συμβούλιο που ε, φυσικά εξυπηρετούνται άλλα συμφέροντα τα οποία δεν ασφισβητώ, καθένα τη δουλειά του κάνει. Αλλά το θέμα είναι ότι τα προβλήματα αυτά δεν θα πρέπει να σχετίζονται με μέτρα τα οποία θα έπρεπε να είναι πολύ απλά. Επίση, είμαι υπέρμαχο και το είπα, αυτό όντω το είπα, όπως είπε και ο κύριος Παστόρ και νομίζω ότι δεν διαφωνώ σε καμία περίπτωση με αυτό που είπε. Βεβαίως πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Είπα ναι, όμως. Ναι, όμως. Θα πρέπει να γίνει βαθμιδών, υπάρχουν κάποιοι ενδιάμεσοι στόχοι οι οποίοι είναι λογικοί και αυτό στο οποίο είμαι αντίθετος είναι να ε, πούμε Απαραίτητο ότι πρέπει να μειωθεί η ελευθερική προσπάθεια κατά 50% για να γίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι και εγώ το έχω δει. Ε, σε κάποια είδη, ανεξάρτητα από αυτό που μας είπε εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν γίνονται τα πράγματα έτσι. Φτάνουμε σε ακραίε ε, θέσεις και όταν ε, προσπαθούμε στην πράξη να τα εφαρμόσουμε, που είναι εκτό από αυτέ τι αίθουσε, είναι στα λιμάνια, στην κοινωνία που ζούμε, είναι πολύ πιο δύσκολο να τα προσωμιώσουμε όλα αυτά, διότι ουσιαστικά λέμε στον κόσμο ότι θα πρέπει κατά 50% να μειώσει το μισθό του. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να έχουμε μια λογική ισορροπία. Βεβαίω και πρέπει να μειώσουμε την αλληλευτική προσπάθεια. Σε αυτό συμφωνώ. Συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόσχημα για να αδρανίσουμε. Αλλά Υπάρχουν πολλά μέτρα τα οποία θα μπορούσαμε να λάβουμε και θα μπορούσαμε να καθίσουμε ώρες να τα συζητάω εδώ, αλλά δεν θα το σας παταλήσω το χρόνο σας έτσι. Εγώ είμαι υπέρμαχος του να καθορίσουμε σαφείς στόχους για όλα τα αποθέματα προκειμένου να φτάσουμε σε ασφαλή βιολογικά όρια. Διότι όταν θα είναι σαφή τα αποθέματά μας δεν θα έχουμε προβλήματα εξάντληση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, σε καμία περίπτωση δεν το έχω δει, ακόμα και στι πιο ακραίε περιπτώσεις. Όταν ένα απόθεμα θεωρούμε ότι βρίσκεται στην... ε, ε ε, στα ασφαλή βιολογικά όρια μπορεί να μην έχει ε, προβλήματα ανανέωση. Μπορεί να διαπιστώσει προβλήματα ανανέωση για ένα χρόνο, αλλά την επόμενη χρονιά θα ανανεωθεί. Και εκεί θα δούμε που καθορίζουμε και το μέγιστο οικονομικό στοιχείο. Οικονομικό στοιχείο σημαίνει όφελο, αλλά υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Υπάρχει και το στοιχείο τη παραγωγή. Θέλουμε να παράγουμε περισσότερο μεταξύ άλλων. Και τέλο, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πω ότι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ε, όπως ε, τα λέει τα πράγματα ο Ντόν Ερνέστο Πένας, εγώ θα υπέγραφα ό,τι μου δίνουν ε, στα τυφλά. Αλλά δεν είναι έτσι, μας δίνουν τα χαρτιά και στην πράξη οι περισσότερες θέσεις είναι ακραίες. Αυτή είναι η βάση. Ευχαριστώ κύριος Παστόρ. Ευχαριστώ. Έχω πολλές ερωτήσεις ε, που οποίες πρέπει να απαντήσω. Θα επιλέξω κάποιες από αυτές. Το πρώτο ερώτημα της Ιζαμπέλη για το MSY ολόκληρο του οικοσυστήματος ε, νομίζω ε, το έχω ήδη καλύψει, ίσως υπήρξε κάποιο πρόβλημα και δεν με καταλάβατε. Ε, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε περί χαμηλού εισοδήματος, το δέχομαι, αλλά ουσιαστικά σας μιλούσα ε, για ε, τη διαφορά ανάμεσα στην οικονομική και τη βιολογική απόδοση και κατά τη γνώμη μου με χαμηλότερη αλλιευτική προσπάθεια, δηλαδή χαμηλότερη θνησιμότητα, μπορείτε να επιτύχετε υψηλότερη οικονομική απόδοση. Η προτείνουν ότι πρέπει να συνεχίσουν τις αναλύσεις τους ε, οι ειδικοί και πρέπει να μετέχουν στην εκπόνηση των πολιτικών. Συμφωνώ και με τον κύριο Πένας ε, ότι δύσκολα μπορώ να φανταστώ οι επιστήμονες ε, να είναι τόσο κοντά στους πολιτικούς γιατί δεν είναι παραγωγικό η αποστολή του επιστήμονα είναι ανεξάρτητος, να εξακριβώνει όλες τις ε, πληροφορίες. Ε, εάν αποφασίσετε ότι θα διατηρηθεί αυτός ο ρόλος, εντάξει, αλλά πιστεύω ότι ελοχεύει πραγματικά ο κίνδυνος να εμπλακούν ε, υπερβολικά στην εκπόνηση πολιτικής οι επιστήμονες και εγώ θα ήμουν κατά αυτής της τάσης. η κυρία εκεί πίσω μου με ρώτησε μήπως θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ξεκάθαροι ως προς τους ορισμούς. Ε, στη συζήτηση έχει προκύψει αυτό το θέμα αρκετέ φορέ. Ε, θα έπρεπε να είμαστε ξεκάθαροι. Για ποιο MSY μιλούμε ακριβώς, για, ποιο... για ποια μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Συνήθω ε, είναι λίγο ασαφής η χρήση του, του όρου αλλά μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα ε, στην εξέταση του MSY σε σχέση με την εκμετάλλευση, δηλαδή πόσα ψάρια θα ψαρέψουμε σε σχέση με το σύνολο του αποθέματος, ε, ε, διάκριση ανάμεσα σε αυτό και το MSY της βιομάζας. Μπορούμε να ελέγξουμε την, την αλίευση, αλλά αυτό που, τη θνησιμότητα επίσης, αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη βιομάζα μέσα στην θάλασσα. Μεσομακροπρόθεσμα ε, ελπίζουμε να έχουμε τα οικοσυστήματα που θα μας δίνουν τις ε, ε, αποδόσεις που επιθυμούμε. Φυσικά δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Θα έλεγα λοιπόν ότι για αυτό το νομοθέτημα που συντάσσετε τώρα θα έπρεπε τουλάχιστον να είστε ξεκάθαροι για την έννοια την οποία, στην οποία βασίζεστε. Ε, μιλάτε για MSY ως προς την απόδοση ή ως προς ε, την θνησιμότητα των ψαριών. Θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι γι' αυτό. Ε, μιλήσατε για την, ε, το στόχο του 2015 για τη θνησιμότητα και για το στόχο του MSY για τη βιομάζα για το 2020. Το πρώτο στόχο πάνω κάτω νομίζω θα τον καταφέρουμε. Για το δεύτερο θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Αν υπάρξουν αλλαγέ στο οικοσύστημα λόγω των κλιματικών αλλαγών και φύγουν κάποια είδη από μια συγκεκριμένη περιοχή, ε, μπορεί να συνεχίσει κανεί την ελίευση ενό μικρότερου αποθέματο με μια θνησιμότητα η οποία όμω ε, θα συνδέεται με το MSY, αλλά δεν μπορείτε να περιμένετε να επανέλθει ε, στην πρώτερη κατάσταση το απόθεμα, ω προ το μέγεθό του δηλαδή. σε σχέση με την παρέμβαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τα συστήματα διαχείρισης ε, και χρήση της έννοιας του, ε, της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης για την εκπόνηση αυτών των σχεδίων, νομίζω ότι ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση από την εμπειρία μου τα τελευταία δύο χρόνια θα έλεγα ότι θα πρέπει να εμπλακούν σε πολύ μεγάλο βαθμό όλοι οι ενδιαφερόμενοι στη διαδικασία. Όταν συζητά κανείς με τους ενδιαφερόμενους φορείς για τις στρατηγικές, Ξέρετε, θα ε, συνεπάγεται αυτό ότι θα υπάρχει και μεγαλύτερη αφοσίωση από πλευρά του ε, σε σχέση με το να του επιβάλλει κάποιο ε, ένα νέο σύστημα. Ε, σχόλια εκτό μικροφώνου. Θα ακούσουμε μόνο την απάντηση του ομιλητή. Ε, σε σχέση με την ε, συνολική θνησιμότητα. Θα μπορούσε να είναι δυνατό αυτό που μας λέτε, αλλά είναι άσκηση ισορροπίας. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τη δοκιμή στη Βαλτική, όπου ουσιαστικά έχουμε τέσσερα ήδη Εκεί μπορείτε να ε, ε βρείτε ισορροπία ανάμεσα στην εκμετάλλευση των ε, θηρευτών και των θηραμάτων αντίστοιχα Δύσκολα όμως μπορείτε να αντιμετωπίσετε την εθνισμότητα για αυτά τα είδη. Ουσιαστικά αν εκμεταλλευτείτε το σύνολο του οικοσυστήματος ε, με ήπιο τρόπο, με σχετικά χαμηλή θνησιμότητα, ε, αυτό θα είναι υποφελές για το, το οικοσύστημα. Ναι, μεν, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι επειδή ε, στοχεύεται στοχεύετε συγκεκριμένα είδη θα επηρεάσετε και τα συγκεκριμένα αποθέματα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ολοκληρώθηκε το πρώτο πάνελ και να περάσουμε στο δεύτερο πάνελ ομιλητών θα ισχύσει το ίδιο χρονοδιάγραμμα, μισή ώρα το πολύ ε, και κατόπιν 45 λεπτά ε, για τη συζήτηση και έτσι θα τελειώσουμε στην ώρα μας. Το δεύτερο πάνελ λοιπόν έχουμε το θέμα της διαχείρισης του στόλου και έχουμε δύο εκπροσώπους. Ο πρώτος ε, είναι ο κύριος Ολιβιέ Γκιαντεχ από το Ιφρεμέρ και κατόπιν έχουμε τον κύριο Πάμπλο Ροντρίγκε Σαγκούν. Καταρχάς όμως ο κύριος Γκιαντεχ ε, καλωσορίσατε και έχετε το λόγο για μισή ώρα το πολύ. Δεν είναι υποχρεωτικό να την εξαντλήσετε. Merci, Madame la Présidente. Euh, merci de... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε στη σημερινή ακρόαση. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τη διαχείριση του στόλου, καθώς και για τη ρύθμιση της πρόσβασης ε, στα αλλιεύματα. Είμαι οικονομολόγος ε, φυσικών πόρων ε, στη μονάδα ε, θαλάσσιας οικονομικής στο Ινστιτούτο Ήφρεμ στη Γαλλία. Θα ήθελα να κάνω την παρουσίασή μου επί τη βάση πέντε σημείων. Πρώτον, το θέμα της υπερδυναμικότητας του στόλου και οι οικονομικές της αιτίες. Δεύτερον, ανάγκη μηχανισμών αποτελεσματικών μηχανισμών πρόσβαση στα για να ρυθμίσουμε αυτό το θέμα της υπερδυναμικότητας. Ε, τρίτο θέμα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διοικητικών προσεγγίσεων σε σχέση με τις εμπορικές προσεγγίσεις. Ε, προσπαθώ να σας κάνω και μία βιοοικονομική ανάλυση για την μετάβαση στο νέο σύστημα, προς το MSY δηλαδή, τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Και μετά ε, το πέμπτο σημείο είναι τα συμπεράσματά ε, λοιπόν, ω προ την υπερβολική δυναμικότητα του στόλου, για έναν οικονομολόγο πρόκειται για ένα θεμελιώδη ζήτημα. Δηλαδή, όταν θέλουμε να διευρύνουμε το θέμα της διαχείρισης αλίας και να αρχίσουμε να εξετάσουμε τη διαχείριση των θαλασσίων οικοσυστημάτων, οι οικονομολόγοι βλέπουν ότι μια βασική αιτία της υπερεκμετάλλευσης σχετίζεται με την υπερβολική δυναμικότητα ε, του στόλου, του ελευτικού στόλου. Και βλέπετε σε αυτό το, σε αυτό το διάγραμμα τον αριθμό των σκαφών, τη χρήση τους, την ονομαστική τους ισχύ κτλ. Τα νέα σκάφη, ε, τα μεταχειρισμένα σκάφη. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι αυξάνεται ε, η δυναμικότητα. Χρησιμοποιήθηκαν οι επιδοτήσεις από για να επανεπενδύσουν στον τομέα. Αυτό παρατηρείται κυρίως στη Γαλλία, αλλά αληθεύει και σε άλλες χώρες. Λοιπόν, ποιοι είναι οι οικονομικοί μηχανισμοί που διέπουν την υπερβολική δυναμικότητα. Θα ήθελα να κάνω κάποιες σημαντικές και παρατηρήσεις. Πρόκειται για κοινού πόρου. Ε, αυτά τα αλλιεύματα είναι κοινοί πόροι και παρουσιάζουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά πριν την ε, εκμετάλλευση δεν μπορεί κανείς να οικειοποιηθεί τα ψαρέψη, δεν μπορεί να τα εκμεταλλευτεί πριν τα ψαρέψει. Επίσης, ε, διαχείριση των ε, κοινών πόρων είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Στον τομέα της αλίας, τα αλλιεύματα εξαρτώνται από την αλλιευτική προσπάθεια που κάνουν οι υπόλοιποι αλίες. Δηλαδή, όταν αλλιεύει κάποιο, ε, μειώνεται το αποτέλεσμα για όλου του υπόλοιπου. Και τι συμβαίνει, γίνεται ένας αγώνας ε, για τα ψάρια ε, που μεταφράζεται σε υπερβολικές επενδύσεις σε σχέση με την παραγωγικότητα των πόρων και άρα προκύπτει η υπερβολική δυναμικότητα του στόλου. Αυτό ασκεί πολύ σημαντική πίεση στους πόρους. Από οικονομικής ε, πλευράς, ε, ε, παρά τις επενδύσεις υπάρχουν οικονομικές ζημιές λόγω του ανταγωνισμού των αλλιέων και όπως είπα και νωρίτερα ασκείται μεγαλύτερη πίεση στα αποθέματα. Ειδού το βασικό πρόβλημα στον τομέα της αλλίας. Ε, υπάρχει μια πολύ σημαντική χρονική διάσταση του ζητήματος, διότι αυτή η πίεση επί των αποθεμάτων αυξάνεται αναλογικά και με την τεχνολογική πρόοδο. Εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό στην κοινωνία στην οποία ζούμε. Αυξάνεται επίση και η ζήτηση. Ε, η κατανάλωση ε, ψαριών στην Ευρώπη διαρκώ ε, αυξάνεται και στο παρελθόν συνέβαινε και αυτό. Υπάρχουν πολλά κίνητρα. Κρατικέ επιδοτήσει, παραδείγματο χάρη, για να αυξηθούν οι ελευτικέ προσπάθειε. Υπάρχουν διάφορε επιστημονικέ δημοσίευσει και μελέτε που το αποδεικνύουν. Λοιπόν, χρειαζόμαστε θεσμικούς, τους κατάλληλους θεσμικούς μηχανισμούς για να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα. Η οικονομική ανάλυση λοιπόν φέρει επί αυτών των ζητημάτων. Alors, qu'est-ce qui peut être fait la, la, la Commission propose un Τι μπορούμε να κάνουμε. Προτείνει μια σειρά ε, ε, ε, μέτρων που μας ενδιαφέρουν. Πρόκειται για ένα γενές πρόβλημα της αλίας, αλλά ε, δεν ε, είναι ανυπέρβλητο. Μπορούμε να το εξοδετερώσουμε αν εφαρμόσουμε τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης. Λοιπόν, αυτό το θέμα της υπερβολικής ε, δυναμικότητας δεν ρυθμίζεται αποκλειστικά και μόνο με μέτρα διατήρησης των αποθεμάτων. Ακόμη και αν εφαρμόσουμε τις ποσοστώσεις και τα τάκα ή το νέο σύστημα, ε, διαχείριση των προστατευόμενων ε, θαλασσίων ε, βιοτόπων. Αυτό αποδεικνύεται και πάλι από επιστημονικές μελέτες. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε και συμπληρωματικά μέτρα για να ρυθμίσουμε το πρόβλημα. Μέτρα διατήρησης με στόχο την διατήρηση των παραγωγικών και αναπαραγωγικών δυνατοτήτων των αποθεμάτων, που όλο και περισσότερο πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ε, θαλάσσια οικοσυστήματα για να συνεχιστούν τα ε, συνέχιστη Ε, συνεχιστεί η ίδια αλλιευτική προσπάθεια, το ίδιο, τα ίδια, το ίδιο επίπεδο αλλιευμάτων ε, για να μειώσουμε τους ε, αντικτύπους που έχει ο στόλος στο θαλάσσιο περιβάλλον κτλ. Χρειαζόμαστε λοιπόν μέτρα ρύθμισης της πρόσβασης για να δώσουμε μια απάντηση. Αυτό όμως δεν είναι πάντοτε απλώς στην εφαρμογή του, δηλαδή Ανάμεσα στους παραγωγούς θα πρέπει να μοιράσουμε ισότιμα τις αλληλευτικές δυνατότητες. Θα πρέπει να εντοπίσουμε δηλαδή τους αλληλείς που δικαιούνται που έχουν μάλλον άδεια αλληλείας, ε, να ε, χρησιμοποιήσουμε τη συνολική ποσότητα και κατόπιν να κάνουμε την κατανομή και να δούμε πόσο μπορεί να ψαρέψει ο καθένας. Αυτό προϋποθέτει ότι θα έχουμε απαντήσει σε δύο ε, ερωτήσεις. Πρώτον, χρειαζόμαστε τη μεταβλητή του ελέγχου Έχουμε τις αλλιευτικές ε, προσπάθειες και τα αλλιεύματα. Εντάξει, έχουμε αυτές τις δύο συνιστώσεις, αλλά θα πρέπει, όπως είπα, να συνυπολογιστεί ε, και ο παράγοντας έλεγχος. Γιατί προηγουμένως αναφέρθηκα και στα διοικητικά μέτρα κατά κόρον αυτά χρησιμοποιούσαμε μέχρι στιγμής. Ε, πρόκειται λοιπόν για άδειε ή ατομικά μη μεταβιβάσιμα δικαιώματα που μπορεί να σχετίζονται με τα αλλιεύματα ή με την αλλιευτική προσπάθεια. Ε, προκειμένου ε, μιλάμε για τη χορήγηση αλλιευτικών αδειών ή ατομικών ποσοστώσεων. Η ατομικων ποσοστων εναλλακτική είναι να βασιστούμε σε μέτρα που υπακούν στις αρχές της αγοράς. Δηλαδή να θεσπίσουμε συστήματα ε, μεταβιβάσιμων ε, αυτή τη φορά ατομικών ε, αλληλευτικών δικαιωμάτων. Αυτά τα μέτρα, τα διαφορετικά είδη μέτρων έχουν εφαρμοστεί στον κόσμο λάκερο. Και υπάρχουν και πολλά συστήματα, συστήματα ε, συνδιαχείρισης και ξέρετε μπορούμε να μάθουμε από ε, τις εμπειρίες άλλων χωρών για να βρούμε τις ε, πιο πρόσφορες θεσμικές λύσεις. λοιπόν, υπάρχουν πλειονεκτήματα και μειονεκτήματα σε κάθε προσέγγιση. Καμία προσέγγιση ε, δεν ε, είναι εύκολη. Ξέρετε ότι είναι πολυδιάστατο το θέμα της αλληλευτικής προσπάθειας. Ε, δηλαδή, ε, στις διάφορες ε, συνιστώσεις μπορούμε να αντικαταστήσουμε ή μάλλον να το πω αλλιώ, αν ε, προσπαθήσετε να επιβάλλετε μείωση του μήκου του σκάφου, θα το αντικαταστήσει αυτό, θα το αντισταθμίσει ο ψαρά, γιατί θα μεγαλώσει το μέγεθο των ματιών, των δικτυών τα κτλ. Ε, σχετικά τώρα με τον περιορισμό των αλλιευμάτων ε, για τα... και τον έλεγχο των αλλιευμάτων, χρειαζόμαστε ένα μεν αλλά χρειαζόμαστε και αποτελεσματικό έλεγχο, παρακολούθηση, άρα μεγαλύτερο κόστος. Επίσης προσοχή γιατί αυτά τα μέτρα μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση των απορρίψεων. Και αυτό πρέπει να το ε, λάβουμε υπόψη. Ε, οι ποσοστώσεις ε, για τις ε, απορρίψεις αυξάνονται και πάντοτε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος θα πρέπει να προσαρμόζουμε λοιπόν τις αλληλευτικές ε, προσπάθειες ε, στον στόλο. Δηλαδή, όταν κάτι επηρεάζει, ένα συμβάν επηρεάζει τη ζωή μιας επιχείρησης ή όταν ε, το βιολογικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι εταιρείε αλλάζει, δύσκολα η διοικητική ε, αρμόδια αρχή μπορεί να περιορίσει τις ε, αλλιευτικές ε, προσπάθειες ανασκάφος. Ένα άλλο πρόβλημα αυτή της διοικητικής, αμυγός διοικητικής προσέγγισης είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις, και θα επανέλθω σε αυτό στη συνέχεια, διαπιστώνουμε ότι ε, ανεπίσημες αγορές ανταλλαγής δικαιωμάτων εμφανίζονται. Αυτό φυσικά είναι ανησυχητικό. Τώρα, υπάρχει, υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, δηλαδή μέτρα που υπακούν στις αρχές της αγοράς. Μπορεί να προκύψει στρέβλωση διότι είναι ατελής ο ανταγωνισμός ή διότι δεν είναι αρκετά πολύ άριθμε οι αγορέ, ούτω ώστε ο οικονομικό πώς να είναι βιώσιμο αυτό το σύστημα μεταβιβασιμότητας των ατομικών ε, αλληλευτικών ε, δυνατήτων. Από τι εμπειρίε μα σε διάφορε χώρε. χώρες βλέπουμε ότι από κοινωνικο-οικονομική άποψη υπάρχουν πολλά μειονεκτήματα ω προ τη μεταβιβασιμότητα των δικαιωμάτων διότι πρώτον μειώνεται ο αριθμό των θέσεων απασχόληση, το έχουμε δει στην Ισλανδία αλλά όχι μόνο. Δεύτερον, συγκέντρωση των ε, δικαιωμάτων σε ένα πολύ περιορισμένο αριθμό χρηστών. Αυτό που ένας οικονομολόγος μπορεί να σας πει από αυτού εδώ είναι ότι οι αγορές είναι, ε, έχουν θεσμικό ε, χαρακτήρα και άρα μπορούν να ρυθμιστούν για να εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον. Εδώ σε αυτό το ε, πίνακα μπορείτε να δείτε τα διάφορα συστήματα ρύθμισης της πρόσβασης που υπάρχουν στις χώρες του ΟΣΑ, χώρες μέλη του ΟΣΑ, και ε, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται λοιπόν σε αυτό το πίνεκα ότι υπάρχουν ε, κάποιες προσπάθειες ε, ρύθμισης που βασίζονται στις προσπάθειες ή στα ισχύοντα αλλιεύματα. Είναι σίγουρα ενδιαφέρον να προχωρήσουμε, να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτά τα συστήματα αλλά το ιδανικό είναι να αναπτύσσουμε συστήματα που είναι προσαρμοσμένα ε, σε κάθε αλίευμα. Στη Νέα Ζηλανδία, παραδείγματο χάρη, υπάρχει ένα σύστημα πλήρω μεταβιβασιμών δικαιωμάτων. Ε, στη Γαλλία, επειδή ξέρω, γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση, δεν υπάρχει καθόλου ε, στην επίσημη αγορά μεταβιβασιμότητα των δικαιωμάτων, αλλά υπάρχει ένα θέμα ποσοστώσεων και αδειών για πολύ συγκεκριμένα είδη ε, ας επανέλθω τώρα πάλι στη Γαλλία. Αυτό το σύστημα βασίζεται σε ή, ε, είδη που εντοπίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και είδη που έχουν τοπικό ενδιαφέρον και ε, οι οργανώσεις παραγωγών αλλά και οι αλληλευτικές οργανώσεις διαχειρίζονται αυτά τα είδη, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο ε, για την αίσια λειτουργία του συστήματος και το τονίζω διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να ε, τονίζουμε το ρόλο όλων των εμπλεκομένων φορέων, όπως οι αλληλευτικές οργανώσεις, ε, να τονίζουμε πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε μηχανισμό ρύθμισης της πρόσβασης. Στο γαλλικό παράδειγμα βλέπουμε ότι αυτά τα μη μεταβιβάσιμα δικαιώματα απαγορεύεται η μεταβίβαση των αλληλευτικών δικαιωμάτων στη Γαλλία. Έγινε λοιπόν μια οικονομετρική μελέτη και απεδείχθη ότι ανεπίσημα σε μια δευτερογενή αγορά ε, ανταλλάσσονται αυτά τα δικαιώματα ταυτόχρονα με τα σκάφη. Γιατί συνδέονται τα δικαιώματα με τα σκάφη. Ε, και το 2003 ε, η... είδαμε ε, ότι το 2, 3, τα δύο τρίτα της αξίας των δικαιωμάτων ανταλλάσσονταν σε αυτήν την δευτερογενή αγορά. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι αν δεν είναι ικανοποιητικά τα μέτρα ε, προκύπτουν αυτόματα ανεπίσημες αγορές ανταλλαγής των αναλυτικών δικαιωμάτων. Ε, πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο που μου φαίνεται ενδιαφέρον σε σχέση με την ανάπτυξη των συστημάτων συνδιαχείρισης Στο περιοδικό Nature δημοσιεύθηκε αυτό το άρθρο. Λοιπόν, έλεγε εκεί ότι οι μηχανισμοί ρύθμιση τη πρόσβαση είναι πάρα πολύ σημαντικοί για τη διαχείριση των αλλιευμάτων, αλλά η ηγεσία, η συνδιαχείριση, η αυτορύθμιση είναι επίση ε, σημαντικοί παράγοντε για την ε, επιτυχή διαχείριση ε, των αλλιευμάτων. Χρειαζόμαστε λοιπόν μηχανισμούς ρύθμισης της πρόσβασης αλλά και θεσμικά ε, πλαίσια που ε, θα εξασφαλίσουν την συμμετοχή των αλλιών που μπορούν να φανούν ε, καινοτόμοι. Et par rapport à ce qui a euh, Λοιπόν, τώρα σε σχέση με την ανάλυση του συστήματος, της μετάβασης μάλλον προς το σύστημα MSY, συμμετείχα σε, μία, σε ένα κίνημα όπου εκπροσωπήθηκαν ε, συμβουλευτικά συμβούλια, επαγγελματίες ε, για να γίνει μια ε, βιοοικονομική ανάλυση στον κόλπο της Γασκόνης για την μετάβαση στο σύστημα MSY για συγκεκριμένα είδη επειδή τα γνωρίζουμε καλά και αναπτύξαμε ένα βιοοικονομικό μοντέλο προσωμείωση ουσιαστικά της δυναμικής των πληθυσμών των ψαριών αλλά και της εκμετάλλευσης αυτών από διάφορα είδη καθώς και τι οικονομικές επιδόσει ε, αυτών των στολίσκων. Ε, το παρουσιάσαμε στην μόνιμη επιστημονική επιτροπή το, για τη διαχείριση των αλλιευμάτων αυτό το πόρισμα και βλέπετε εδώ πέρα στο πρώτο διάγραμμα την αύξηση της ε, βιομάζας που συνδέεται με ε, πάγιο τάκ 400.000 τόνων σε σχέση με ένα μεταβαλλόμενο τάκ. Ε, στην πρώτη περίπτωση ε, παραμένουν, ε, στην, δεν αυξάνονται τα αλλιεύματα. Ε, όπως είπε και ο κύριος ε, Παστόρε, ε, εάν υιοθετηθεί το MSY μπορεί να αυξηθεί η οικονομική επίδοση των στολίσκων και τα κέρδη για τους αλληλείς. και όπως λέγαμε και στην αρχή της ε, παρουσίασής μου, ε, το κέρδος ενός ε, σημαίνει ζημιά για όλους τους υπόλοιπους. Άρα χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό ρύθμισης κατάλληλο για κάθε συγκεκριμένο αλίευμα. Θα κλείσω κάνοντας κάποιες παρατηρήσεις από οικονομικής πλευράς το θέμα της διαχείρισης υπερβολικής δυναμικότητας του στόλου ε, είναι μείζον θέμα. Μία από τις λύσεις ε, θα είναι η εξατομίκευση ε, των αλλιευτικών δικαιωμάτων. Αυτό μπορεί να βασιστεί σε έλεγχο των αλλιευμάτων εφόσον εν γέννη ελέγχουμε τις ε, αλλιευτικές προσπάθειες, ε, ε, άρα μπορεί αυτό να συνηγορεί υπέρ των ατομικών ποσοστών. Όπως σας είπα και νωρίτερα, για να σημειώσουμε επιτυχία χρειαζόμαστε τα προσφορότερα συστήματα σε σχέση με κάθε είδος αλλιεύματος. Η ρύθμιση της ε, πρόσβασης ε, δεν είναι ένα στοιχείο που επαρκεί από μόνο του. Άλλες ε, συνιστώσεις απαραίτητες είναι ένα καινοτόμο σύστημα συνδιαχείρισης για να σημειωθεί επιτυχία διότι για να έχουμε, σημειώσουμε επιτυχία στον έλεγχο θα πρέπει να συμμετάσχουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. πρόκειται Λοιπόν, για ευαίσθητα ζητήματα και συνήθως δημιουργούνται και παρανοήσεις ε, όταν μιλάμε για διατήρηση. Όταν, αν εξατομικευτούν τα δικαιώματα, προσδιορίζονται και αποκτούν μια συγκεκριμένη εμπορική αξία ε, και ε, γίνονται αυτεπάγγελτα, αν θέλετε, μεταβιβάσιμα αυτά τα δικαιώματα. Ο ρόλος των αρχών είναι η ρύθμιση της μεταβασιμότητας των δικαιωμάτων για να είμαστε αποτελεσματικοί και για να είναι δίκαιο ε, το σύστημα. Και για πολλά αλλιεύματα <clears throat> υπάρχουν ήδη ε, τέτοια συστήματα σε άλλες χώρες του κόσμου. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι η ρύθμιση της πρόσβασης στα ε, πρέπει να γίνει αμελητή, να βρούμε ε, καινοτόμες ε, οικοσυστημικές ε, μεθόδους συνδιαχείρισης, αλλιώς θα έχουμε πολύ χαμηλές επιδόσεις στον τομέα της αλίας Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Γκουγιάντερ, και τώρα... τα θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και για το δυναμικό της αλίας και για το μοντέλο διαχείρισης. Και τώρα επόμενος εμπιλητής είναι ο κύριος Παύλο Ροντρίγκε Σαργκούν, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση παραγωγών κατεψυγμένου τόνου. Να σας ζητήσω. Να σας δώσουμε λοιπόν το λόγο, κύριε Ροντρίγκε Σαούν. Bueno, muchas gracias. Eh... Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω την πρόεδρο τη Επιτροπή Αλληλείας, την Κάρμεν Φράγα, διότι μου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσω εδώ στην συνεδρίαση της Επιτροπής Αλληλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ευχαριστήσω και τους Ευρωβουλευτές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, όλους όσους ε, συμμετέχουν σε αυτή τη ε, συνεδρίαση. Δεν θα είναι και τόσο επιστημονική παρουσίασή μου ε, θα είναι λίγο μία εικόνα της ε, εικόνας του τομέα του κατεψυγμένου τόνου. Να σας πω καταρχάς ότι η οργάνωσή μας περιλαμβάνει 20 σκάφη ε, κατεψυγμένου τόνου ε, από την χώρα των Βάσκων. Πρόκειται για σκάφη τα οποία είναι κατασκευασμένα στην πλειονότητα του στη χώρα των Βάσκων και ε, επειδή πρόκειται για βιομηχανική αλληλεία, παρόλα αυτά να σας πω ότι έχει μια πολύ οικογενειακή δομή, σχεδόν παραδοσιακή. Ε, φέτος συμπληρώνει τα 50 χρόνια μίας εκ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνουμε. Είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο, διότι δείχνει ότι δεν είμαστε άρτια φιχθέντες σε αυτή την αλληλεία. Έχει 50 χρόνια περίπου που ασχολούμαστε με τον κλάδο και θα θέλαμε να συνεχίσουμε άλλα 50 χρόνια να δραστηριοποιούμαστε στον ίδιο κλάδο. Μισό λεπτό να βρω πώς πάει η διαφάνεια. Καταρχάς λοιπόν να σας δώσω κάποια προκαταρκτικά στοιχεία για το τι ακριβώς αλλιεύουμε. Αλλιεύουμε τροπικό τόνο. Ο τροπικός τόνος περιλαμβάνεται μεταξύ των φινοειδών ε, είναι ένα τμήμα του και σε γενικές γραμμές ο κατανολητής ε, και το ευρύ κοινό θεωρεί ότι ένας τόνος υπάρχει, αλλά στην πράξη έχουμε πολύ διαφορετικά είδη μεταξύ τους ε, με πολύ διαφορετικά οικονομικά, βιολογικά στοιχεία και δεν έχει καμία σχέση για παράδειγμα η αλία του ερυθρού τόνου με την αλία του τροπικού τόνου που αλλιεύουμε εμείς με τα ε, σκάφη μας. Εδώ βλέπετε λίγο πολύ τα ετήσια αλλιεύματα. Έχουμε τα στοιχεία για το 2008 των θηνοειδών. Από τα 4 εκατομμύρια τόνους που αλλιεύθηκαν, η αλλιεία του τροπικού τόνου, ε, που είναι ουσιαστικά ο χιτρινόπτερος και, και η παλαμίδα, είναι περίπου στο 1,5 ε, εκατομμύριο τόνους. Η κατάσταση του τροπικού τόνου, όπως σας έλεγα προηγουμένως, ε, δεν έχει καμία σχέση με άλλη μορφή αλίας στην όπως για παράδειγμα του ερυθρού τόνου. Έχουμε πολύ γρήγορους ρυθμούς αναπαραγωγής, ε, μικρά και μεσαία μεγέθη, που σημαίνει ότι έχουν και μικρό ε, προσδόκιμο ζωής και στην περίπτωση των ειδών αυτών, ουσιαστικά δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση δυνατότητα υπερεκμετάλλευσης στην ε, μεγάλη ε, πλειονότητα των περιπτώσεων είμαστε μέχρι τα τρία χρόνια κύκλο ζωής και σε καμία περίπτωση δεν έχουμε υπεραλίευση. Ε, πρόκειται για ένα απόθεμα το οποίο έχει κάποια χαρακτηριστικά που το διακρίνουν από οποιαδήποτε πρόβλημα υπερεκμετάλλευσης. Να σας πω επίσης ότι ο Ευρωπαϊκός Στόλος Τινοειδών είναι τελείως διαφορετικό ε, το μοντέλο. Ε, πρόκειται για σκάφη τα οποία είναι εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν μέτρα τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία μεταφέρονται απευθεία ε, ε, στην νομοθεσία και επομένω όλα αυτά τα σκάφη πρέπει να πληρούν όλους τους κανόνες και επιπλέον πρέπει να πληρούνται και οι κανόνες που απαιτούν και οι χώρες τις οποίες αλλιεύουμε. Ε, για παράδειγμα, τα σκάφη μας θα πρέπει σε πολλές περιπτώσεις να διαθέτουν ε, διπλά δορυφαρικά συστήματα ελέγχου, διότι από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται η συγκεκριμένη διάταξη, ενώ για παράδειγμα στι Σεϊχέλε, για να λιεύσει κάποιο τα ύδατα των Σεϊχελών, πρέπει να υπάρχει μια διάταξη δορυφορικού ελέγχου που ε, καθορίζεται από την νομοθεσία των Σεϊχελών. Για την αλληλεία λοιπόν αυτή να σας πω ότι ε, στην αλία του κυτρινόπτερου τόνου δεν γίνεται απαραίτητα μεταφορά και εκφόρτωση στο λιμένα, σε αντίθεση με την αλία της παλαϊμίδας που είναι υποχρεωτική εκφόρτωση και επομένως η εκφόρτωση σημαίνει ότι θα υπάρχει έλεγχος και συγκεκριμένη ε, ανιχνεσιμότητα, αρκετά σημαντική. Εδώ έχουμε κάποια στοιχεία για τον αριθμό των ευρωπαϊκών ε, σκαφών ε, γρηγρή που αλλιεύουν στα ε, ύδατα αυτά. Έχουμε 24 θυναλιευτικά που αποτελούν το 15% του παγκόσμιου στόλου σε σύνολο. 24 στον Ατλαντικό, 26 στον Ινδικό και 4 στον Ειρηνικό, 54 στο σύνολό τους. Και ουσιαστικά πρόκειται για σκάφη τα οποία αλλιεύουν στα ασιατικά και λατινοαμερικανικά ύδατα. Και εδώ έχετε και τα στοιχεία που αλλιεύουμε εμείς ε, σε, σχέση, σε σύγκριση με το παγκόσμιο ε, αλλιεύμα. Εδώ βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε κατά βάση αλληλεία στον Ατλαντικό και στον Ινδικό ωκεανό. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και αλληλεία στον Ειρηνικό ωκεανό, αλλά είναι μικρή. Και εδώ πρέπει να πω ότι υπάρχουν και τα θέματα των αλλιευτικών ε, συμφωνιών σύμπραξης και στην περίπτωση του Ατλαντικού ωκεανού, όπως βλέπετε και στο διάγραμμα, υπήρχε μια πολύ σημαντική μείωση τα τελευταία χρόνια στον αριθμό των ε, συμφωνιών που διαπραγματεύτηκαν και αυτό για το στόλο μας που ε, περιορίζεται στους ωκεανούς αυτούς είναι σημαντικό το πρόβλημα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο ε, αντιμετωπίζει ο στόλος μας στον Ειδικό ωκεανό είναι η πειρατεία. Τα θηναλιευτικά είναι αρκετά ευάλωτα για δύο λόγους. Πρώτον, διότι για λόγους αλληλείας θα πρέπει να βρίσκονται σε ανοιχτή θάλασσα για μεγάλο χρονικό διάστημα και επίσης είναι πολύ χαμηλό το κήτος του σκάφους και επομένως είναι πάρα πολύ ευάλωτα και αυτό είναι ε, ε κάτι το οποίο διαπιστώσαμε από το 2005 και μετά όταν είχαμε τις πρώτες πειρατικές επιθέσεις των Σομαλών στον Ινδικό ωκεανό. Στο 2008 είχαμε ε, την πρώτη ε, επιδρομή σε ένα σκάφος του οργανισμού μας. Το 2009 είχαμε τη δεύτερη και αυτό υποχρέωσε τους ε, πλειοκτήτες να λάβουν συγκεκριτικά μέτρα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει και κάποια μονάδα ασφαλείας επί του σκάφους για να μπορεί κάποιος να αλλιεύει στα ύδατα του Ινδικού ωκεανού και παρά το γεγονός αυτό είχαμε αρκετές επιθέσεις ε, και καταλήψεις. Ε, πέρσι είχαμε, συγγνώμη, τον προηγούμενο μήνα είχαμε ένα πολύ σημαντικό κύμα το οποίο δεν οδήγησε σε κατάληψη του σκάφους αλλά ε, καθημερινά υπάρχουν απειλές, υπάρχουν πληροφορίες για ομάδες πειρατών οι οποίες εξακολουθούν να διαστηροποιούνται στη θάλασσα. Είναι αλήθεια ότι οι διεθνείς δυνάμεις ασφαλείας ε, δραστηριοποιούνται επίσης. Ε, σήμερα το πρωί άκουσα τον επικεφαλής της επιχείρησης Αταλάντα ε, να, να λέει ότι ε, λείπουν πάρα πολλές ε, μονάδες και βρίσκονται περίπου στα όρια και έκανε έκκληση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να γνωρίζουν ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται και θα πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο να αντιμετωπιστεί. Τα σκάφη έχουν βέβαια και ιδιωτική ε, μονάδα ασφαλεία συνήθως, αλλά παρόλα αυτά ε, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι σημαντική η παρουσία στον Ινδικό ωκεανό και θα πρέπει να επιληθεί το βασικό πρόβλημα που είναι ότι υπάρχουν διαρθρωτικές ελλείψεις ε, στη Σομαλία, αλλά γι' αυτό δεν μπορεί να λυθεί μία νυχτή και επομένως θα πρέπει στην θάλασσα να υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Υπάρχουν και επιπτώσεις που αντιμετωπίζει ο στόλος μας ε, λόγω του προβλήματος της πειρατείας. Υπήρξαν κάποια σκάφη που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον Ινδικό ωκεανό. Υπάρχουν επιπτώσεις ε, διότι κάποια σκάφη πρέπει να ε, συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται και να έχουν ασφάλεια επί του σκάφους. Επομένως υπάρχουν πολύ σημαντικά ε, διοικητικά κόστη, υπάρχει πολύ σημαντική επιβάρυνση και πρέπει ο καθένας να αναλαμβάνει ε, μόνος του τα έξοδα της ε, ιδιωτικής ασφάλειας για να μπορεί να παραμείνει στα ανοιχτά της θάλασσας και επίσης είναι και το γεγονός ότι πρέπει να εργάζονται υπ' αυτά στα συνθήκα στον ειδικό κενό. και επομένως επειδή μου δίνεται εδώ η δυνατότητα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αν δεν υπήρχε η πλήρη συνεργασία των πληρωμάτων μας ε, στα σκάφη, μάλλον οι επιχειρήσεις μας θα είχαν ε, βαγίσει προπολού. Ε, όπως σας είπα, αλλιεύουμε σε διεθνή ύδατα, στην Αφρική κυρίως, και χάρη στην παρουσία μας ε, εκεί, ε, έχουν ανθίσει αρκετές, ε, αρκετά σημαντικές επιχειρήσεις μεταπίεσης. Το γνωρίζει άλλωστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόσφατος υπήρχε αποστολή του Κοινοβουλίου στις Ιχέλες και είδατε ε, η διεισόμαση της οικονομικές συνέπειες ε, τις θετικές οικονομικές συνέπειες ε, στην περιοχή, διότι υπάρχουν επιχειρήσεις μεταποίησης και δίνονται δυνατότητες και για εξαγωγές χάρη στη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Στόλου. Όσον αφορά τη διαχείριση των δυνατοτήτων μας, ε, να πω ότι υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές από τη ΦΑΟ που λένε ότι θα πρέπει να γίνεται έλεγχος ε, και σωστή διαχείριση, αλλά επισημαίνεται επίσης ότι υπάρχουν και κάποια είδη τα οποία ε, είναι αντικείμενο υπεραλίευσης. Για τον τροπικό τόνο νομίζω ότι πόρο απέχουμε από την υπεραλίευση και καθημερινά προσπαθούμε να έχουμε μέτρα τα οποία χρησιμοποιούνται για άλλα ε, είδη στόλων και άλλα είδη αλλιευμάτων. Στον Ατλαντικό, ο Ευρωπαϊκό στόλος είναι πολύ πιο κάτω από τα ποσοστά αναφοράς που καθορίζει η ICAT και νομίζω ότι ε, υπήρξε και σημαντική μείωση ευρωπαϊκών σκαφών στον Ατλαντικό ωκεανό. Ε, και είχαμε πολύ σημαντική βελτίωση του αποθέματος στην περιοχή. Στον Ινδικό ωκεανό και λόγω της πειρατείας και λόγω του γεγονότος ότι αρκετά σκάφη αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την αλία στον Ινδικό ωκεανό, το τμήμα του στόλου που είναι ε, στην περιοχή είναι πολύ κάτω από τα επίπεδα που καθορίζει η Περιφερειακή Οργάνωση Αλίας του Ινδικού Ωκεανού. Ε, τα ποσοστά τα οποία καθορίζονται για τον ευρωπαϊκό στόλο είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά που επιτυγχάνονται. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε υπεραλίευση παράκτιου στόλου ούτε στον Ινδικό ούτε στον ε, Ατλαντικό Ωκεανό. Όπως σας έλεγα, αυτό που θέλουμε είναι να διασκεδάσουμε λίγο τις αμφιβολίες. Ξεκινάμε από την προϋπόθεση της υπερεκμετάλλευσης, κάτι το οποίο είναι πολύ σύνηθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για υπεραλίευση ε, ειδών, ε, ενώ δεν ισχύει για όλα τα είδη και θέλουμε να έχουμε μείωση και μείωση του στόλου. Εμείς δεν ε, εντασσόμαστε στην όλη συζήτηση και θεωρούμε ότι είναι λανθασμένο το γεγονός ότι ε, στόλοι όπως το δικό μας, που είναι ευρωπαϊκός <coughs> στόλος ε, που έχει συγκεκριμένη παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο, ε, προσπαθούν να μας πείσουν ότι πρέπει να μειώσουμε το στόλο μας και να σταματήσει η αλίευση. Δεν νομίζω ότι μας αφορά αυτή η συζήτηση. Πρόκειται για μια συζήτηση η οποία περιλαμβάνει και το τομέα μας, ενώ κανονικά ότι δεν θα έπρεπε και αν συνεχιστεί θα αναγκαστούν τελικώς ε, οι πλειοκτήτες μας να ε, αλλιεύουν με σημαίες ε, χωρών που είναι πολύ λιγότερο απαιτητικέ. Και φυσικά εδώ βλέπετε και μία σύγκριση με τον υπόλοιπο στόλο που έχουμε που αλλιεύει ε, οι περισσότεροι αλλιεύουν στην Ασία και εδώ στα πλαίσια αυτά μπορείτε να δείτε τι διαφορά υπάρχει ως προς το κόστος για το γεγονός ότι ένα ευρωπαϊκό σκάφος ε, είναι γεγραμμένο στα ευρωπαϊκά μητρώα και πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις και απαιτήσει. Δεν αναφέρομαι στην αλία και μόνο, υπάρχει και επίπεδο υγείας, ε, υγιεινής συνθήκες και βλέπετε ότι το κόστος διαχείρισης Ενό ισπανικού σκάφου για παράδειγμα σε σχέση με τις υπόλοιπες τριστήλες όπου έχουμε σκάφη σημαία Ταϊβάν ή ε, ε, σημερινού και ούτω καθεξής είναι πολύ διαφορετικό. Πρόκειται λοιπόν για ένα θέμα το οποίο είναι υπαρκτό και έχει και σχέση με τη συνέχεια και το μέλλον αυτού του στόλου. Βιωσιμότητα τώρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία και νομίζω ότι συμφωνεί και η επιστημονική κοινότητα. Ο τροπικός τόνος είναι ένα απόθεμα το οποίο βρίσκεται σε πολύ ευνοικέ συνθήκε σε σχέση με τα υπόλοιπα αλλιευτικά είδη. Ε, σε όρου ICAT ε, υπήρχαν κάποιες εκστρατείε ε, σε κάποιες οργανώσεις που προσπαθούν λίγο να στιγματίσουν τον στόλο που ε, ψαρε, αλλιεύει και τα παραλιεύματα που αλλιεύονται. Είναι πάρα πολύ χαμηλά τα ποσοστά παρελευμάτων που έχουμε εμείς ε, στην αλία που κάνουμε και ο το ο μέας μας πολλές φορές ε, ξεχωρίζει γιατί είναι πολύ δραστήριος και προσπαθεί ε, να μετριάσει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η αλληλεία, όπως όλες τις δραστηριότητες στο θαλάσσιο περιβάλλον. Έχουμε μια σειρά από δραστηριότητες. Επαναλαμβάνω ότι τα προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται είτε μέσω ευρωπαϊκής ε, ενίσχυσης ε, από το GAP ε, ε, και από αντίστοιχα προγράμματα, προγράμματα για να μετριάσουμε τις επιπτώσεις από τις αλλιευτικές δραστηριότητες και ε, όπως σας είπα, αν τα δούμε όλα αυτά στο παγκόσμιο πλαίσιο της συγκεκριμένη αλλίας, ε, αν δείτε ότι αν υπάρχει ένας τομέας ο οποίος διακρίνεται επειδή ακριβώς είναι τόσο δραστήριος είναι ο ευρωπαϊκός τομέας. Ολοκληρώνοντας να σας πω ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ενιαίο μοντέλο για τη διαχείριση όλων των αλλιευτικών ειδών. Η κατάσταση των τροπικών θηνοειδών είναι αρκετά ευνοϊκή. Ε, εργαζόμαστε σε ένα ε, πλαίσιο διάφανο από πλευράς ρυθμιστικής. Ε, υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο πάρα πολύ ισχυρό και αυτό μεταφράζεται, όπως σας είπα, σε υψηλό κόστος εκμετάλλευσης και το κόστος αυτό είναι για τα σκάφη μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χρειάζεται πρώτη ύλη. Υπάρχει ένας μεταποιητικός τομέας που χρειάζεται να λάβει πρώτη ύλη από το στόλο μας και ε, ταυτόχρονα ε, τα σκάφη αυτά είναι ένας τομέας πάρα πολύ σημαντικός και επειδή ακριβώς ο τομέας των θηνοειδών είχε πολύ σημαντική συμμετοχή για την υγεία του τομέα, ενός τομέα ο οποίος είναι πολύ καλά πλαισιωμένο στην περιοχή μας, στη χώρα των Βάσκων, αλλά και σε άλλες περιοχές, στη Γαλλικία, σε περιοχές οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αλία αυτή. Η σύστασή μας λοιπόν είναι αν θέλουμε να υπάρχει βιωσιμότητα, που είναι και ο στόχος μας, θα πρέπει να ε, ευνοηθούν η στόλοι μας όπως ε, για παράδειγμα ο Ευρωπαϊκός Παράκτιος Στόλος που έχει ε, όλα τα μέσα και εφαρμόζει όλους τα μέτρα σωστά. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να επιτευχθούν νέες συμφωνίες και εγώ επιτρέψτε μου να σας πω ότι θα πρέπει να παραμείνουν και οι παρούσες συμφωνίες. Όλοι γνωρίζουμε ότι λόγω της μεταρρύθμισης που γίνεται αυτή τη στιγμή στην κοινή αλληλευτική πολιτική με κριτήρια και νέε απαιτήσει μπορεί και να ε, ελοχεύει κίνδυνος για όλες αυτές τις συμφωνίες και να γίνει αυτό που συνέβη στις προηγούμενες, στην προηγούμενη μεταρρύθμιση, συγγνώμη, που είχαμε σημαντική μίεση των αλληλευτικών συμφωνιών. Θα έχουμε ανανέωση σε μεγαλύτερο αριθμό των ε, αλληλευτικών συμφωνιών θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας, θα πρέπει να παραμείνει αυτό το δίκτυο διαχείρισης ε, των συμφωνιών αλληλείας και θεωρούμε ότι βοηθά τον τομέα να επικεντρωθεί στα ύδατα των ε, παράκτιων ε, περιοχών και για μας υπάρχουν και κάποιες δυσκολίες για οικονομικούς αλλά και για λόγους διαφάνειας. Τέλος, και ολοκληρώνω, Δεδομένου ότι μιλάμε για αλληλεία σε διεθνή ύδατα την οποία διαχειρίζονται οι περιφερειακές οργανώσεις αλληλείας θα πρέπει να γίνει διαχείριση από τις περιφερειακές οργανώσεις αλληλείας και επομένως ε, να λαμβάνονται μονομερώς εσωτερικά μέτρα για τα ευρωπαϊκά σκάφη τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη το διεθνές πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιούμε θα μας φαίνεται ε, ότι μας επιβαρύνει και θα ήθελα να επισημάνω ότι η πολιτική βιωσιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι συνεπής και να ε, συνάδει και με την εμπορική πολιτική. Ε, θέματα για παράδειγμα της ε, γεωγραφικής ένδειξης για τις χώρες όπως είναι η Παππούα, η Γουινέα και άλλες θα είναι καταστρεπτικά και θα δημιουργήσουν προβλήματα όχι μόνο στον ευρωπαϊκό τομέα αλλά και σε όλες τις χώρες ε, της Αφρικής των οποίων η βιωσιμότητα θεμελιώνεται στην παρούσα κατάσταση. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να είναι ανταγωνιστική ε, και παραγωγική σε άλλους τομείς εάν ε, αρχίσει να καταφθάνει αλίευμα μεταποιημένο από την Παππούα Νέα Γιουνέα με ασιατικά προϊόντα, που είναι ο φόβος που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο ε, θα στραφεί εναντίον μας, αλλά θα στραφεί και εναντίον των χωρών της ε, Αφρικής, οι οποίες ε, μπορούν να είναι βιώσιμες μόνο εάν διατηρηθεί η κατάσταση ως έχει. Υπάρχουν πολλές θέσεις απασχόλησης οι οποίες κινδυνεύουν να χαθούν ε, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Αφρική ε, λόγω ε, των μέτρων αυτών να είμαστε αυστηροί ως προς τη βιώσιμότητα, αλλά να προσέξουμε και τους εμπορικές πτυχές. Ε, ορισμένες φορές σκοφεύουμε και μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε χωρίς να τηρούνται υγειονομικοί κανόνες, χωρίς να τηρούνται κοινωνικοί κανόνες και νομίζω ότι αυτές οι διαφορετικές θέσεις που έχουμε ε, σε επιχειρησιακό επίπεδο και βλέπουμε για παράδειγμα ένα ευρωπαϊκό σκάφος ε, που φροντίζει να τηρεί όλους τους κανόνες και να δίνεται κατάλληλη αποζημίωση στο πλήρωμα και να υπάρχουν ανθρώπινες ε, συνθήκες ε, εργασίας και ε, διευκολύνονται τα ελάχιστα πρότυπα και από την άλλη διευκολύνουμε και ασιατικές χώρες να ενταχθούν ε, στα ύδατά μας και νομίζω ότι όλα αυτά είναι επιβλαβή και θα πρέπει να σας επιστήρω την προσοχή και σε αυτό το πρόβλημα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ροντρίγες Σαγκούν, διότι μας παρουσιάσετε τα προβλήματα του στόλου που αλλιεύει εκτός ευρωπαϊκών υδάτων, θυναλιευτικού στόλου σε αυτή την περίπτωση, η κυρία Ρόντουστ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις και ελπίζω να μου απαντηθούν πρώτες μου ερωτήσεις αφορούν τον κύριο Ολιβιέ Γκουαντέρ από τη Γαλλία, ο οποίος αναφέρθηκε στη, στο υπερδυναμικό όσον αφορά τα σκάφη. Αυτό το δυναμικό έχει μειωθεί, όμως ο στόλος έχει αυξηθεί. Ε, πρέπει να το εξετάσουμε αυτό ε, με προσοχή, διότι μακροπρόθεσμα μπορεί αυτό να οδηγήσει σε κοινωνικά προβλήματα. Το ερώτημα μου είναι, έχετε αναλύσει τι σημαίνει αυτό το γεγονός ε, και τι, πώς θα εξηγήσουμε στους αλληλείς ότι έχουμε υπερδυναμικό σε ορισμένους τομείς ε, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα από κοινωνικής πλευράς. Τι προτάσεις έχετε. Εν συνεχεία, στον τελευταίο μιλητή ε, δεν Σημείωσα το όνομά του, είναι ο κύριος Ροντρίγκε Σαγκούν. Αυτό το οποίο δεν μπορώ εγώ να εξηγήσω ως απλή πολίτης, βλέπω τεράστια σκάφη ε, τα οποία κυκλοφορούν και από την άλλη πλευρά βλέπω πειρατικά σκάφη ε, τα οποία δεν μπορούν να συλληφθούν από τις, τα ραντάρ και από το GPS. Ε, δεν μπορούν να ανοιχνευθούν. Πώς δικαιολογείται αυτό. Αναφέρατε ότι για την ανείχνευση και την καταπολέμηση της πειρατείας έχετε προσλάβει ε, ε, προσωπικό ασφαλείας ε, και θέλω να ξέρω πόσο κοστίζει όλη αυτή η εκστρατεία, όλη αυτή η η ασφάλεια την οποία χρειάζεστε. Όλη η διεθνή κοινότητα είναι ενωμένη στην καταπολέμηση της πειρατεία αυτού του φαινομένου. Σε αυτό συμφωνώ. Αλλά τι προτάσεις έχετε για μας στην Επιτροπή Αλία, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Επίσης όσον αφορά τις ε, περικοπέ στην ε, στο διοικητικό κόστος, τι προτείνεται και σε αυτό το τομέα. Ε, έχουμε ακούσει πολλές φορές ε, ότι ε, πολλοί αρμόδιοι κάθονται στους ε, πύργους τους απομονωμένοι και δεν έχουν άμεση σχέση με, τη, με τους αλείς, με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην αλία. Πώς θέλετε εσείς να προωθήσετε τη βιώσιμη αλία. Ρωτώ, ο δικός σας ο στόλος, τα δικά σας σκάφη αλλιεύουν βιώσιμα θα σημειώσατε ότι Α, είπετε ότι με τη νέα αλλιευτική πολιτική θα πρέπει να συνάψουμε περισσότερες συμφωνίες και να ε, ε, περιλαμβάνουν το στοιχείο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύτιμο, αξιόλογο και πρέπει να περιληφθεί και είπατε ότι στη δική σας αλία, στο δικό σας τύπο αλίας δεν έχετε υπερδυναμικό. Δεν έχετε πλεονάζον δυναμικό. Σημαίνει αυτή η σας παρατήρηση ότι θέλετε να αυξήσετε το στόλο σας. Να αυξήσετε το δυναμικό. Αυτά προς το παρόν. Η κυρία... Η κυρία Μπαρέα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε θα τους πάρω ανάποδα τους ομιλητές. Ε, να πω στον ε, τελευταίο ομιλητή ότι εγώ είμαι υπέρ των διεθνών ε, συμφωνιών αλίας για διάφορους λόγους, γιατί θεωρώ ότι η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοηθά να βελτιώνεται η κατάσταση σε χώρες που δεν σέβονται τη βιωσιμότητα. Η βιώσιμη αλληλεία σε περιοχές στις οποίες υπάρχει έλλειψη πόρων δεν θα εφαρμόζεται και επίσης ε, ε, για τα θέματα ασφαλείας εμείς θα θέλαμε να συνεχίσει η επιχείρηση Αταλάντα ε, παρά το γεγονός ότι ακούσαμε εδώ ότι μάλλον δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι και ε, εμείς θα το κυνηγήσουμε αυτό το θέμα. Για τον πρώτο μιλητή θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. αναφερθήκατε σε ένα θέμα το οποίο φαίνεται να είναι ταμπού και αναφέρεται λίγο το θέμα της αλλιευτικής προσπάθειας. Η αλλιευτική προσπάθεια είναι ουσιαστικά οι μέρες στη θάλασσα. Και μας είπατε ότι υπάρχει δυνατότητα να επιληθεί το πρόβλημα και μας είπατε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε το σύστημα διαχείρισης της ελευτικής προσπάθειας ε, σε συνδυασμό με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση και μας είπατε ότι υπάρχει και σχετική πείρα και ήταν θετική η πείρα αυτή. Ε, υπάρχουν κάποια θέματα βέβαια τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως τμήμα της λύσης ε, της κοινή ελευθερικής πολιτικής. Ε, επίσης είπατε ότι ε, στη Γαλλία είναι απαγορευμένο, αλλά είπατε ότι υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή σε άλλες χώρες και ότι υπάρχει μεταφορά ε, των σκαφών. Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα. Η κυρία ευχαριστώ και τους άλλους ομιλητές. Ε, ευχαριστώ τους δύο ομιλητές. Θα ήθελα να ρωτήσω τον τελευταίο ομιλητή για τον κατεψυγμένο τόνο. Μιλήσατε για την ε, κατανομή των ελευτικών δικαιωμάτων και ότι βλέπετε ότι χάνετε τα δικαιώματά σας, τα παραδοσιακά, ιστορικά, αλληλευτικά σας δικαιώματα ε, έναντι από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα χάνετε δηλαδή προς όφελος εκείνων. Τώρα παραδοσιακά αλλιευτικά δικαιώματα των πλουσίων χωρών δεν μπορούν να ισχύσουν εσαΐ, ε, διότι υπάρχουν και άλλα μέρη του κόσμου, άλλες χώρες αναπτυσσόμενες, υποανάπτυξη, οι οποίες έχουν και αυτές το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην ε, ε, παγκόσμια αλλιευτική προσπάθεια. Πρέπει λοιπόν να γίνει σεβαστό το αμοιβαίο αυτό δικαίωμα ε, και η πλούσια πλευρά του κόσμου, η πλούσια, η ευημερεύουσα πλευρά πρέπει να λάβει υπόψη τα δικαιώματα και των άλλων. Αυτό είναι περισσότερο μια δήλωση που είχα να κάνω και όχι τόσο ερώτημα, αλλά έχω και μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Ε, στην ανακοίνωση για την εξωτερική πολιτική... Ε, στα πλαίσια της κοινή αλλιευτικής πολιτικής αναφέρονται οι αλλιευτικές ε, παραχωρήσεις που πρέπει να είναι υποχρεωτικές. Όμως εξαιρείται τα σκάφη τα οποία δίνεται να αλλιεύουν ή υπό τις διατάξεις των διμερών συμφωνιών, διμερών αλλιευτικών συμφωνιών. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, πώς, ε, γιατί το κάνατε αυτό, γιατί κάνατε αυτή την εξαίρεση και τι επίπτωση θα έχει αυτή η εξαίρεση. Και πάλι αναφέρ, αποτείνουμε στον κλάδο και ρωτώ. Τι επιθυμείτε εσείς, ε, θέλετε να έχετε ένα σύστημα ITQ στα RFNOs και ε, στον πρώτο μιλητή, τον κύριο Γκαντιέ, ε, θα ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τη διαχείριση της ελευτικής προσπάθειας. Θέλετε να μειώσετε την προσπάθεια. Υπάρχουν μερικά καλά θετικά παραδείγματα στον κόσμο όπου η διαχείριση, τα διαχειριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν στην ελευτική προσπάθεια αποδείχθηκαν επιτυχή. Υπάρχει άλλος που επιθυμεί να ε, παρέμβει, παρακαλώ. Ε, κύριε Πουλπάου Μπαραντίκα, να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές και να πω το εξής. Όσον αφορά τα μεταβιβάσιμα δικαιώματα, να πω στον πρώτο μου μιλητή ότι είχαμε διάφορες εμπειρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διαφορετικά αποτελέσματα και αυτή η δυνατότητα μεταβίβασης των δικαιωμάτων θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μονοπόλια. Θα μπορούσε να δημιουργήσει και συγκέντρωση δικαιωμάτων εις βάρος ε, άλλων μορφών αλίας ή θεωρείτε ότι από άποψη οικονομικής ε, βιωσιμότητας θα μπορούσε να είναι εφικτό σε συνδυασμό και με όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Και να πω επίσης στον κύριο Ροντρίγκε Σαγκούν όσον αφορά την επιχείρηση Αταλάντα αναφερθήκατε και σε ένα από τα σκάφη στα οποία υπήρξε επίθεση, να πω ότι η επιχείρηση Αταλάντα δεν δημιουργήθηκε για να προστατεύει τα λιευτικά σκάφη. Εδώ στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου έγινε μια συζήτηση και εγκρίθηκε και ένα σχετικό ψήφισμα και στο ψήφισμα καταλήξαμε σε συμφωνία πολλές ε, δυσκολίες και συμπεριλάβαμε και τα πιο ευάλωτα σκάφη, τα οποία είναι τα πιο ευαίσθητα ε, στο θέμα της επιχείρησης Αταλάντα. Η επιχείρηση Αταλάντα λοιπόν δεν δημιουργήθηκε για να παράσχει αυτή τη μορφή στην προστασία και παρόλα αυτά καταφέραμε να τα συμπεριλάβουμε στο ψήφισμά μας. Μας δώσατε στοιχεία. Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο στο Κοινοβούλιο να δώσουμε την εικόνα που μας δώσατε εσείς σήμερα και να μιλήσουμε για τον κλάδο ε, των, ε, καταψυκτικό, ε, των θυναλιευτικών καταψυκτών και να πούμε ότι είναι σκάφη τα οποία τηρούν την ομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι είναι πολύ αυστηροί, ότι δεν παραβιάζουν την ομοθεσία, ότι σέβονται τα ύδατα στα οποία αλλιεύουν και μπορούν να οδηγήσουν και σε οικονομική ανάπτυξη. Ελπίζω από σήμερα να αλλάξει η εικόνα που υπάρχει για τα σκάφη αυτά και να ε, συμμερίζονται όλοι την εικόνα που μας δώσατε και οι ευρωβουλευτές και ελπίζω να μπορέσουν να έχουν επιχειρήματα και στοιχεία για να δείξουν ότι υπάρχει και μια πραγματικότητα που διαφέρει ε, από αυτήν που μας πλασάρουν κάθε φορά. Συμφωνώ απολύτω και το έχουμε πει επανειλημμένως ότι πρέπει να γίνεται μια πολιτική που θα είναι πιο συνεκτική μεταξύ των ε, αλληλευτικών δικαιωμάτων και των εμπορικών συμφωνιών. Ακόμα και εδώ στην Επιτροπή Αλληλεία ε, έχουμε διστάμενε απόψει ε, στις αλληλευτικέ συμφωνίες, διότι φαίνεται ότι οι αλληλευτικέ συμφωνίες τείνουν να να είναι ε, παράπλευρα ζητήματα τα οποία δεν συζητούν στις εμπορικές συμφωνίες. Ελπίζουμε λοιπόν να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που να συνεχίσουν να ε, προχωρούν το θέμα των συμφωνιών με τρίτες χώρες που δεν είναι υποφελής μόνο για μας αλλά και για τρίτες χώρες που αναγκάζονται να τηρήσουν τα ευρωπαϊκά κριτήρια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μια-δυο ερωτήσεις. Καταρχάς, για αυτά που είπε ο κύριο ε, Ροντρίγκε Σαγκούν, παρά το γεγονό ότι ξεφεύγουμε λίγο από το σημερινό θέμα, αλλά επειδή είστε εδώ, θα ήθελα να πω αυτό που είπε η Επίτροπος ε, της Προάλλης στο Συμβούλιο Υπουργών, ως προς τη δυνατότητα ο κοινοτικό στόλο ε, να πληρώνει δικαιώματα αλληλείας ε, απλώς και μόνο επειδή αλλιεύει ε, στην, ε, σε συγκεκριμένες περιοχές περιφερειακών οργανώσεων αλληλείας. Όταν τη ρώτησαν αν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει το θέμα αυτό δεν απάντησε σαφώς αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Θα ήθελα να ξέρω την άποψή σας επ' αυτού. Για τα όσα είπατε επίσης, θα ήθελα να θέσω και μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι ο κύριος Ροντρίγκης Αγιούν είπε τουλάχιστον αυτό αντιλήφθηκα εγώ, ότι η διαχείριση των δυνατοτήτων θα πρέπει να είναι διαφορετικά ε, για τα σκάφη που αλλιεύουν αποκλειστικά εκτός των ε, κοινοτικών υδάτων, διότι εκεί υπάρχουν και οι εντολές για και τις συστάσεις για την ε, υπεραλίευση, που είναι διαφορετικές από αυτές που έχουμε για τα σκάφη που αλλιεύουν εντός των ευρωπαϊκών υδάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να το εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο. όσον αφορά τα όσα ακούσαμε από τον πρώτο μιλητή, αν κατάλαβα καλά, εσείς είστε υπέρ της ε, μεταβίβασης ατομικών δικαιωμάτων αλίας, ε, παρά το γεγονός ότι στο τέλος μας είπε ότι θα μπορούσαν να προκύψουν και προβλήματα. Νομίζω όμως, και αυτό έχει σημασία, ε, ότι η αρχή των μεταβιβάσιμων ατομικών δικαιωμάτων είναι ένα μοντέλο το οποίο είχε και σωστή λειτουργία και ακόμα και πιο συντηρητικές χώρες όπως για παράδειγμα η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, ο Καναδάς και οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ε, εφήρμοσαν αυτή τη μορφή στα συστήματα και προφανώς θα μπορούσαν να υπάρξουν και κάποιες αρνητικές συνέπειες και αυτό είναι που προσπαθούμε να μετριάσουμε. Ε, η αρχή είναι χρήσιμη, αυτό έχει σημασία να το αναφέρουμε και αποδείχθηκε ότι ήταν το πιο αποτελεσματικό μέτρο για τη μείωση των δυνατοτήτων και να υπάρχει και μεγαλύτερη οικονομική απόδοση και ότι τα αρνητικά στοιχεία όπως για παράδειγμα ε, η συγκέντρωση, εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι τόσο μεγάλη η συγκέντρωση του αλληλευτικού τομέα διότι δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το συγκεντρωτισμό ο τομέα αλλά Εάν αυτά φοβάται ο τομέα μπορεί να υπάρχουν και ρήτρε διασφάλιση, είτε σε περιφερειακό επίπεδο είτε σε όποιο επίπεδο θέλετε. Η αρχή θεωρούμε ότι είναι καλή και είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε οποιαδήποτε ρήτρα διασφάλισης που θα μπορούσε ε, να καθησυχάσει όσους φοβούνται φαινόμενα συγκεντρωτισμού ή τη μείωση των θέσεων εργασίας. Η μείωση των θέσεων εργασίας η οποία θα μπορούσε να υπάρξει σε πρώτο στάδιο θα μπορούσε να τη δει κάποιο και από την αντίθετη πλευρά. Εάν ε, δεν ε, χρησιμοποιηθεί το σύστημα αυτό στο μέλλον, θα μπορεί να υποδεινωθεί ο τομέα τη αλίας και να χαθούν ακόμα περισσότερε θέσει στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτέ τι πτυχέ. Να δώσω λοιπόν καταρχά τον νόμο λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατόπιν να δώσω το λόγο στους ομιλητέ. Έχουμε τρία τέταρτα στη διάθεσή μας αν μετά από όλες αυτές τις απαντήσεις ε, θέλει κάποιος άλλος να κάνει κάποια επιπλέον ερώτηση, εγώ θα σας το επιτρέψω. Καταρχάς να δώσω το λόγο λοιπόν στους ομιλητές, ο κύριος Πένας ε, καταρχάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να αναφερθώ στην παρέμβαση του κυρίου Γκιατέχ και να τον ευχαριστήσω για την παρουσίασή του γιατί εγώ δεν έχω και τίποτα να προσθέσω από αυτά που είπε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμμεριζόμαστε σε μεγάλο βαθμό, αν όχι και όλη την ανάλυση που σάνατε. Συγχαρητήρια λοιπόν, διότι έχουμε απόλυτη σύμπτωση απόψε. Να θίξω όμως ένα από τα θέματα τα οποία ανέφερε στα συμπεράσματά του ο κύριος Γκουγιαντέρ για να ε, σταθώ και σε ένα θέμα που ανέφεραν πολλοί από τους ομιλητές σήμερα είπατε ότι η μεταβίβαση ατομικών δικαιωμάτων αλληλεία θα μπορούσε να είναι ρυθμισμένη. Αυτό είναι και το κλειδί της υπόθεσης. Αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα σύστημα μεταβίβασης δικαιωμάτων που δεν σαν αγοραπολισία ε, τύπου χρηματιστηρίου που δεν ρυθμίζεται σε καμία περίπτωση. Κάθε άλλο. Εμείς προτείνουμε ένα σύστημα μία αγοραπολισία δικαιωμάτων αλληλείας ρυθμισμένη και επιμένω σε αυτό θα το πω χιλιάδες φορές αν χρειαστεί. Πρέπει να υπάρχει ρύθμιση διότι υπάρχουν ε, πάμπολες φωνές και εντός κοινοβουλίου και εκτός κοινοβουλίου που είναι αντίθετες στην ιδέα του συστήματος μεταβίβασης ατομικών δικαιωμάτων αλληλείας και αναφέρονται σε δυνητικά προβλήματα τα οποία ε, ίσως είναι και βέβαια. Ο κίνδυνος, για παράδειγμα, υπερβολικής συγκέντρωση σε, ε, λίγα ε, ε, χέρια, σε ολιγοπόλιο. Υπάρχουν και συγκεκριμένοι τομείς του στόλου που μπορεί να διαπιστώσουν ότι θα αγοράσουν όλα τα δικαιώματα λία τους, οικονομικά συμφέροντα πολύ πιο ισχυρά και θα υπάρχει μία απώλεια δικαιωμάτων ε, αλληλείας σε κάποιες περιοχές. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ε, θεωρούμε ότι αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να τύχουν ε, ρύθμισης. Ο συγκεντρωτισμός δεν μπορούμε να πούμε απαραίτητα ότι είναι κακός. Ένα κάποιο επίπεδο συγκεντρωτισμό είναι απαραίτητο ε, και πρέπει να το λάβουμε υπόψη ως μέσο για την αντιμετώπιση της υπεραλίευσης. Αυτό που θέλουμε είναι η υπερβολική συγκέντρωση δικαιωμάτων σε λίγα χώρια να μην υπάρχει γιατί θα ήταν ανεπιθύμητη. Αλλά αυτό μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Σε πολλές χώρες του κόσμου που υπάρχει το σύστημα μεταβίβασης δικαιωμάτων υπάρχουν διάφορα συστήματα τα οποία περιορίζουν ακριβώς τη συγκέντρωση των δικαιωμάτων στους λίγους είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ρυθμίσουμε και εάν τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι είναι απαραίτητο και σε εθνικό επίπεδο, μπορούν κάλλιστα να το ρυθμίσουν και σε εθνικό επίπεδο. Ένα ακόμα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι πρέπει να καθοριστεί ένα σύστημα στο οποίο είτε θα απαγορεύεται είτε θα, θα χρησιμοποιείται ως ανασταλτικός παράγοντας ένα στοιχείο το οποίο δεν θα επιτρέπει στους πλειοκτήτες να... Ε, ε, πατάξουν ουσιαστικά εντό εισαγωγικών την ε, μικρή κλίμακα αλία. Ε, αυτό γίνεται γιατί δίνεται στη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αποκλίνονται αυτά τα δικαιώματα λία σε σκάφη μικρότερα των 2 μέτρων. Πρόκειται για λίγα σκάφη, αλλά σε πολλά κράτη-μέλη ε, η πλειονότητα του στόλου αποτελείται από μικρά σκάφη. Είναι σημαντικό λοιπόν το μερίδιο που θα αποκλειστεί. Υπάρχουν όμως και άλλες εναλλακτικέ εκδοχές. Το μοντέλο της Δανίας για παράδειγμα. Στη Δανία ένας πλειοκτήτης με μεγάλα σκάφη μπορεί να αγοράσει ε, δικαιώματα πλειοκτήτη με μικρά σκάφη, αλλά σε αυτή την περίπτωση του επιβάλλεται και μία ποινή. Και αν ε, ε, ο πλειοκτήτης μικρών σκαφών είχε 100 δικαιώματα, ο πλειοκτήτης μεγάλων σκαφών δεν παίρνει 100, παίρνει λιγότερα ακριβώς γιατί έχει μεγαλύτερα σκάφη. Αυτό που προσπαθώ να σας αποδείξω είναι ότι μπορούν να υπάρχουν μέτρα που μπορούν να μετριάσουν τις αρνητικές συνέπειες. Αυτό λοιπόν που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να καθορίσει ένα σύστημα ε, και να υπάρχει ένα σύστημα αγοράς το οποίο όμως θα είναι ρυθμισμένο. Και εμείς στην πρότασή μας προσπαθούμε να έχουμε κάποια ελάχιστα πρότυπα τα οποία θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα και από εκεί και πέρα να υπάρχει μεγάλο περιφοδόριο ευελιξία στα κράτη-μέλη για να μπορούν να καθορίσουν ε, δικλείδες ασφαλείας ανάλογα με την κάθε χώρα οι οποίες εξ όσων αντιλαμβανόμαστε μπορεί να έχουν και διαφορετικές πραγματικότητες να αντιμετωπίσουν. Τώρα για την παρέμβαση του κυρίου Ροντρίγκε ε, Σαγούν να κάνω δύο διευκρινήσεις. Καταρχάς ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την τάση να μιλάει για υπεραλίευση σε όλους τους πόρους είπατε. Όχι, εμείς λέμε ότι υπάρχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό, πάρα πολύ υψηλό, απαράδεκτα υψηλό υπερεκμετάλλευση πόρων από πλευρά. Ε, του Ευρωπαϊκού Στόλου, αλλά δεν τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσιβούλ, τσουβάλι. Αν υπάρχει κάτι το οποίο λειτουργεί σωστά, το λέμε. Και αν πρέπει να λεφθούν μέτρα για ένα συγκεκριμένο απόθεμα, όλα αυτά βασίζονται στις καλύτερες ε, επιστημονικές πληροφορίες που διαθέτουμε. Εάν ο τροπικός τόμος, τόνος, και το γνωρίζουμε, δεν αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή προβλήματα εκμετάλλευσης, η πολιτική μα προσαρμόζεται σε αυτό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, χρησιμοποιεί ε, όλα τα αποθέματα και όλα τα ε, θέματα αλίευσης και να τα εξετάσεις στο ίδιο πλαίσιο. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να την κατηγορήσετε αν θέλει να μειώσει, ότι θέλει να μειώσει το στόλο μέχρι το 2002. Ε, που υπήρχαν τα πολιετή προγράμματα μείωσης του στόλου. Από το 2002 και μετά δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μείωσης του στόλου και τώρα με το σύστημα ποσοστώσεων και μεταβιβάσεων δικαιωμάτων που προτείνουμε, προσέξτε, προτείνουμε για τους τομείς του στόλου που υπόκεινται σε συστήματα μεταβίβασης δικαιωμάτων, δεν θα πρέπει να υπάρχει πολιτική περιορισμό του στόλου. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα στοιχεία τώρα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει τον αριθμό των σκαφών υποχρεωτικά. Το αντίθετο, ε, η όλη πολιτική των μεταβιβάσεων, ε, της μεταβιβάσεως δικαιωμάτων Ε, θεωρείται ότι καλύτερο να αξιολογείται από τον κλάδο. Δηλαδή ο κλάδος να καθορίσει ποια είναι η καλύτερη δυνατότητα αλίευσης για την εκμετάλλευση των, μετα... των δικαιωμάτων αλίευσης που διαθέτει. Και η πολιτική αυτή απομακρύνεται από την ε, ε, θέση των Βρυξελών να μειώσει το στόλο. Δηλαδή εμείς δεν θα σας πούμε ποιος είναι ο στόλος σας, απλώς σας λέμε ότι πρέπει να διατηρήσετε κάποια βιώσιμα δικαιώματα λίας και εσείς θα καθορίσετε ποια είναι τα ιδανικά για να αλλιεύσετε, επιμένω με βιώσιμο και αποδοτικό τρόπο. Επίσης, ε, τα όσα έθεσε ο κύριος Ροντρίγκε Αγούν για τις νέες συμφωνίες, σας διαβεβαιώ ότι και εμείς θα θέλαμε να συνεχίσουμε με την πολιτική συμφωνιών με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των συμφωνιών για τα ε, θηνοειδή. Οι ανησυχίες βέβαια του τομέα είναι ότι κάποιες από τις ιδέες που θέλει να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως για παράδειγμα να βελτιώσει τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για να μπορούμε να αξιολογήσουμε πολύ καλύτερα από ό,τι σήμερα ε, ποιες είναι οι συνέπειες ε, της αλληλείας από τις τρίτες χώρες. Ή επίσης ε, το σκεπτικό βάσει του οποίου οι πλειοκτήτες θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στα θέματα των δικαιωμάτων αλληλείας, η επισης το σκεπτικο βαση του οποιου οι πλειοκτητες θα πρεπει να συμμετεχουν περισσοτερο στα θεματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά θεωρούνται επιπρόσθετες δυσκολίες για την σύναψη συμφωνιών. Όμως πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει το θέμα αυτό να το δούμε από ένα πρίσμα στρατηγικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι συμφωνίες με τρίτες χώρες σε αρκετά διεθνή <coughs> χώρα ε, έτυχαν ε, επικρίσεων για πολλούς λόγους. Πολλές φορές λένε ότι τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκμεταρεύονται τα αποθέματα των αναπτυσσόμενων ε, μικρών χωρών και τους επικρίνει κάποιος γι' αυτό. Στο Μπόε υπάρχει ένα πολύ σαφές σκεπτικό που λέει ότι τα δημόσια κονδύλια για να διασφαλίσουμε πρόσβαση των ε, ευρωπαϊκών σκαφών ε, στα ύδατα τρίτων χωρών είναι μια μορφή ενίσχυσης προς τις χώρες αυτές. Οι συμφωνίες αυτές λοιπόν μακροπρόθεσμα ε, απαιτούν και την εξέβριση λύσεων σε αυτά τα προβλήματα, σε αυτές τις επικρίσεις. Το να πούμε ότι οι πλειοκτήτες θα πληρώνουν πρόσβαση είναι και ένας εξαιρετικός τρόπος για να απαντήσουμε στους ισχυρισμούς του ΠΟΕ ότι οι συμφωνίες είναι <coughs> ενίσχυση. Εάν καθορίσουμε μια σαφή διάκριση μεταξύ της βοήθειας προς την τρίτη χώρα για την ανάπτυξή της και ε, καταβολή ενός τιμήματος για την άδεια, ε, είναι σαφές ότι ε, ε, εάν την άδεια την πληρώνει ο πλειοκτήτης δεν μπορεί να θεωρείται ενίσχυση. Και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για να προστατεύσουμε και το όλο σκεπτικό των συμφωνιών αλληλείας από τις επικρίσεις ε, νομικού ή πολιτικού χαρακτήρα που έρχονται από όλες τις πλευρές. το ίδιο φυσικά ισχύει και για την επίκριση που γίνεται παραδοσιακά στις, ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πηγαίνουμε και αλλιεύουμε στις αναπτυσσόμενες χώρες και αν θέλουμε πραγματικά να σταματήσουμε να είμαστε αντικείμενο επίθεσης θα πρέπει να βελτιώσουμε τις επιστημονικές μας γνωμοδοτήσεις και να είμαστε βέβαιοι ότι αυτά που αλλιεύουμε εμείς αυτές τις χώρες είναι πράγματι αυτό που οι παράκτιες χώρες δεν θέλουν να αλλιεύσουν. Και πραγματικά ε, ε, αλλιεύουμε τα πλεονάσματά τους. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ε, διασφαλίσουμε αυτές τις συμφωνίες. Τώρα για το θέμα της ε, Παππούας Νέας δεν είμαι εγώ πλέον αρμόδιος, αλλά γνωρίζουμε τι δυσκολίες μπορεί να δημιουργηθούν και ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συνεχίσει αυτή την πολιτική και να δει τι αποτελέσματα θα έχει, ε, προκειμένου να δει και κατά πόσον θα επανεξετάσει το ζήτημα. Δεν μπορώ να σας το πω σήμερα αυτό κυρία Πρόεδρε, αλλά είμαστε εν γνώση του θέματος και θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε. Η κυρία Ρόντου έθεσε μια ερώτηση που δεν ήταν για μένα, αλλά επιτρέψτε μου να απαντήσω εγώ. Τι γίνεται με τα κοινωνικά προβλήματα που ε, σχετίζονται με την υπεραλίευση. Εάν πούμε εμείς ότι, κοιτάξτε να δείτε, στο τάδε είδος υπάρχει υπεραλίευση. Ποια είναι η κοινωνική λύση. Καταρχάς, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το εξή. Πολύ σημαντικό. Ο τρόπος αντιμετώπισης της υπεραλίευσης αυτή τη στιγμή είναι ε, επιδοτήσεις για τις απορρίψεις. Ε, οι ενισχύσεις για τις απορρίψεις δεν είναι κοινωνικό μέσο. Τα χρήματα πηγαίνουν στον πλειοκτήτη. Αυτό το οποίο υπερασπίζονται λοιπόν οι πολλοί δεν είναι κοινωνικό μέτρο και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Ένα το κρατούμενο αυτό. Από εκεί και πέρα αυτό που θέλουμε είναι να συνδυάσουμε την πολιτική της αγοράς δικαιωμάτων αλληλείας με μια πολιτική δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, συμπληρωματικών θέσεων και ε, ενισχυτικών προς τις ε, παράκτες περιοχές. Αυτό θα το εξηγήσουμε πιο αναλυτικά όταν θα παρουσιάσουμε τον κανονισμό για το μελλοντικό διαρθρωτικό ταμείο και εκεί θα δείτε ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και το είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, δεν θα προτείνει ενίσχυση για τις απορρίψεις, αλλά θα υπάρξει ενίσχυση για τη δημιουργία συμπληρωματικής οικονομικής δραστηριότητας ή εναλλακτικής οικονομικής δραστηριότητας στις παράκτιες αλληλευτικές περιοχές. Αυτή λοιπόν είναι η εναλλακτικη οικονομικης δραστηριοτητας απάντηση που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να προσπαθήσω τώρα να απαντήσω και στην ερώτηση της κυρίας Λεβίν για το κατά πόσον ε, το θέμα των ε, δικαιωμάτων μεταβίβασης εφαρμόζεται σε διεθνή ε, αλλιεύματα τα οποία διαχειρίζεται οι περιφερειακές οργανώσεις και όχι τρίτες χώρες. Όταν τα σκάφη μας ε, προσεγγίζουν τα τρίτη χώρας, πρέπει να τηρήσουμε την νομοθεσία των τρίτων αυτών χωρών. Επομένως, μπορούν να αλλιεύσουν μόνο μετά από άδεια από αυτές τις τρίτες χώρες. Μπορούμε να καθορίσουμε ένα σύστημα ανταλλαγή ποσοστώσεων. Αλλά αν ανταλλάσσουμε ποσοστώσει και το παράκτιο κράτο διαφωνεί και δεν μα δίνει άδεια για την αλλιεύση είναι άχρηστε οι ανταλλαγέ ποσοστώσεων. Γιατί να έχουμε λοιπόν ένα σύστημα όταν εξαρτόμεθα από τις άδειε από τρίτη χώρα. Μάλλον δεν είναι το πλέον κατάλληλο μέσο. Γι' αυτό ακριβώ και δεν προτάθηκε κάτι τέτοιο. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να πω το εξή Θα εφαρμοστούν τα δικαιώματα μεταβίβασης ε, σε ε, σκάφη τα οποία λεύουν εκτός ε, υδάτων Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Σε κάποιε περιπτώσεις, όπω για παράδειγμα στην περίπτωση του τροπικού τόνου, δεν υπάρχουν περιορισμοί. Δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου τίποτα να μεταβιβάσουμε, διότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στις ποσοστώσεις. Επομένως, επειδή ακριβώ δεν υπάρχουν περιορισμοί στις ποσοστώσεις, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το σύστημα γιατί τι θα μεταβιβάσουμε. Υπάρχει ε, μια γενικότερη ε, δυνατότητα μεταβίβασης, αλλά δεν υπάρχει κάτι να καθορίσουμε. Αν όμως υπάρχει, για παράδειγμα, περιφερειακή οργάνωση αλλίας όπως η ΝΑΦΟ, για, που υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης δικαιωμάτων, γιατί να μην ε, προτείνουμε εκεί μεταβίβαση δικαιωμάτων. Γι' αυτό προτείνουμε κάποια πράγματα στα πλαίσια συγκεκριμένων οργανώσεων, θα πρέπει να υπάρχει δικαίωμα. Στα τροπικά είδη τόνου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή περιορισμός ε, στα περισσότερα είδη. Και η τελευταία ερώτηση που σημείωσα είναι η ερώτηση της κυρίας Φράγα για το κατά πόσον θα έχουμε ένα συγκεκριμένο καθεστώς στόλου για τρίτες χώρες. Δεν το εξετάζουμε αυτό ενδεχόμενο, γιατί αυτό που εξετάζουμε είναι για όλους τους τομείς στους οποίους ε, εφαρμόζεται το σύστημα μεταβίβασης δικαιωμάτων να υπάρχει μια απελευθέρωση της πολιτικής στόλου, δηλαδή να μην υπάρχει περιορισμός για τον στόλο. Αυτό είναι το σκεπτικό μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ένα σχόλιο μόνο. Την ενίσχυση για τις απορρίψεις τις λαμβάνει ο πλειοκτήτης, αλλά υπάρχουν και κοινωνικά ε, δικαιώματα, κοινωνικές ενισχύσεις, αν δεν κάνω λάθος. Το πλήρωμα, για παράδειγμα, που σχετίζεται με τις απορρίψεις δεν είναι μόνο για τον πλειοπτήτη, αλλά μπορεί να δίνονται και κάποια ε, επιπλέον για κοινωνικούς λόγους, εκτός και ανάλεξη νομοθεσία. Η βασική, όχι. Συνοδευτικά μέτρα, ναι. Ναι, ναι, κοινωνικά συνοδευτικά μέτρα τα οποία σχετίζονται με τι απορρίψει. Αλλά κανεί δεν μας ε, απαγορεύει να έχουμε αυτά τα συνοδευτικά κοινωνικά μέτρα είτε σχετίζονται με την ενίσχυση απόρριψη, είτε σχετίζονται με την αγορά ε, μεταβάσιμων δικαιωμάτων. Είναι ε, ανεξάρτητα. Λοιπόν, ο κύριος Γκουγιαντέρ. Παρακαλώ. Ε, Σας ευχαριστώ για το θέμα της που σχολιάζεται μόλις τώρα, όντως είναι σημαντικό το διακύβευμα. Αληθεύει ότι μειώνονται οι θέσεις απασχόλησης ε, στον κλάδο ε, την τελευταία 20 ετία λόγω κυρίως της αντικατάστασης ε, της εργασίας από το κεφάλαιο. Η προοπτική μεταρρύθμισης και επαναπροσανατολισμό της αλίας προς το MSY έχει ως στόχο να αναπαραγάγει προστιθέμενη αξία στον κλάδο αυτό. Αυτή η προστιθέμενη αξία θα μπορούσε να κατανεμηθεί ανάμεσα στην, ε, ε, στο κέρδος για το κομμάτι κεφάλαιο και το κέρδος για τους εργαζόμενους. Επίσης μπορούμε να έχουμε ε, αλληλεία λιγότερο εντατική ως προς το κεφάλαιο και άρα θα είναι υπέρ της απασχόλησης. Το θέμα είναι βέβαια πώς θα μεταβούμε στο νέο σύστημα. Δεν είναι εύκολο και χρειάζονται σίγουρα συνοδευτικά μέτρα οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα χρειάζεται ίσης ευρηματικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μπορούσαμε ε, να ε, βελτιώσουμε την επιλεξιμότητα των ε, μέσων, των αλληλευτικών μέσων ή δάνεια προς τους αλληλείς, διότι γνωρίζουν με κάποιες ζημιές, αλλά θα αντισταθμιστεί αυτό με μελλοντικά κέρδη ίσως. Βεβαίω ε, θα χρειαστεί οι τράπεζε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να χορηγήσουν αυτά τα δάνεια. Και ελπίζω ότι οι οικονομικέ συνθήκε θα επιτρέψουν ε, την αποπληρωμή των δανείων. Πανάκια δεν συνιστά ε, είναι αυτή η λύση. Τώρα, σε σχέση με την διαχείριση από πλευρά των αλληλευτικών ταμείων, αυτό που είπατε, δεν σημαίνει ότι αυτόματα θα εφαρμόσουμε τη λύση όπως την περιγράψατε. Υπάρχουν ε, ακραίες ε, περιπτώσεις ε, όπως αλληλεία ορισμένων ειδών ε, κοντά στη ΣΥΠΑ ε, με κάποια ε, ορθότερη διαχείριση τελικά καταλήξαμε σε 15 ημέρες αλίας το χρόνο για ορισμένα είδη. Είναι ακραίο αυτό και καταψήξαν ουσιαστικά τις αλληλευτικές προσπάθειες. Υπήρχε υπερβολική συγκέντρωση της προσφοράς. Και το 94-95 δεν θυμάμαι, άρχισε να εφαρμόζεται ένα σύστημα μεταβάσιμων ε, δικαιωμάτων και εκεί ε, προσαρμόστηκαν και αλληλευτικέ ε, προσπάθειε και υπήρξε πιο ισότιμη κατανομή σε ολόκληρο το χρόνο. Έτσι μπορούσαν οι επαγγελματίες να εκμεταλλευτούν καλύτερα την παραγωγή τους για τα νοπά ψάρια. Δεν υπάρχει καμία θαυματουργή λύση, καμία πανάκια. Θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις λύσεις μας, όπως σας έλεγα, σε κάθε αλίευμα. Ε, με μακροπρόθεσμα σχέδια διαχείρισης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ροντρίγες Ναι. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω λίγο τις ε, ερωτήσεις που μου θέσατε. Καταρχάς κάποιος είπε ότι εάν από τεχνολογική σκοπιάς ε, δεν είναι ε, δυνατόν να βρούμε τους πειρατές, ε, τι πρέπει να γίνει. Το πιο απλό παράδειγμα είναι ο, σταλό, ο στόλος μας, ο οποίος από τεχνική σκοπιά είναι πολύ καλά εξοπλισμένος. Έχουμε δύο καταλήψεις σκαφών. Δεν είναι πάντα δυνατό λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε. Πολλές επιθέσεις ε, γίνονται σε σκάφη ε, σε ύψη κάτω από τα 5 μέτρα, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα ανοιχνεύσουν οι συσκευέ επί του σκάφου. Επίσης, ε, θα πρέπει ένα ε, σκάφος να έχει τα δίχτυα του στο νερό και αν υπάρξουν πληροφορίες ότι μπορεί να πλησιάζει ένα πειρατικό σκάφος και είναι ύποπτο, δεν είναι τόσο απλό να σηκώσει τα δίχτυα και να φύγει. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να καθυστερήσει και να πάρει και ώρες. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ ευαίσθητο σκάφος. Ε, αναφερόμαστε σε σκάφη τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένου υλικού και πολλές φορές ε, είναι πολύ εύκολο να τα ανοιχνεύσουν ε, τα σκάφη που δεν μπορούμε να ανοιχνεύσουμε εμείς με τις συσκευέ που έχουμε επί του σκάφους. Αυτό που ζητάμε είναι να συνεχίσει ενισχύ η επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνεχίσει την προσπάθεια και δεν το κάνουμε εμείς χρειάζονται περισσότερες μονάδες στη θάλασσα διότι έχουν χαλαρώσει λίγο τα πράγματα ε, προσφάτως και θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη παρουσίαση, παρουσία σκαφών ε, προστασία στον Ινδικό ωκεανό. Πρόκειται για μια τεράστια έκταση που τρία-τέσσερα σκάφη δεν επαρκούν. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμό και περισσότερε πληροφορίε που τη ζητούμε πάντα από πλευρά Ευρώπη. Στην επιχείρηση Αταλάντα θα πρέπει να γνωρίζουμε πού βρίσκονται συνήθως τα πολεμικά σκάφη για να μπορέμε να διαθέτουμε και εμείς πληροφορίες και κατά κάποιο τρόπο να καθησυχάζονται. Αλλά πάντα δεν μας έδιναν πληροφορίες από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν δεν ήταν για την καλή συνεργασία με την Ισπανική κυβέρνηση για το θέμα αυτό, θα ήμασταν μάλλον αρκετά παροπλισμένοι. Όσον αφορά τη διατήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμεί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αν υπάρχει ένα στόλο που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι ο ευρωπαϊκό στόλο. Ένα ναυτικό βάσει τη δική μα ε, ε νομοθεσία μένει τρει μήνε στη θάλασσα και δύο σπίτι του. Ένα Ταϊβανό μπορεί να βρίσκεται τρία χρόνια στη θάλασσα χωρί κανένα δικαίωμα ε, και όχι μόνο σε μισθοδοτική σκοπιά αλλά σε εργασιακό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε λίγο πολύ πιο ρεαλιστικά τα πράγματα. Στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, είχαμε τη ε, διαπραγμάτευση της συμφωνίας. Στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης δεν τέθηκε κανένα τεχνικό ζήτημα. Οι αρχές ε, το μόνο που είπαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ε, τι θέλετε. Θέλετε να μου επιβάλλετε μία ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μία εμπορική συμφωνία αλλιάς. Ε, κατανοώ ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστές όταν θέτουμε, θέτουμε τέτοια θέματα. Θα πρέπει ε, να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην Καμπόν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σωματικό πρόβλημα από τις πληροφορίες που έχω εγώ, αλλά ε, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Στι συμφωνίε των χωρών ΑΚΕ υπάρχουν επίσης ε, ρήτρε για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι ανάγκη υπάρχει να εισάγονται αυτά τα στοιχεία στις αλληλευτικές συμφωνίες, οι οποίες το μόνο που θα κάνουν ε, είναι να δημιουργήσουν πολύ περισσότερε δυσκολίε και όχι πλέον εκτίματα. Ε, θα χαθεί μια λευτική συμφωνία ε, την οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξανασυνάψουμε διότι άπαξ και σταματήσει να γίνεται μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτη χώρα κατά πάσα πιθανότητα όταν πάψουν οι διαπραγματεύσεις ε, δεν συνεχίζεται η συμφωνία είναι πολύ περιορισμένε οι δυνατότητε να συνεχιστούμε. Τώρα, το ζήτημα του να καταβάλλονται δικαιώματα για την αλληλεία στην ε, ανοιχτή θάλασσα έχει μία λογική. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στι περιφερειακέ οργανώσει αλληλεία. Αλλά αυτό που δεν θα θέλουμε είναι να μην χρησιμοποιείται όπω ε, πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση ω πειραματόζω. Πηγαίνουμε πάντα στο Α με τα σκάφη μα, για παράδειγμα, για να δούμε κατά πόσον μπορεί να γίνει μεταβίβαση δικαιωμάτων και τελικώ όλα αυτά οδηγούν σε μείωση της ανταγωνιστικότητας του στόλου μας. Επικρίσεις για τις αλλιευτικές συμφωνίες, λέει ο κύριος Πένας, και ότι είναι ενισχύσεις. Εγώ δεν αρνούμαι ότι είναι Υπάρχουν και επικρίσεις για τις ενισχύσεις. Μπορεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρχουν περισσότερα ωφέλη. Ε, δεν είναι ενισχύσεις τα, η ενίσχυση για τη ε, διάλυση ενός σκάφους. Αν υπάρχει για παράδειγμα ε, Αλληλευτικό απόθεμα από ένα σκάφος ε, της Ταϊβάν. Η κατάσταση πώς έχει. Δεν τηρούνται ούτε εργασιακά δικαιώματα. Από μισθούς μηδέν. Ε, και είναι δυνατόν να είναι το ίδιο ε, και να συγκρίνονται τα ίδια με τα δικά μας τα σκάφη αυτοί που δεν πληρώνουν κανένα δασμό και που εμείς πληρώνουμε και δασμούς ε, και τηρούμε συγκεκριμένα ε, όρια. Δεν επιδοτούμε τελικώς στα σκάφη αυτών των τρίτων χωρών. Και τέλο, θα ήθελα να ζητήσω συνοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μα είπαν ότι υπάρχουν κατευθυντήριε γραμμέ από το 2004 που λένε ότι τα ε, που αλλιεύουν σε διεθνή ύδατα ε, προστατεύονται. Υπάρχουν προβλήματα ανταγωνιστικότητα και θα πρέπει να ζητήσω συνοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να πω ότι είναι ασυνεπές αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς στηρούμε τους κανόνες, λέτε ότι πρέπει να πληρώνουμε δικαιώματα στην ανοιχτή θάλασσα. Ζητώ συνοχή. Είναι ένα στόλο ο οποίο έχει πρόβλημα ανταγωνιστικότητα και θα πρέπει να τον υποστηρίξουμε, διότι έχουμε ένα στόλο ο οποίο πληρεί τι καλύτερε και τι περισσότερε προποθέσει παγκοσμίω και δεν μπορεί να λέμε ότι δεν μπορούμε να τον ενισχύσουμε και τον, να τον υποστηρίξουμε. Μου φαίνεται ότι δεν έχουν καμία συνέπεια τόσο ακούγονται. Και τέλο, για το σχόλιο τη κυρία Λεβίν, και το γεγονό ότι πρέπει να δεχτούμε με καλό μάτι τη μεταφορά δικαιωμάτων αλληλεία των ανεπτυγμένων χωρών προς ε, λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε, αναφερόμαστε σε μεταναστευτικά είδη. Δεν αναφερόμαστε σε είδη τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι ιδιοκτησία των χωρών. Πρόκειται για πόρου που επειδή είναι μεταναστευτικά είδη θα μπορούν να βρίσκονται σε συγκεκριμένα ύδατα. Οι χώρες αυτές δεν έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν αυτούς τους πόρους. Δεν την έχουν. Και το μόνο που προσπαθούμε να κάνουμε όταν γίνονται τέτοιες συζητήσεις είναι να έχουμε το ίδιο με αυτό που γίνεται στην Κάνα. Έχουν έρθει και έχουν εγκατασταθεί οι Κορεάτες ε, στην Κάνα και εκμεταλλεύονται τους σπόρους στην Κάνα. Τι γίνεται στην Ανέγου Ινέα, αυτό που θα γίνει είναι ότι θα έρθουν οι Φιλιππινέζοι, οι Ταϊβανέζοι και θα ε, τα μετατρέψουν σε εργοστάσια την Ανέγου Ινέα, θα ψαρεύουν εκεί και μάλιστα θα τους ε, εγκρίνει και η παγκόσμια κοινότητα η κατάσταση της Ευρώπης δεν μπορεί να είναι μια κατάσταση που να λέμε όλο χαρά ότι είμαστε ανεπτυγμένη χώρα. Υπάρχουν άλλες χώρες ε, οι οποίες μπορεί να θεωρούνται λιγότερο ανεπτυγμένες. Και αν δεν υποστηρίξουμε τον ευρωπαϊκό στόλο, ένα τομέας ο οποίος αποτελεί πρότυπο και από τον οποίο εξαρτώνται πάμπολες θέσεις εργασίας έχει ένα ζωφερότατο μέλλον. Αναφερόμαστε σε θέσεις εργασίας, συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Το να λέμε όλο χαρά ότι πρέπει να δεχτούμε τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων μας σε τρίτες χώρες ε, και ότι αυτά είναι ο νόμος της ζωής και τα πράγματα ελέγχουν, με συγχωρείτε, αλλά εγώ αυτή τη συζήτηση αρνούμαι να την κάνω. Bueno. <laughs> Por Dios. Προς Θεού, τρεις άνθρωποι θέλουν να μιλήσουν μετά από όσα είπατε. Πέντε λεπτάκια για να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίασή μας. Θα δώσω το λόγο στους τρεις κυρίους και κανείς άλλος στη συνέχεια, διότι δεν θα έχω χρόνο εγώ να ολοκληρώσω με την ημερήσια διάταξη. Από τα αριστερά προς τα δεξιά. Παρακαλώ. Χαβιέρ Γκαράτ, πρόεδρος της Europest, της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης που προστατεύει τα δικαιώματα των πλειοκτηκτών. Ήθελα να αναφερθώ και στο πρώτο και στο δεύτερο πάνελ, γιατί δεν μιλήσαμε στο πρώτο πάνελ. Για το πρώτο πάνελ θα ήθελα να πω ότι μου άρεσαν πάρα πολύ οι δύο παρεμβάσεις των ομιλητών, μου φάνηκαν πολύ λογικές και ρεαλιστικές. Δεν είχαν καμία σχέση με τις απόψεις άλλων ανθρώπων που δεν είναι καθόλου ρεαλιστικές. Και καταλήγω στο εξή συμπέρασμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, εκτιμήσουμε τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση και το μόνο που μπορούν να κάνουν οι επιστήμονες είναι να μας δώσουν προσεγγιστικά στοιχεία για την ε, μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Και ε, να ολοκληρώσουμε την τελευταία φράση του κυρίου Παστόρ ότι μπορούν να αξιολογήσει ο επιστήμονα, αλλά δεν μπορεί να λαμβάνει απόφαση. Και να λάβουμε υπόψη και αυτό που έλεγε ο κύριο Πένα, ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και άλλοι φορείς προσπαθούν να λαμβάνουν τις αποφάσεις επιστήμονες και αυτό αποδεικνύεται σε πολλές περιφερειακές οργανώσεις ελίας όπου η εντολή που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να υπογράφει αποκλειστικά βάσει τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και μάλιστα στην χειρότερη δυνατή περίπτωση και όχι στην καλύτερη περίπτωση προς όφελος του ελευτικού στόλου. Και επίσης η μέγιστη βιώσιμη απόδοση θα πρέπει ε, να χρησιμοποιηθεί ώστε οι ενδιαφερόμενοι να οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Τη σήμερον ημέρα κανείς δεν αμφισβητεί το στόχο της της βιώσιμης απόδοσης παρά το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθεί από επιστημονική σκοπιά. Αυτό το οποίο αμφισβητούμε όλοι, όπως αποδείχθηκε σήμερα και από αρκετού, είναι η ημερομηνία του 2015. Όχι γιατί δεν μα αρέσει, αλλά γιατί γνωρίζουμε ότι είναι αδύνατο για κάποια είδη να φτάσουν στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση το 2015. Και όπω έλεγε ο κύριο Πένα, ακόμα και αν σταματήσουμε να αλλιεύουμε ε, κάποια συγκεκριμένα είδη. Πρόκειται για μια χρονολογία η οποία δεν μπορεί να θεωρείται κανόνας, θα πρέπει να είναι απλώς μια ημερομηνία προσανατολισμού ώστε να φροντίσουμε τα περισσότερα είδη και οι πληθυσμοί των αποθεμάτων να αρχίσουν να αυξάνονται. Μας απογοητεύει ιδιαίτερα το θέμα αυτό όταν συζητάμε με διαφόρους οι οποίοι έχουν αυτή την ε, ημερομηνία του 2015 ως θέσφατη. Τα ε, βιολογικά όρια ασφαλείας τα οποία εφαρμόζονται ε, ε, εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν είναι, έχουν επιτευχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να επιτύχουμε αυτό το στόχο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης στο μέτρο του δυνατού. Μία ερώτηση που ακόμα δεν έχει απαντήσει κανείς παρά το γεγονός ότι έχει τεθεί πολλές φορές και ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί. Στην αλληλεία πολλαπλών ειδών πώς θεωρείτε ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή τη ε, μέγιστη βιώσιμη απόδοση, γιατί ακόμα δεν κατάλαβα. Για το δεύτερο πάνελ και εμείς ως Ευρωπαίοι συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει υπεραλίευση σε συγκεκριμένους τομείς του στόλου. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό που δεν θέλουμε είναι να γενικευθεί διότι όπως είπαμε στην περίπτωση των θηνοειδών είναι πολύ συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ε, στον ευρωπαϊκό στόλο σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει υπεραλίευση. Αυτό που πρέπει ε, να πούμε είναι ότι πρέπει να δρούμε αναπερίπτωση, αναείδος και αναείδος αλίας. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη νέα τεχνολογία που έχουμε επί του σκάφους. Πολλές φορές θεωρείται ότι η νέα τεχνολογία ως κάτι κακό και με περισσότερες δυνατότητες αλίας. Έχουμε βάσει αυτής της νέας τεχνολογίας πιο σύγχρονα σκάφη περισσότερη ασφάλεια για το πλήρωμα, ε, επισητιστική ασφάλεια και επίσης βελτιώνεται η επιλογή μεταξύ των ειδών αλίας. Αυτή είναι προσωπική πείρα ε, που είχα πρόσφατα σε ένα σκάφος ε, στη Μεσόγειο με αλίας αρδέλας Με τις συσκευές που έχουμε μπορούμε να γνωρίζουμε επακριβώς το μέγεθος της αρδέλας και ο υπεύθυνο αλλιέα, αυτό που κάνει, και αυτό έγινε σε αυτή την περίπτωση, είναι να μην συνεχίσει να αλλιεύει αν δεν είναι σωστό το μέγεθο. Όταν θα βρει το σωστό μέγεθο, τότε ρίχνει το δείχνη του και συλλέγει τα ψάρια με το νόμιμο μέγεθο των 22 εκατοστών που επιτρέπεται. Να μην καταδικάζουμε τι νέε τεχνολογίε, γιατί χάρη σε αυτέ τι νέε τεχνολογίε έχουμε περισσότερη ασφάλεια επί του σκάφου, επισητιστική ασφάλεια και καλύτερη δυνατότητα επιλογή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Σύντομα σα παρακαλώ, γιατί αλλιώ δεν θα μπορέσω να δώσω δώσω το λόγο στους τρεις ομιλητές. Σας παρακαλώ να είστε πιο λακωνικοί. Εκπροσωπώ την Ένωση που υπερασπίζεται τα δικαιώματα του στόλου στη Κανάρια νησιά. Είμαι πρόεδρος της Ένωσης και ασχολούμαι με τις απεντήσεις ε, στις τρίτες χώρες στο Μπιλμπάο. Ε, υπάρχει αλεία των ε, Συνεδών, αλλά όχι μόνο. Ε, νομίζω ότι δεν πρέπει να ισχυριζόμαστε οτιδήποτε. Πολλές περιοχές εξαρτώνται από αυτή την αλεία. Ε, θα πρέπει να απασχολούνται περισσότεροι ντόπιοι να εφαρμόσουν το σύστημα της εθελοντικής εκφόρτωσης κτλ. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να μιλήσω για τα δικαιώματα. Είναι απαραίτητο ένα τέτοιο σύστημα, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστεί όπως ε, στην Κίνα. Γιατί όμως ε, νομίζω ότι πρέπει να εφαρμοστεί ε, το σύστημα στην Κίνα και όχι μόνο σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η αλληλεία ε, γίνεται με όρους απαράδεκτους για τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κανείς δεν λέει τίποτα γι' αυτό. εγώ λέω ότι από όσο αντιλαμβάνομαι πρέπει να υπερασπιστούμε ε, και τα δικαιώματα των κρατών μελών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 17% των μέτρων αποσκοπούν στη μείωση της δυναμικότητας ε, του στόλου μας και νομίζω ότι αυτό θα συνεχίσει μέχρι το 2013. Ταυτόχρονα ακούμε σχόλια από άλλες πλευρές σχετικά με την εκμετάλλευση των πόρων ε, των μη ανεπτυγμένων χωρών, αλλά ταυτόχρονα μας λένε ότι δεν θα δοθούν επιδοτήσεις για την απόσταση των παλαιών σκαφών. Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να αποχωρήσουν οι διερμηνείς σε ένα δευτερόλεπτο, κύριε Πένας. Ευχαριστώ. Ήθελα να σχολιάσω ένα ζήτημα που ακόμη δεν αναφέρθηκε. Πρέπει να μελετήσουμε αυτή τη μελέτη αντικτύπου που ανέφερε η κυρία Λέβιν και τα προβλήματα που εντοπίζονται εκεί για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, στην ε, Γαλλικία θα χαθούν πάνω από 3.000 ε, θέσεις απασχόλησης αν ισχύσουν αυτά τα μέτρα που προτείνονται για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. κατόπιν, τι θα γίνει με την απαγόρευση των απορρίψεων. Εντάξει, είναι σωστό το μέτρο, αλλά δεν νομίζω ότι δίνουμε μια σφαιρική λύση. Τους δεν δέχονται αυτό το μέτρο πολλά Θα πρέπει να διασφαλίσουμε μια σταθερότητα στον κλάδο. Η Κομισιόν για τρία λεπτά αν μπορεί να απαντήσει. Θα κάνω μια απόπειρα κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, το πώς ε, θα λειτουργήσει η μέγιστη βιώσιμη απόδοση στα ε, στην αλληλεία πολλαπλών ειδών. Το λέω όλη την ημέρα. Δεν υπάρχει μαγικός τύπος. Υπάρχει η δυνατότητα να δούμε αλληλεία να δούμε τι συμβατότητα υπάρχει μεταξύ μέγιστη βιώσιμη απόδοση για κάθε είδο και από εκεί και πέρα να δούμε μέχρι ποιου σημείου μπορούμε να έχουμε ένα επίπεδο αλληλεία σε ένα είδο που θα οδηγεί σε υπερεκμετάλλευση ή υποεκμετάλλευση σε σχέση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση των άλλων ειδών που συνδέονται με τη συγκεκριμένη αλληλεία. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί και οι συμβιβασμοί ε, και αυτό που ζητάμε από τους ε, επιστήμονες είναι ε, να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τα διάφορα μοντέλα μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Από εκεί και πέρα μπορούμε είτε να αποφασίσουμε ότι θα προσαρμοστούμε στο επίπεδο μέγιστης βιώσιμης απόδοσης ε, του είδους ε, που υπερεκμεταλλευόμαστε περισσότερο και από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε μέσω τεχνικών μέτρων να προσπαθήσουμε να κάνουμε διαχωρισμό στο μέτρο του δυνατού των διαφόρων ειδών ή να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν ενδιάμεσο τύπο εκτίμησης της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Δεν υπάρχει μαγική συνταγή, πρέπει να τα δούμε όλα ένα περίπτωση και να προχωρούμε σιγά σιγά ε, για να βλέπουμε πώς μπορούμε να έχουμε την εφαρμογή της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης ώστε ε, αυτό που είπε ο Νόλη σήμερα να ισχύει. Δεν αναφερόμαστε σε μαγικούς αριθμούς, θέλουμε απλώς να ξεκινήσουμε να προχωράμε στη σωστή κατεύθυνση και να φροντίσουμε να προχωρήσουμε αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα με τα πολιετή σχέδια. Τα πολιετή σχέδια βασίζονται σε αυτή την έννοια και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα να γίνει ξεχωριστή συζήτηση σε κάθε περίπτωση για την κατάλληλη εκτίμηση της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και πώς μπορούμε να την εφαρμόσουμε στην περίπτωση του κάθε είδους. Τώρα, για το όσα είπε ο κύριος Φοντάν, σημειώνω το θέμα της Κίνας. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι χωρίς να ξεκινήσουμε πολιτικές συζητήσεις, δεν είναι και ε, στο απειρόβλητο η Κίνα. Δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά στα πλαίσια του κανονισμού ε, του εφαρμοστικού για την παράνομη λαθρέα και αναρχιαλία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κάνει ε, έρευνες και αποστολές ε, και πρακτικές σε πολλές χώρες του κόσμου και σας διαβεβαιώ χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες ότι δεν υπάρχει ούτε μία χώρα στον κόσμο που να είναι στο απειρόβλητο. Δεν υπάρχει καμία χώρα που να είναι στο απειρόβλητο, επαναλαμβάνω. Ε, μια μικρή διόρθωση. Εγώ δεν είπα ακριβώς, ε, δεν θυμάμαι τουλάχιστον να είπα ότι το 2000, από το 2002 και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενδιαφέρεται να ε, ενισχύσει διάλυση σκαφών. Απλώς λέω ότι δεν έχουμε ως προσανατολισμό τη μείωση του στόλου και αυτό είναι σημαντικό και η διαφορά είναι σημαντική. Δεν λέμε ότι πρέπει να λέμε οπωσδήποτε στο κράτος μέλος ότι πρέπει να μειώσετε το στόλο σας. Απλώς λέμε ότι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν κάποια ποσοστά υπεραλίευσης και αντιλαμβανόμαστε ότι για να τα λύσουμε υπάρχει και ένα κονδύλιο παροπλισμού σκαφών και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν το ε, κονδύλιο αυτό για τον παραπλησμό των σκαφών τα κράτη-μέλη είναι διαφορετικός. Άλλοι δαπανούν πολλά κονδύλια και κάποιοι άλλοι δαπανούν λιγότερα. Δεν είναι μια πολιτική που κατευθύνει τα κράτη-μέλη, απλώς διατίθεται στα κράτη-μέλη κονδύλια για τον παραπλησμό των σκαφών, ώστε ο καθένας να τα χρησιμοποιεί βάσει του εθνικού του σχεδίου για την ε, δημιουργία θέσεων ε, και την απώλεια θέσεων εργασίας. Ναι, υπάρχει απώλεια θέσεων εργασίας, αλλά και στη διατήρηση της κατάστασης όσο έχει πάλι θα χαθούν θέσεις εργασίας. Πριν από τη μεταρρύθμιση και πάλι υπάρχουν ε, απώλεια θέσεις εργασίας. Εγώ επισκέφτηκα και χώρες που θεωρούνται ως ε, πρότυπα αλλιευτικής διαχείρισης, χώρες στις οποίες ζηλεύει ο κόσμος όλος και εκεί υπάρχει ε, μεγάλο πρόβλημα με την απώλεια θέσεων εργασίας, ιδίως όσον αφορά το θέσει εργασίας επί των σκαφών. Άλλο είναι από εκεί και πέρα οι βιομηχανίες που σχετίζονται με την αλληλεία, με μεγάλη προστιθέμενη αξία και δυνατότητα να δημιουργήσουν θέσει εργασίας στις παράκτης κοινότητες. Αλλά το θέμα των θέσεων εργασίας δεν θα πρέπει να το βλέπουμε μόνο ε, ως θέση εργασίας ε, πληρώματος. Ε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Μπορούμε να είναι περισσότερε ή λιγότερε, αλλά δεν μπορούμε να το αποφεύγουμε το θέμα των θέσεων εργασία και θα πρέπει να τα βλέπουμε μόνο ε, με συνολική προοπτική. Όχι μόνο τι χάνεται ω πλήρωμα, αλλά και τι μπορούμε από εκεί και πέρα να αντισταθμίσουμε με συμπληρωματικέ δραστηριότητε σε παράκτιε κοινότητε που έχουν ε, πολύ σημαντικέ δυνατότητε δημιουργία θέσεων εργασία. Δύο τελευταίε παρατηρήσει, Κάρμενα, μου επιτρέπει. Ένα λεπτό και μόνο η μέγιστη βιώσιμη απόδοση δεν είναι περιβαλλοντικός στόχος, είναι στόχος ο οποίος θέλει να εξεύρει ισορροπία μεταξύ της βιολογικής, της κοινωνικής και της οικονομικής βιωσιμότητας. Επομένως δεν είναι όνο περιβαλλοντικός στόχος. Και τέλος, ο κύριος Σουάρε έχει απόλυτο δίκιο, η διαδικασία διαβούλευσης για την προετοιμασία της ε, πρότασής μας έλαβε τη μεγαλύτερη υποστήριξη από πλευράς κρατών μελών και από τους ενδιαφορομένους ε, για το ζήτημα της διατήρησης και η διαβούλευση είναι και για να εισακούονται και οι προτάσεις σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν άκουσε την άποψη της πλειοψηφίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν με τα τελευταία σημεία της ημερήσιας διάταξης, ε, ανακοινώσεις ε, για τις αποφάσεις των συντονιστών. Εάν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, επειδή ε, καθυστερήσαμε και είχαμε και τις προφορικές ερωτήσεις, θεωρούμε ότι εγκρίνονται. επόμενη συνεδρίαση 12 Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ όλους, ιδιαίτερα τους εισηγητές και όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση σήμερα το απόγευμα, τους ομιλητές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Πρόεδρος ευχαριστεί και τους διερμηνείς. Πέρα συνεδρία.